αλλά και για απλούς Ευρωπαίους πολίτες. Να σας υπενθυμίσω ότι στις 4 Ιουλίου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ένα ψήφισμα για τις ηλεκτρονικές μαζικές παρακολουθήσεις ε, Ευρωπαίων πολιτών και ζήτησε από την Επιτροπή μας, την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών και παραθέτω εδώ να κάνει μία εισβάθος έρευνα για το θέμα αυτό σε συνεργασία με το ε, εθνικά κοινοβούλια και εμπειρογνώμονες Ευρωπαϊκής Ένωσης των Πολιτειών και να αναφέρει τα όσα ε, θα διαπιστώσει πριν από το τέλος του έτους. Συνεργαζόμαστε με τις αρμόδιες επιτροπές, οι οποίες ε, μπορεί να ενδιαφέρονται για το θέμα αυτά, παραδείγματος χάρη η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και Διεθνούς Εμπορίων και καθώς επίσης και τον αρμόδιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις διμερείς σχέσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και επίσης ε, η συνεδρία είναι αυτή ανοιχτή και σε συναδέλφους ε, από ε, άλλες επιτροπές ή εκπροσώπους εθνικών κοινοβουλίων που ασχολούνται και αυτοί από την πλευρά τους με το θέμα αυτό. Πρόκειται για μια συζήτηση η οποία είναι ανοιχτή για τους Ευρωπαίους πολίτες. Το βασικό θέμα το οποίο συζητούμε αφορά τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών σε περίπτωση παρακολούθησης και ο συνάδελφος Κλοντ Μωράες είναι ο αρμόδιος εισηγητής. Σήμερα το πρωί εγκρίθηκε η πρόταση του συζητητή και έχουμε τέσσερις μήνες για να κάνουμε την έρευνα διότι φτάνουμε ε, προς το τέλος της ε, θητείας μας γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό ώστε να μπορέσουμε να ψηφίσουμε την έκθεση ε, στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών μέχρι το Δεκέμβριο και να περάσει στη συνέχεια από την Ολομέλεια του Ιανουαρίου και να ψηφιστεί και εκεί. Να σας πω ότι υπάρχει συνεργείο ε, από τη Γερμανία που ε, μαγνητοσκοπεί την ε, συνεδρίαση και αυτό στα πλαίσια του ντοκιμαντέρ του David Barnett ο, για τα θέματα αυτά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το ντοκιμαντέρ θα ολοκληρωθεί και αυτό μέχρι το τέλος της θητείας. Παρακολουθούν τις εργασίες μας από τον Ιανουάριο του 2012 και τούδε και παρακολουθούν πολύ στενά τον τρόπο με τον οποίο ο νέος κανονισμός για την προστασία των δεδομένων ε, θα ψηφιστεί εδώ από το Κοινοβούλιο και πώς γίνεται η συζήτηση εδώ στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Έχουν μαγνητοσκοπηθεί πολλές από τις συνεδριάσεις μας ήδη και ε, συνεχίζουν φυσικά και θα συνεχίσουν και στο μέλλον. Να περάσουμε τώρα στη συνεδρίασή μας. Θα μιλήσουμε λοιπόν με ε, δημοσιογράφους που κάνουν σχετική έρευνα και θα ασχολούνται με τα θέματα αυτά ε, και θα κάνουμε και εμείς τη σχετική μας έρευνα. Γι' αυτό ακριβώς και ξεκίνησε, ξεκινά αυτή η συνεδρίαση και θα ακούσουμε κάποιους εξ αυτών. Ε, στα θέματα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων. Μας ενδιαφέρουν τα θέματα των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ε, το δικαίωμα στην αποζημίωση και στην ε, αποκατάσταση και επίσης ε, όλα όσα προβλέπει η Ευρωπαϊκή Χάρτα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων που αποτελούν ένα απόσπαστο τμήμα της συνθήκης της Λισαβόνας. Γι' αυτό ακριβώς και καλωσορίζουμε εδώ τους προσκεκλημένους μας σήμερα το απόγευμα. Καταρχάς, τον κύριο Ζακ Φολερού, Καλωσορίσατε, ορίσατε, δημοσιογράφος από την εγνωσμένου κύρους εφημερίδα Le Monde, η οποία δημοσίευσε εφημερίδες για ένα γαλλικό σύστημα για τη συγκέντρωση ε, όλων των μορφών των ηλεκτρονικών δεδομένων. Στη συνέχεια, ο κύριος Jacob Applebaum, δημοσιογράφος ερευνητής, υπεύθυνος λογισμικού και ερευνητής ασφάλειας ε, ε, πληροφορικής ε, με το πρόγραμμα TOR και τρίτον μέσω βίντεο διάσκεψης διότι δεν μπορεί να παραστεί εδώ στη συνεδρίαση ο κύριος Άλαν Ρουσπρίτζερ, ο οποίος είναι ο αρχισυντάκτης ε, της Guardian και θα συμμετέχει εδώ σε μια βίντεο διάσκεψης στις 4.30. Θα γίνει επίσης και μία βίντεο διάσκεψη με τον Glenn Greenwald, το οποίος είναι πολύ γνωστός ε, γιατί έχει ένα ιστολόγιο ε, με τον τίτλο «Ασφάλεια και Ελευθερία» στην Guardian. Είχε δεχτεί να συμμετάσχει από τη Βραζιλία. Δυστυχώς ε, τελικώς αυτή η βιντεοδιάσκεψη δεν μπόρεσε να γίνει. Επομένως, θα ακούσουμε μόνο τον κύριο Ρους Πρίτζερ σήμερα το απόγευμα. Θα σας ενημερώσω λίγο καλύτερα για το πρόγραμμα στη συνέχεια και τώρα να ακούσουμε τους δύο προσκεκλισμένους μας που είναι εδώ παρόντες, τον κύριο Φολορού καταρχάς και κατόπιν τον κύριο Άπελμπαμ. Κύριε Φολορού, έχετε το λόγο. Διαδικαστικό, πραγματικά όμω διαδικαστικό. Yes, sorry, I think... Ναι, ζητώ συγγνώμη κυρία Μορβάη. Γιατί ματαιώθηκε η βίντεο διάσκεψη, ε, θα μας ενδιαφέρε να μάθουμε το λόγο. Είναι θέματα προγραμματισμού, είναι στη Βραζιλία αυτή τη στιγμή και δεν μπορούσαμε καιρός να το προγραμματίσουμε. Πάντως θα φροντίσουμε σε επόμενη συνεδρίαση να πραγματοποιηθεί είναι πολύ σημαντικός ο χρόνος και αγωνιζόμαστε να τελειώσουμε πριν το τέλος του έτους. Ε, αργότερα, εν ευθέτω χρόνο, θα ε, συναντηθούμε, θα κάνουμε τη διάσκεψη. Έχουμε για σήμερα τρεις δημοσιογράφους και θα είναι αρκετά ενδιαφέρον. Αρχίζουμε λοιπόν, ο κύριος Πολυγού πρώτος. Ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Ε, να πω δύο λόγια μόνο από την Ναταλή Νουγκερέντ που είναι η διευθύντρια της εφημερίδας Le Monde και ε, σε ό,τι αφορά σήμερα είναι ευθύνη των δημοσιογράφων να εξηγήσουν τη δουλειά τους στη Γαλλία ακόμα θεωρείται ίσονο σημασία αυτή η παραβίαση των ε, ατομικών και δημοσίων ελευθεριών. Εγώ παρίσταμαι απλούστατα ως δημοσιογράφος για να σας εξηγήσω τι κάναμε, πώς εργαστήκαμε και τη σειρά των άρθρων ε, που μας επέτρεψαν να αποκαλύψουμε αρχές Ιουλίου την ύπαρξη ενός συστήματος υποκλοπών ε, μαζικό και μαζικής ε, αποθήκευσης πληροφοριών ατομικού προσωπικού χαρακτήρα στη Γαλλία που διέφευγε κάθε έλεγχο, είτε είναι αυτός διοικητικός είτε είναι πολιτικός. Ε, μετά από τις αποκαλύψεις που έγιναν για το σύστημα PRISM, κάναμε αυτή την έρευνα. Στη Γαλλία, σε αντίθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες του Ηνωμένου Βασίλειο, όλα τα τεχνικά μέσα της χώρας για υποκλοπές ηλεκτρονικών σημάτων δεν είναι σε ξεχωριστή υπηρεσία όπως είναι τα διάφορα συμβούλια ασφαλείας, υπηρεσίες ασφαλείας των Αγγλοσαξώνων. Αυτό είναι μονοπόλιο μιας υπηρεσίας πληροφοριών DGSE στα γαλλικά που είναι η υπηρεσία πληροφοριών και κάνει κατασκοπία εκτός των γαλλικών συνόρων. Ε, η DGSE λοιπόν από το 2005, 2006 και 2007 σε αυτή την τριετία απέκτησε τεχνικά μέσα ε, πάρα πολύ σημαντικά που χρηματοδοτήθηκαν, εγκρίθηκε η χρηματοδότηση από τη Βουλή ε, για να αναπαθμιστεί τεχνολογικά, έτσι το παρουσιάζουν οι αρχές της χώρας, για να έχουμε τα μέσα που θα μας επιτρέπουν ε, τις ηλεκτρονικές υποκλοπές, να εξασφαλιστούμε σε περίπτωση ηλεκτρονικού πολέμου και να εξασφαλίσουμε και την κυριαρχία μας για τη συλλογή πληροφοριών και να είναι πραγματικά γαλλικής κοπής ε, όλο αυτό το σύστημα. Ε, θα έρθω στη συνέχεια στους λόγους που ενδεχομένω ε, εξοπλίστηκε έτσι ηλεκτρονικά η Γαλλία και τι προβλήματα προέκυψαν. Για μας το θέμα δεν ήταν αν είναι καλό ή κακό οι βασικές δυτικές χώρες να καταπολεμούν την τρομοκρατία. Αυτό που μας ενδιαφέρει ήταν ο έλεγχος, πώς ελέγχονται όλα αυτά. Αυτή βάση δεδομένων όμως που αποθηκεύει, σε αντίθεση με τα όσα δημοσίως λέγονται, αποθηκεύει επί χρόνια και διατηρεί δισεκατομμύρια στοιχείων και δεν είναι αποκλειστική χρήση αυτής της υπηρεσίας πληροφοριών, η οποία είναι εξωτερική, εκτός των γαλλικών συνόρων. Αλλά στη Γαλλία υπάρχει και ένα σύστημα που θεωρεί ότι αυτή η σημαντική βάση δεδομένων σε ένα από τους ε, μεγαλύτερους υπολογιστές, τον πιο ισχυρό, ε, είναι κάτι που χρησιμοποιούν και άλλες γαλλικές υπηρεσίες πληροφοριών που υπόκεινται στο γαλλικό νόμο και εργάζονται εντό των γαλλικών συνόρων, στην επικράτεια της χώρας. Και καθημερινά ε, ανατρέχουν σε αυτά τα στοιχεία ερήμην των ελεγκτικών μηχανισμών. Γι' αυτό εμείς κάναμε αυτές τις αποκαλύψεις αρχές Ιουλίου. Τι σημαίνει αυτό. Σήμερα η γαλλική ε, αντικατασκοπία ή ακόμα και το τελωνίο ή ε, ε, το οικονομικό έγκλημα, η καταπολέμησή του, το ΣΔΟ ας πούμε, μπορεί να μπει σε ένα κομπιούτερ και να ζητήσει πληροφορίες για τον οποιοδήποτε πολίτη. Μπορεί να είναι κάποιοι που θεωρητικά έχουν σχέση με την τρομοκρατία ή με αξιόπινες πράξεις, αλλά υπάρχουν κάποιοι κανόνες για να υπάρξει αυτή η πρόσβαση αυτός που ζητεί την πληροφορία θα πρέπει να εντάσσεται σε κάποιους νόμους της χώρας. Στην προκείμενη περίπτωση όμως δεν υπάρχει κανένας που να δίνει ε, την έγκριση για τη συλλογή των στοιχείων, για την επεξεργασία τους ε, και στη συνέχεια τη διατήρηση και αποθήκευσή τους. Υπάρχει ένα παράλληλο σύστημα ανεξέλεγκτο το οποίο εγγράφεται πραγματικά σε αυτά που αποκάλυψε ο Έντουαρτ Σνόουντεν για την ύπαρξή του πρίσμου. Δηλαδή, μια χώρα μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας που έχει σημαντικά ε, μέσα για μαζική υποκλοπή στοιχείων, για μαζική αποθήκευση, θεωρεί ότι ε, είναι απλώς ένα θέμα της εκτελεστικής εξουσίας και ανεξέλεκτα μπορεί να κάνει αυτές τις ενέργειες και στη συνέχεια να διαχειρίζεται αυτό το υλικό. Στη Γαλλία, βεβαίως, Υπάρχει νόμος σχετικά που αφορούσε στην αρχή τις τηλεφωνικές υποκλοπές, τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. Υπάρχει ακόμα αυτός ο νόμος. Υπάρχουν αρμόδια όργανα ε, που θα πρέπει να απευθύνονται σε αυτά οι υπηρεσίε πληροφοριών, η αστυνομία όταν θέλουν να παρακολουθούν ε, τα τηλέφωνα Γάλλων πολιτών. σε λέγεται αυτός ο οργανισμός και υπάρχει. Αλλά ε, για τα στοιχεία, τα μεταστοιχεία εντό εισαγωγικών, μετά την επεξεργασία που αποθηκεύονται, η Sense.es δεν έχει ούτε τα μέσα, δηλαδή ούτε το προσωπικό διαθέτει, ούτε το τεχνικό, αλλά ούτε το δικαίωμα να προβαίνει σε τέτοιες ενέργειες για να κοιτάει τι γίνεται σε αυτή την τράπεζα δεδομένων. Δηλαδή, ε, όλα αυτά τα αποκαλύψαμε αρχές Ιουλίου και... Πώς να το πω... Προκάλεσαν περιέργως μικρή αντίδραση αυτές οι αποκαλύψεις. Γι' αυτό έρχομαι ενώπιον σας σήμερα. Δηλαδή, επί της ουσίας, μια χώρα σαν τη Γαλλία, με τέτοια παράδοση, με πολύ συγκεντρωτική χώρα, η Πέμπτη Γαλλική Δημοκρατία, θεωρεί ότι ε, δεν τρέχει και τίποτα. Δεν είναι τόσο ασυνήθιστο να έχει ένα κράτος τέτοια τεχνικά μέσα και να κάνει τέτοια χρήση. Ε, καταρχήν θετική αξιολογείται αυτή. Για μας αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια φτώχεια στη Γαλλία ως προς ε, τους ελέγχους της εξουσίας τα αντίβαρα. Τώρα περιορίζεται μόνο στο τεχνικό πλαίσιο αυτή η συζήτηση. Ε, τι δυνατότητες έχουμε δορυφόρους, κοριούς, ε, υποβρύχια, καλώδια μπορούμε να υποκλέπτουμε. Περισσότερο τεχνική είναι λοιπόν η συζήτηση παρά ως προς τα δικαιώματα. Και ποιος είναι ο περίμετρος, η περίμετρος, συγγνώμη, και ο περίγειος και ποια είναι η ελευθερία των πολιτών και τα δικαιώματά τους και πώς προστατεύεται η ιδιωτική ζωή του καθενός. Ή ακόμα και ολοκλήρων κρατών είναι επιχειρήσεων. Και σήμερα για μας ο μόνος πολιτικός πρωταγωνιστής που αντέδρασε είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και η Επιτροπή σας. Και θα μπορούσε κανείς να αναρωτηθεί γιατί. Το Κοινοβούλιο αντιδρά με σοβαρότητα, ίσως τελικά διότι δεν περνάει τόσο πολύ από το χέρι του ε, να αλλάξει αυτή την κατάσταση και νομοθετικά. Γιατί τελικά, και μιλώ για την Γαλλία, γιατί τη χώρα αυτή ξέρω καλύτερα. Η Γαλλία γιατί αντέδρασε τόσο λίγο ή ε, ακόμα και στις αποκαλύψεις για το πρίσμα, ε, για την ε, Αμερικανική Υπηρεσία Εθνικής Ασφαλείας που υποκλέπτει ή παρακολουθεί κυβερνήσεις, επικοινωνίες μεταξύ Γάλλων Υπουργών. Γιατί δεν εδρασε τόσο ε, χλιαρά η Γαλλία. Οι χώρες δεν έχουν βεβαίως την οικονομική δυνατότητα ισχύ, ούτε καν την ισχύ που έχουν οι Ηνωμένε Πολιτείε. Αλλά μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών υπάρχει μια αρχή αποτροπή, ας πούμε. Δεν μπορεί η Γαλλία να μπει σε μια λογική τέτοια κλιμάκωση τη κατάσταση με τι Ηνωμένε Πολιτείε. Υπάρχει μεγάλο κίνδυνο τελικά να δούμε την Ουάσιγκτον αντιδρά λέγοντα, αποκαλύπτοντα μάλλον αυτά που κάνει η Γαλλία. Που παρακολουθεί κάποιου γείτονέ τη, ίσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ποιο ξέρει. Όλα αυτά τα στοιχεία λοιπόν μας ενδιέφεραν. Ε, είναι σε εξέλιξη ακόμα αυτή η προσπάθεια. Ας πούμε το γαλλικό σύστημα συλλογής και διατήρησης και αποθήκευσης δεδομένων δεν είναι ακόμα γνωστό. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι συμφωνίες υπάρχουν ανάμεσα στις γαλλικές υπηρεσίες ε, ε, πληροφοριών και τις βασικές τηλεφωνικές εταιρείες Orange, SFR, Bouygues, Free Όλες αυτές οι εταιρείε τηλεφωνίας έχουν κάνει συμφωνίες με το κράτος και τις μυστικές υπηρεσίες, αλλά δεν ξέρουμε τι είδους είναι αυτές. Όπως και στις Ηνωμένε Πολιτείε οι ομολόγοι τους έχουν ε, καταρχήν συμφωνία με τηλεφωνικές εταιρείε για να μπορούν να υποκλέπτουν και να παρακολουθούν τις τηλεφωνικές και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Παραμένουν πολλές ε, γκρίζες ζώνες. Η μόνη απάντηση που είχαμε εμείς στην αποκάλυψή μας προήλθε από μια κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία ε, που ασχολείται με τις πληροφορίες και έχει ως αποστολή να αποπειράται, και το τονίζω αυτό, προσπαθεί απλώς να ελέγχει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι γαλλικές μυστικές υπηρεσίες. Είναι πολύ πρόσφατη αντιπροσωπεία της Βουλής από το 2007 με πάρα πολύ περιορισμένες εξουσίες. Παράδειγμα, μπορούν να συναντούν μόνο τους διευθυντές των γαλλικών ε, μυστικών υπηρεσιών. Δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε έγγραφα και στοιχεία παρά μόνο πάρα πολύ περιορισμένοι και επίσης τα μέλη ε, ε, είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας της Βουλής ή ο πρόεδρος άλλων επιτροπών σημαντικών που δεν μπορούν να αφιερώσουν τόσο πολύ χρόνο σε αυτή τη δραστηριότητα. Σταματώ εδώ γιατί φαντάζομαι οι ερωτήσεις και απαντήσεις θα είναι πιο ενδιαφέρουσες. Εμένα ως δημοσιογράφο τι μου κάνει εντύπωση. Επευθύνθηκα σε διάφορους αρμοδίους φορείς στη Γαλλία και εκπροσώπους εξουσίας και βλέπω ότι οι Γάλλοι βουλευτές δέχονται έτσι, ανερυθρίαστα ότι οι κρατικές υπηρεσίες μπορεί να έχουν το ελεύθερο. Απολύτως. Ε, αυτό το έχουν κάνει κτήμα τους. Δηλαδή την, ε, παραβίαση του ελεγκτικού ρόλου την έχουν απολύτως ε, υιοθετήσει. Αντιδρούμε εμεί οι δημοσιογράφοι και όχι οι βουλευτές. Ε, μας λένε, ε καλά πώς κάνετε έτσι, δεν τρέχει και τίποτα. Ε, και όταν μιλούμε με τις υπηρεσίες και με εκπροσώπους που πρόσκυνται στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, που εργάζονται ακόμα και στο Πρωθυπουργικό Γραφείο ή και σε ε, υπευθύνους ηθήνοντες των υπηρεσιών πληροφοριών που δέχονται τη συζήτηση, πέρα από την απάντηση επί της ουσίας, κάθε φορά μας λέγουν και σε μένα επανειλημμένως μου το έχουν πει, «Μα γιατί αγωνιάτε και ανησυχείτε» Δεν υπάρχει λόγος, διότι αυτοί που διαχειρίζονται αυτά τα στοιχεία, τις μαζικές υποκλοπές, είναι δημοκράτες Γάλλοι, ε, διέπονται από αισθήματα ευγενή. Ναι, εντάξει, αυτό μπορεί να ισχύει, αλλά υπάρχουν και άλλοι που έχουν πρόσβαση σε αυτές τις ε, πληροφορίες και δεν ξέρουμε τι χρήση γίνεται. Αλλά λέει ναι, μην ανησυχείτε, είναι μια τεχνολογική δυνατότητα, είναι σε καλά χέρια και δεν χρειάζεται ιδιαίτερο έλεγχο, δεν θα ε, συμβεί τίποτα. Και πάλι είναι θέμα αρχή όμω. Γι' αυτό είναι σημαντική η νομοθεσία, διότι αν δώσουμε αυτή την απαλλαγή και, και την ε, ε, εικόνα που μας δίνουν να την πιστέψουμε ότι είναι για την καταπολέμηση τρομοκρατίας και της διάθεσης των όπλων. Όλα αυτά καλά. Αλλά όταν δεν υπάρχει έλεγχος μπορεί ο καθένας να το διαστρεβλώσει και να το χρησιμοποιήσει για ιδιωτελείς σκοπούς και προσωπικούς και αστυνομικούς και πολιτικούς. Το έχουμε ξαναδεί αυτό. Στην Προεδρία του Νικολά Σαρκοζή είδαμε ότι υπήρξαν κάποια σκάνδαλα τα οποία σήμερα έχουν επιβεβαιωθεί ότι η δικαιοσύνη είχε διαστρεβλωθεί για να προστατεύει πολιτικά συμφέροντα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο έλεγχος, ένα αντίβαρο στην εξουσία αυτή. Βγαίνουμε από το κράτο δικαίου. Και εμείς ως δημοσιογράφοι και η Ναταλή Κερέτ που ξέρετε, ίσως δεν ξέρετε, ανέλαβε τη διεύθυνση της εφημερίδας μου αρχές του 2013, θέλει να διατρανώσει ότι δημοσιογράφος ίσον πολίτης. Ε, η άσκηση της δημοσιογραφίας δεν είναι μεχόμενη η δημοσιογραφία αυτή, απλώς υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα των πολιτών. Δεν είμαστε μεσιανιστές, ε, ούτε θεωρούμε ότι έχουμε καμιά αποστολή, τη δουλειά μας κάνουμε. Ε, επαγρυπνούμε και ελπίζουμε και οι δικές σας εργασίες στο Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες να οδηγήσουν και σε κάποια μεγαλύτερη συνειδητοποίηση. Εγώ είμαι συγκρατημένα αισιόδοξο, πάρα πολύ συγκρατημένα, για να μην πω απεσιόδοξο, για το τι μπορεί να συμβεί στη Γαλλία. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Φολορού, επίση ευχαριστούμε που ήσασταν σύντομο και ακριβή. Και τώρα ο κύριο Άπελμπαουμ έχει το λόγο. Ορίστε. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Είναι τιμή μου να παρίσταμε εδώ, όπου έρχομαι για πρώτη φορά. Θα ήθελα έτσι να δούμε όλο το τοπίο. Γιατί ξέρετε έχω εμπειρία, επί δεκαετία ε, έχω δουλέψει στο δίκτυο ανωνυμίας που χρησιμοποιεί ο κόσμο τόσο ώστε να αποφύγει κάποιο είδους ε, έλεγχο, παρακολούθηση, λογοκρισία, διάφορες, ε, διάφορες τέτοιες και κάποιο software που έχει να κάνει με αυτά. Επίσης έχω κάνει ρεπορτάζ ελεύθερα, αλλά επίσης έχω υποστεί ο ίδιος παρακολούθηση από προγράμματα συναφή με αυτό που συζητούμε. Οπότε και οπωσδήποτε θα πρέπει να σας πω για το θέμα μας. Αλλά θα ήθελα να δούμε, όπως είπα, την ευρύτερη εικόνα, το ευρύτερο τοπίο. Πέρα από τον Σνόντεν, πέρα από τις καταδόσεις, είναι το ότι η NSA έχει ένα γενικό, γενικότατο κατασκοπικό πρόγραμμα, το οποίο ακόμη δεν έχει περιγραφεί στον κόσμο. Δηλαδή ότι το FBI και η CIA επίσης έχουν παρόμοια προγράμματα. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν ο κόσμος λέει για αυτά τα προγράμματα που είναι σαν φυλακή, τι θα πει αυτό. Θα πει ότι πρόκειται για ένα πρόγραμμα σύμφωνα με το οποίο ε, κάποιοι σε νομικά πρόσωπα, σε εταιρείε, σε μη κερδοσκοπικούς φορείς. Αυτοί είναι συνένοχοι με το ΣΥΠΗΝ. Και αυτό. Οπότε το, έτσι, έτσι κάνουμε στη ΣΥΠΑ. Ας πούμε, η Google, η Yahoo, το Skype, η Microsoft έχουν τέτοια συστήματα μέσα στο δίκτυό τους. Και εκουσίως και εν γνώση τους λαμβάνει χώρα μια τέτοια διαδικασία παρακολούθησης. Και υπάρχουν επίσης και κάποια πάρα πολύ σημαντικά νομοθετήματα τα οποία ονομάζονται ε, κάτι σαν επιχειρηματικά, επιχειρησιακά αρχεία ε, και υπάρχουν και εις βάρος μου τέτοιοι φάκελοι. Και εγώ είμαι φαγγελό, θα σα πω άλλη φορά αυτή την ιστορία. Οπότε, αυτά φυσικά και θεωρούνται αντισυνταγματικά. Ε, υπάρχει τέτοια γνωμοδότηση. Πάντω, η κάθε υπηρεσία έχει κάτι τέτοιο από πλευρά τη NSA, τη Εθνική Υπηρεσία Ασφάλεια. Άρα, δεν είναι θέμα μεταδεδομένων. Είναι φάκελοι. Οτιδήποτε δηλαδή δημιουργεί μία, ένα νομικό πρόσωπο ή κάποιο φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο υπάρχει εκεί. Οπότε μέσα από τους υπολογιστές, μέσα από τη λειτουργία της εταιρείας, τα πάντα εκτός αν υπάρχει ρητή μνήμα προς το αντίθετο, έχουμε αυτό που το λέμε φυλακή. Πάντως δεν πρόκειται μόνο για ένα, ένα λογισμικό, ένα πρόγραμμα αυτό που λέγεται prison φυλακή. Υπάρχει και κάτι άλλο, άλλο όνομα για κάποιες εταιρείε που ίσως δεν ταιριάζουν ακριβώς αυτό. Λέγεται αυτό upstream. Αυτό είναι, κάτι, είναι περιγραφικό. Δηλαδή, το θέμα είναι τι γίνεται λόγω τεχνολογικής. Ε, υποτίθεται ότι αυτό δεν γίνεται σε συνεργασία με τον παρακολουθούμενο. Παρακολουθείτε η αδίποτε επικοινωνία συγκεκριμένου νομικού προσώπου. Και αυτό ονομάζεται upstream ε, και υπάρχει το σύστημα Tempura το οποίο είναι ένα άλλο σύστημα το οποίο το τρέχουν με βασίλειο. Και αυτό προσωμιάζει με το upstream γιατί ακριβώς καλύπτει ό,τι μπαίνει και ό,τι βγαίνει στο διαδίκτυο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο κάθε λοιπόν δεδομένων περνάει μέσα από το τέμπορα και κρατάτε εκεί δεν είναι μόνο ε, τα μεταδεδομένα, όλα τα δεδομένα, τέτοιο σύστημα επομένως. Σαν το πρίσμ σαν το πρίσμ, όχι πρίσμ, πρίσμ, ε, κάνει αυτή την παρακολούθηση, είναι κάτι το οποίο είναι απίστευτο, δεν έχει γίνει ποτέ πριν. Θυμάστε πώς είχε φοβηθεί ο κόσμος όταν εμφανίστηκε το Έσελαν. Όταν αποκαλύφθηκε λοιπόν αυτό στον κόσμο, τότε δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι θα μπορούσε αυτό να, να, να, να, να λάβει τέτοιες μορφές, πολύ χειρότερες όπως είναι τις σημερινές, γιατί το Έσελον είναι παιχνιδάκι, είναι, είναι, είναι παιχνιδάκι για παιδιά που φτιάξαν οι χάγκε. Γιατί αυτά τώρα που αποκάλυψε ο Σνόντεν, σε σχέση με αυτά τα σημερινά προχωρημένα συστήματα που είναι τόσο προχωρημένα που δουλεύουν με έναν τρόπο που έχει ως εξή. Πρώτα πρώτα ε, έχουμε τα νομικά, το, νομικό πλαίσιο, μετά έχουμε την παρακολούθηση, κατασκοπία και τρίτον η τρίτη φάση, το πως το πρόγραμμα Gini που πρόσφατα αποκαλύφθηκε από την Washington Post που το Gini είναι ένα μόνο από αυτά γιατί τακτική εκμετάλλευση, ένα από τα αυτά προγράμματα και θέλουν να δουν επομένως τι κάνεις. Οπότε και δεν μπορούν να, να το upstream, δεν μπορούν να πάρουν τις πληροφορίες από το Google, οπότε τι κάνουν, χακάρουν, μπαίνουν μέσα στον υπολογιστή σου. Και ε, στο Washington Post πρόσφατα είπε ότι έχουμε δεκάδες χιλιάδων συστημάτων που ακριβώς ε, έχουν παγιδευτεί με τέτοιο τρόπο από το πρόγραμμα Genie, αλλά υπάρχουν και άλλα. Και άλλα. Μου είναι οικεία, δεν έχουν αποκαλυφθεί στον κόσμο, αλλά θα υπάρξει αποκάλυψη όταν αυτά στοχεύσουν συγκεκριμένους ανθρώπους, συγκεκριμένο λογισμικό και αυτό γίνεται για κάποιους που δεν είναι τρομοκράτες. Κάποια θέματα λοιπόν υπάρχουν σε αυτά τα έγγραφα σημαίνουν ότι τελικά μόνο κατά εξαίρεση παρακολουθούνται οι τρομοκράτες. Αν έχουμε 30 παρακολουθούμε, ένας από αυτούς θα είναι τρομοκράτης ε, φοβερό είναι, πολύ ανησυχητικό είναι αυτό. Γιατί έτσι σημαίνει ότι οποιοδήποτε παρακολουθείται, μπορεί να παρακολουθείται. Και από αυτού, από, από μια μεγάλη ομάδα προσώπων, να είναι φερόμενοι ως τρομοκράτε, δηλαδή να μην έχουν καν παραπεμφθεί, ερευνηθεί, καταδικαστεί ω τρομοκράτες, ένας-δύο μόνο. Αυτοί επομένω. ε, υφίστανται αυτή την τύχη παρά το ότι δεν ε, έχουν καταδικαστεί, χαρακτηριστεί. Κανείς αυτούς δεν είναι τρομοκράτης. Μόνο κάτι εξαίρεση. Άρα θα πρέπει να δούμε πώς όλα αυτά συναρμόζουν. Γιατί είπαμε, είναι μάτι ο κανείς να προσπαθεί να καταλάβει την τεχνολογία. Να, να δούμε τι είναι αυτά τα οποία μπορεί να καταλάβει ο κόσμος. Έχουμε το πρόγραμμα τα πέντε μάτια. Και έχουμε υπηρεσίε ε, από Νέα Ζηλανδία, Καναδά, ε, υπήρχε συμπληροφωνία δηλαδή από, από Νέα Ισλανδία, Αυστραλία, Καναδά, Ηνωμένο Βασίλειο και Αμερική, παρά την, αμερι την, την επάσταση που έγινε κατά τον, ε, του, του, του επικισμού Βρετανού, έγινε ε, ε τέτοιου είδου συμφωνία, τέτοιου παρακολούθηση από του Βρετανού. Τι είναι αυτό, συνταγματικό, είναι αυτό δημοκρατικό, αυτό στηρίζει τη, χώρα μου. δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ακριβώ όταν η NSA η δική μας παρακολουθεί του Βρετανού, ...έχει αυτή τα ίδια θα πούνε. Αυτή είναι λοιπόν θέση οι υπηρεσίες, η NSA, η GCSQ, είναι η εταίρη πρώτου επίπεδου. Η BND είναι η γερμανική υπηρεσία που θεωρείται υπηρεσία τρίτου επίπεδου. Υπάρχει μια ποσόστοση στην καθεμία θα πρέπει μένω και ο τέρος τρίτου επίπεδου, θα πρέπει κάτι να εισφέρει στην εταιρική αυτή σχέση. Δεν είναι τόσο σαφές πώς λειτουργεί αυτή η εταιρική σχέση, αλλά υπάρχει αυτή η ενδιαφέρουσα διάκριση μεταξύ διαφορετικών επίπεδων. Αυτό τελικά συναρμόζεται και χρησιμοποιείται κατά διάφορους φοβερούς τρόπους. Ας πούμε υπάρχουν κάποιες βάσεις δεδομένων για υπογραφές όπου υπάρχει αυτή η υπογραφή, το αποτύπωμα τέλος πάντων τη φωνή μας, ε, υπάρχουν τα, το αριθμό τηλεφώνου μας, το email μας εκεί πέρα και κάθε φορά που κάποιος παίρνει ένα καινούριο gadget και βάζει εκεί το όνομά του, ένα από αυτά τα, τα στοιχεία που έχει η βάση δεδομένων, τότε συνδέεται και αυτό με τη βάση δεδομένων. Και επομένως υπάρχει ένα σύστημα παρακολούθησης οποιοδήποτε, οποιοδήποτε επί της γης και υπάρχουν και κάποια συστήματα γεωγραφικού εντοπισμού, η ΕΝΕΣ έχει ένα σύστημα όπου εντοπίζουν τον κόσμο και έχουν, έχουν αυτό το, το αστιάκι και λένε τους ε, ανοιχνεύουμε και τους ξεπαστρεύουμε. Οπότε όλα αυτά τα δεδομένα της παρακολούθησης ε, τι είναι τελικά, είναι κάτι σαν ε, ρομπότ, υπτάμενα, το οποίο σκοτώνει τον κόσμο χωρί να τον έχει περάσει από δίκη, επομένως τελικά υπάρχει βέβαια επίπτωση πάρα πολύ απτή όπως το να χτυπήσει κανείς κάποιον με πύραυλο. Όλα αυτά είναι κατά κάποιο τρόπο παθητικά. Η τακτική βέβαια εκμετάλλευση δεν είναι καθόλου παθητική, αλλά δεν είναι παθητική η NSA. Αυτό είναι ένας μύθος. Υπάρχουν, υπάρχουν δηλαδή κάποιοι, ε, κάποιοι μαθηματικοί εγκέφαλοι εκεί πέρα με τα παλτά τους ε, κουκουλωμένοι που κάθονται και μουτζουρώνουν χαρτιά. Δεν είναι καθόλου έτσι η NSA. Είναι απίστευτο, είναι απίστευτη που δουλεύουν εκεί είναι καλοί, πολύ καλοί. Γι' αυτό και μερικοί από αυτούς επειδή είναι καλοί, όπως ο Σνόντεν και άλλοι στο παρελθόν, ε, την κοπάνισαν και, και προέβησαν σε καταγγελίες. Ε, κάνουμε πάρα πάρα πολύ ενεργές και ενεργητικές ε, επιχειρήσεις. Δεν είναι διαταγές τους πράκτορες της NSA να πάνε σε κάποια πόλη, να εισδύσουν, να μπουν σε, σε κάποια δίκτυα κάποιων. Αυτό είναι τρομερό. Είναι εκπαιδευμένοι αυτοί. Όπως είναι εκπαιδευμένος, όπως ξέρει τη δουλειά του ο διαρρήκτης, ξέρουν και αυτοί πώς θα μπουν στο δίκτυο του σπιτιού. Είναι τρομακτικά αυτά. Εξορισμό, είναι, εγκρυπτό και απαραβίστο, αντιδημοκρατικά και αυτοί που που κάνουν τις παρακολουθήσεις είναι με ένα εμπιστή για την επιχείρηση, για την ε, υπηρεσία, αλλά είναι αμόρφωτη. Ξέρετε, ούτε mail δεν μπορεί να στείλουν. Βάζουν άλλους συναδέλφους να τους γράψουν τα, τα, τα mail τους. Μπορούν να ξέρουν να κάνουν ε, μια τεχνική δουλειά, αλλά δεν ξέρουν κάτι απλό. Και η ίδια η αρχιτεκτονική αυτών των συστημάτων είναι έτσι επίτηδες. Ξέρουμε ας πούμε για το φαξ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρακολουθήθηκε είχε παγίδευση δηλαδή κάποιον φαξ από το τέμπους. Κάποια προκωδικοποιημένα δεδομένα που περάσουν από το φαξ τα είχαν ε, παγιδεύσει από πριν, μπορέσαν να τα μαζέψουν, άρα δηλαδή μπορούν, έχουν και την επιλογή του επιθετικού όπλου. Και αυτό έχει να κάνει με την κλίμακα από οικονομικής πλευράς που συντρέχει και έτσι θα πρέπει να μην ξεχνούμε ότι η υπηρεσία πληροφοριών των ΗΠΑ δεν δίνει δεκάρα για το κοινοτικό δίκαιο. Δεν δεσμεύεται από αυτό. Λέτε εσείς για ισορροπία, για αναλογικότητα, για μέτρα κατά της τρομοκρατίας. Μα τι, τότε θα πει η Εθνική Πίεση Πληροφοριών ότι εγώ θα παρακολουθήσω όλο τον κόσμο. Έτσι έγινε και με την υπόθεση Αθήνα στην, ε, στην Ελλάδα. Γιατί δεν ξέρουμε αν ήταν οπωσδήποτε η, αν ήταν αλλά ξέρουμε ότι και βουλευτές και από τον Πρωθυπουργό παρακολουθήσανε. Ε, κάποιοι πάρα πολύ ικανοί, πολύ ισχυροί. Και δείτε, ενώ παλιά είχαμε την ε, στρατιωτική αντιπαράθεση, τώρα έχουμε κάποιου πίσω από ένα κομπιούτερ οι οποίοι μπορούν να, έχουν, να, να χτυπήσουν τελευταία γραμμή άμυνα, που είναι ο Πρωθυπουργό τη χώρα. Βρέθηκε, βρέθηκε το τηλέφωνό του στο σπίτι του του Πρωθυπουργού. Ναι. Και αυτό που το έκανε αυτό. Ο Πρωθυπουργό τι να κάνει, δεν, δεν ήξερε, τι, να, τι, τι μπορούσε να κάνει. Βλέπετε λοιπόν πόσο όλα αυτά αλλάζουν την ισορροπία δυνάμεων πάρα πολύ. Επομένω, πέραν αυτού, Έχουμε διάφορα κέντρα στον πλανήτη, εδώ και εκεί. Συγγνώμη, αισθητήρε, αισθητήρε. Και αυτοί οι αισθητήρε, μπορείτε να σκεφτείτε πώ είναι, έτσι το κάνω και εγώ. Ε, να έχουμε μια γεωγραφική σφαίρα και να έχουμε του αισθητήρε και μπορεί η Εθνική Πληροφορία όλα αυτά να τα παρακολουθήσει γιατί έχει δορυφόρου και υπάρχουν και άλλοι δορυφόροι πίσω από του δορυφόρου τηλεπικοινωνία. Ε, τι νομίζετε κάνουν αυτοί οι δεύτεροι δορυφόροι. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που αξίζει να ερευνηθούν. Ρίξτε όμω μια ματιά τι γίνεται με το διαδίκτυο και τα τηλέφωνα. Όταν η Αμερικάνικη ΚΙΠ δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε ένα σύστημα με κάποιο είδου συνεργασία ή κάποιο είδου πρόγραμμα ε, ε, συμμετοχής πληροφοριών, τότε μπαίνει, α πούμε είδαμε ότι έχουν κάλυψη σε κάποια μέλη που γνωρίζουμε ότι οποιοδήποτε κράτο δεν θα έδινε εκουσίως αυτά τα δεδομένα. Ε, πού τα βρήκανε αυτά, έχουν βάλει κάτι μέσα στο σύστημα και τα πήραν αυτά τα δεδομένα. Και κάνανε σε πραγματικό χρόνο τέτοια έρευνα, βγάλανε από όλη αυτή την σφαίρα πληροφόρησης, την ηλεκτρονική, ό,τι θέλανε και τα βάλανε ε, σε αυτή τη βάση δεδομένων. Μιλάμε τώρα για πάνω από 100 χρόνια κατά τα οποία παίρνουν δεδομένα. Ε, λοιπόν, είναι πλανητικό το σύστημα παρακολούθησης δεν έχει να κάνει με τον νόμο, δεν έχει να κάνει με τη δικαιοσύνη. Τι ελπίδα έχουμε. Η μόνη μας ελπίδα είναι να έχουμε κάποιο είδους κωδικοποίηση για να αλλάξουμε το πώς μπορούμε να απαξιώσουμε αυτά τα οποία δεν μπορούμε να σταματήσουμε να μας τα παρακολουθούν, να μας τα κατασκοπεύουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Αμπλουμπαμ, πριν ξεκινήσει η συζήτηση, θα ήθελα να σας πω τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Στις 4.30 σε 3 τέταρτα περίπου έχουμε προγραμματίσει τη βίντεο διάσκεψη με τον τρίτο προσκεκλημένο μας, τον κύριο Ρος Μπέτσερ, τον ε, ε, αρχισυντάκτη Ρους τον αρχισυντάκτη της Guardian News και Νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε τη συζήτηση στο μεταξύ, να ακούσουμε τον εισηγητή, τους και όδες εισηγητές και να αφήσουμε το λόγο από εκεί και πέρα στα μέλη που θέλουν ε, να παρέμβουν. Να σας υπενθυμίσω όμως ότι εδώ γίνεται μια κρόαση. Θέλουμε λοιπόν να συζητήσουμε και να θέσουμε συγκεκριμένες ερωτήσεις ε, στους ε, προσκεκλημένους μας. Και να μην χρονοτριβούμε με πολιτικές δηλώσεις, να επικεντρωθούμε στις παρουσιάσεις που ακούσαμε από τους δημοσιογράφους, ε, τους οποίους καλέσαμε εδώ για να ε, μιλήσουν σε αυτή την ακρόαση και θα ήθελα να το έχετε κατά νου αυτού πριν λάβετε το λόγο. Ο κύριος Κλόντ Μωρέας καταρχάς, ο εισηγητής. Thank Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τους δημοσιογράφους για την παρουσία τους εδώ, διότι ουσιαστικά είναι αγγελιαφόροι των ε, καταγγελιών ε, που γίνονται και τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα για τα όσα έχουν κάνει ε, και αυτούς και τον κύριο Ρας διότι είναι η κοινωνή των μηνυμάτων που μας στέλνουν αυτοί οι οποίοι κάνουν τις καταγγελίες. Ο κύριος Φολορούς, τα άρθρα του στη ε, έγραψε κάποια πράγματα τα οποία και έλευθερα, διότι αυτή τη στιγμή εμείς εδώ σήμερα δεν ακούμε μόνο τι έγινε με το PRISM, που είναι το αμερικανικό πρόγραμμα, αλλά εξετάζουμε και τι έγινε με Ευρωπαίους πολίτες ε, και τα δεδομένα ε, τα οποία διέρευσαν. Και εσείς στα άρθρα σας εξηγήσατε πως η Γαλλική Υπηρεσία Πληροφοριών είχε πρόσβαση σε δεδομένα και στοιχεία πολιτών της. Και φυσικά εσείς τα άρθρα σας εξηγήσατε πώς η αστυνομία και άλλες υπηρεσίες είχαν πρόσβαση σε στοιχεία τα οποία ε, στην πραγματικότητα θα έπρεπε να έχουν πρόσβαση μόνο οι υπηρεσίες πληροφοριών. Και για να συνεχίσω, ε, επειδή ο πρόεδρος μας είπε να είμαστε ακριβείς, ε, θεωρώ ότι εσείς ως δημοσιογράφοι μπορείτε να έχετε άποψη για το τι συνέβη στη Γαλλία διότι δεν έπρεπε αυτά τα στοιχεία να ε, δοθούν οπουδήποτε αλλού και αν αυτό συμβαίνει στη Γαλλία γνωρίζουμε ότι φυσικά θα μπορούσε να συμβαίνει και σε άλλα κράτη-μέλη. Και στόχος της έρευνάς μας δεν είναι απλώς ε, να ε, επικεντρωθούμε στο τι συμβαίνει μεταξύ ημών και Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και τι συμβαίνει σε κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά πόσον υπάρχει νομική βάση για να υπάρχει ε, μεταφορά στοιχείων ε, στη Γαλλία ή σε οποιαδήποτε άλλη ε, χώρα μέλος και θα πρέπει να διαπιστώσουμε αν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει σε κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν συμβαίνει εδώ και αρκετό καιρό στη Γαλλία και αν συνέβαινε τώρα, συνέβαινε πριν στο παρελθόν, αν συνέβη πολύ πριν γίνει η καταγγελία από τον Έντορτ Σνόντεν και εάν ξαφνικά βρέθηκαν οι δημοσιογράφοι οι οποίοι μας εξηγούν τι συμβαίνει. Αυτή είναι η ερώτηση μου λοιπόν για σας ε, στη Λεμόντ και για τον κύριο Applebaum να πω ότι ήταν ε, τόσο ε, πολλά όλα αυτά τα οποία μας είπατε, πραγματικά εμπλουτίσατε τη συζήτηση που θα μπορούσαμε να σας καλέσουμε σε αρκετές και διαφορετικές ακροάσεις. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξή, λοιπόν μέσα σε όλα αυτά που μας είπατε. Ε, για να τα δούμε λίγο όλα στη σωστή τους αναλεγία. Αναφερθήκατε στο τεμπόρα όλα τα θέματα που αφορούν τα κράτη-μέλη. Μία ερώτηση αν όντω όλα αυτά συμβαίνουν, θα θε, ήθελα την ανάλυση σας για το τι γίνεται με αυτές τις πληροφορίες. Γιατί γίνεται αυτή η μαζική μεταφορά στοιχείων. Γιατί επενδύονται δισεκατομμύρια σε αυτές τις ε, ε, μεταφορές στοιχείων. Ε, μας ενδιαφέρει μόνο η τρομοκρατία. Πώς το αναλύετε εσείς το θέμα. Ευχαριστούμε τον Κλοντ Μοράς και γιατί ήταν τόσο ακριβής και τήρησε το χρονοδιάγραμμα και ήταν εύστοχα αυτά που μας είπε. Στη συνέχεια και σκιώδεις ο κύριος Άξελ Φως, καταρχάς. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ είμαι. Ακουστικά μάλλον θα χρειαστείτε. Dank für... Ευχαριστώ πολύ για τα όσα μας είπατε και τις μαρτυρίες που μας ε, μεταφέρετε. Καλό θα ήταν ε, να μάθουμε την άποψή σας και θα με ενδιαφέρει προσωπικά το ψάχνετε. Έω ε, προ το εξή, μιλήσατε για υποκλοπέ στοιχείων και παρακολουθήσει και βέβαια το επικρίνουμε και δεν το θέλουμε σε τέτοιο βαθμό. Αλλά πώ θα χρησιμοποιούν αυτά τα στοιχεία που συλλέγονται έτσι μαζικά. Έχετε να μα πείτε τίποτα περισσότερο. Μα πραγματικά χρησιμοποιούνται για να εκβιάζονται άλλες χώρες. Αυτό εννοείται, δεν το είπατε ρητά. Χρησιμοποιούνται για εμπορικό σκοπό, εμπορική κατασκοπία, οικονομική κατασκοπία. Και από πλευρά σας, στις νέες τεχνολογίες και στις νέες δυνατότητες και τα επιτεύγματα που έχουμε σήμερα. υπάρχει μεγαλύτερη ή μικρότερη δυνατότητα παραβίασης των δεδομένων και μεγαλύτερη ή μικρότερη ασφάλεια. Γιατί πάντα βρισκόμαστε σε μια λεπτή ισορροπία ανάμεσα στην ιδιωτική ζωή αφενός και στην προστασία του δημοσίου συμφέροντος αφετέρου και του κοινωνικού συνόλου. Εσείς έχετε κάποιες ιδέες γι' αυτό. Ένα αυτό, ένα δεύτερο. τα γνωρίζετε, αυτά γνωρίζετε κάποια ε, ασυνείδητη ή λιγότερο υπεύθυνη χρήση αυτών των στοιχείων έχετε αποδείξει από τις μυστικές υπηρεσίες. Ε, χρησιμοποιούνται δηλαδή για δόλιους σκοπούς. Η κυρία Νετβέλτ που είναι σκιώδη συγκήτρια. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τους δύο μιλητές μας. Ε, άκουσα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτά που μας είπατε. Νομίζω ότι το βασικό ερώτημα αυτής της έρευνας δεν θα είναι τόσο τι γνωρίζουν οι κυβερνήσεις γι' αυτό, γιατί θα είναι πολύ πιο εύκολο να καθορίσουμε τι δεν γνωρίζουν, γιατί είναι πολύ λιγότερα αυτά που δεν γνωρίζουν, αλλά γιατί φαίνεται να έχουν αποτύχει οι έλεγχοι και το σύστημα ε, λογοδοσίας. Ε, γιατί δεν έχουν καταφέρει τα θεσμικά όργανα να έχουν ένα σύστημα το οποίο να μας επιτρέπει ε, να μην ξεφεύγουν τα πράγματα από τα όρια όπως συνέβη σε αυτή την περίπτωση. Εσείς είστε εδώ ως εκπρόσωποι των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Θα ήθελα να ξέρω τι συνέπειες υπάρχουν και στον τύπο, διότι αυτό δεν αφορά απλώς και μόνο τον κάθε πολίτη, αλλά αφορά και την ελευθερία του τύπου, όπως ε, είδαμε με τους δημοσιογράφους της Guardian και θα ήθελα να γνωρίζω πώς ε, ε, αντιδρούν οι συνάδελφοί σας σε αυτό. Ε, τι λένε οι ενώσεις δημοσιογράφων, οι συνδικαλιστικές σας οργανώσεις. Γνωρίζετε για παράδειγμα κατά πόσον εσείς παρακολουθείστε ή σας έχει παρανοχλήσει, πιέσει κάποιος, οι αρχές, Μήπως ε, οι συνάδελφοί σας θεωρούν ότι εάν ο δημοσιογράφος της ε, Guardian αποτελεί αντικείμενο παρενόχλησης θα μπορούσε να συμβεί και κάτι αντίστοιχο και σε αυτούς κάποια μέρα. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό για την ελευθεροτυπία ανησυχούν οι δημοσιογράφοι, μήπως ε, εύλογα ανησυχούν οι δημοσιογράφοι και ε, εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μήπως θα έπρεπε και ε, από την άλλη άκρη του Ατλαντικού να ενωθείτε και να προσπαθήσετε να επαγρυπνείτε για τη δημοκρατία, να ασκήσετε αυτό σας το δικαίωμα σωστά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Άλμπραχτ. Ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ και για αυτές τις πολύ ενδιαφέρουσες απαντήσεις και παρατηρήσεις. Κάποιες ερωτήσεις. Ο κύριος Φουλωρού καταρχάς αναφέρθηκε την ανάγκη να υπάρχει έλεγχος. Έλεγχος σημαίνει να γνωρίζουμε εάν υπάρχει κάτι το οποίο πηγαίνει στραβά ή αν λειτουργούν όλα τα πράγματα σωστά. Και φυσικά αυτό είναι το θεμελιώδης μας δικαίωμα. Και το ερώτημά μου είναι το εξή. Υπάρχουν και νομικές ανησυχίες. Έχετε εσείς νομικές ανησυχίες ή και οι συνάδελφοί σας. Ε, τι γνωρίζετε <laughs> εσείς για αυτά τα προγράμματα ε, εγώ αν ε, ε, ακούσω για αυτά τα προγράμματα από κάποιο νομικό, θεωρώ ότι όλα αυτά δεν συνάδουν με τα αποτελέσματα των αποφάσεων του δικαστηρίου στο Στρασβούργο. Η Γαλλία έχει υπογράψει και αυτή τη χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων και είναι θεμελιώδες ερώτημα το τι κάνει και θα ήθελα να ξέρω πώς το αντιμετωπίζει αυτό η Γαλλία και ε, πώς αντιμετωπίζετε και εσείς αυτά τα ερωτήματα. Και επίση εμείς, επειδή ακριβώ βρισκόμαστε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και επειδή υπάρχουν οι Ευρωπαϊκές Συνθήκες και η Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ε, μας ενδιαφέρει να μας πείτε κατά πόσον θα πρέπει να ισχύει η δεσμευτική χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων και για αυτά τα προγράμματα και για αυτές τις παρακολουθήσεις. είναι κάτι το οποίο θα λάβετε υπόψη σας, θα υπάρχει κάπου στο έργο σας. Και τον κύριο Άπολμπαμ θα ήθελα να το ρωτήσω. Αν υπάρχει συνεργασία μεταξύ αυτών των προγραμμάτων και με άλλες υπηρεσίες πληροφοριών των κρατών μελών, αν έχετε κάποιες πληροφορίες επ' αυτού, ιδίως ε, ε, όσον αφορά αυτό το πρόγραμμα για το ε, X-Score που υπάρχει δυνατότητα σε πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο σε στοιχεία και φυσικά αφορά πολλές υπηρεσίες πληροφοριών και τι γίνεται με αυτούς που σε τελικό στάδιο συλλέγουν τις πληροφορίες που δεν είναι ε, απαραίτητος οι υπηρεσίες πληροφοριών, όπως είπατε και εσείς ε, μπορεί να είναι και οι υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών. γνωρίζουμε κάτι για το νομικό πλαίσιο στο οποίο δραστηριοποιούνται. Εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα, υπάρχουν κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων που ισχύουν και για την Google ή τη Yahoo που δραστηριοποιούνται εδώ στην Ευρωπαϊκή Αγορά. Υπάρχουν σχετικές συζητήσεις ε, για την νομοθεσία ε, και λέγεται ότι δεν επιτρέπεται βάση και τις κείμενες Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων να αποκαλύπτονται αυτά τα στοιχεία και να διαβιβάζονται αυτά τα στοιχεία χωρίς να υπάρχει μια συνθήκη αμοιβαίας αναγνώρισης. Θα ήθελα λοιπόν να μας δώσετε κάποιες περαιτέρω πληροφορίες εσείς. Ευχαριστώ. Κυρία Ένστε, επίση και ο και μετά οι λοιποί συνάδελφοι. Παρακαλώ το χρόνο να σκέφτεστε. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους δύο μιλητές μας και εμπειρογνώμονες. Δύο υποερωτήσεις έχω. Ακούγοντας όλα αυτά που μας περιγράφετε, βλέπουμε να καταραίει ένας μύθος ότι ε, η πληροφορία και η πληροφόρηση έχει να κάνει και με την αυτοδιάθεση του καθενός. Δηλαδή, ο καθένας δεν μπορεί να διαχειρίζεται τις πληροφορίες που τον αφορούν. Ε, καταργείται απολύτως αυτό το ατομικό δικαίωμα. Θα ήθελα να ρωτήσω το δημοσιογράφο της ε, Le Monde, τον κύριο Φολονό, ποια είναι η ελευθεροτυπία τώρα ε, και η προστασία των πηγών είναι δεδομένη, υπάρχει ακόμα αυτό το γεγονός, μπορείτε να εξασφαλίσετε τις πηγές σας. Δηλαδή, δεν πρόκειται μόνο για τους δημοσιογράφους τους ίδιους, κάποιοι σας δίνουν τις πληροφορίες και χρειάζεται απολύτω προστασία των πηγών αυτών. Είναι εξασφαλισμένη ακόμα, είναι δεδομένη, είναι πολύ σημαντικό το πρόβλημα αυτό. Και κάτι που με ενδιαφέρει εδώ ιδιαίτερα είναι το εξή. Έχει αλλάξει η δουλειά σας, η δημοσιογραφία δηλαδή, είναι διαφορετική η προσέγγιση ε, πλέον ε, για να πληροφορήσετε τις καταστάσεις και πώς εξασφαλίζονται όχι μόνο οι δημοσιογράφοι αλλά όλοι οι ενεχόμενοι που σας ενημερώνουν και σας τροφοδοτούν με πληροφορίες. Αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Και ένα ακόμα. Ο έλεγχος. Ακούμε όλα αυτά που μας λέτε και πώς έχει προκύψει αυτό το παγκόσμιο φακέλωμα, το ηλεκτρονικό, που έχει ξεφύγει από κάθε όριο και δεν μπορεί κανείς να το φανταστεί, τότε πραγματικά τι είναι το θέμα του ελέγχου. Εμείς πάντα ζητούμε εδώ κοινοβουλευτικό έλεγχο και στα κράτη-μέλη της Ένωσης αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πάντα να υπάρχει έλεγχος για να ε, μην έχουμε αυτές τις παρακολουθήσεις. Υπάρχουν κύριε Applebaum ε, δυνατότητες πραγματικές από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Μέχρι πού μπορεί να ελέγχει μια βουλή αυτές τις καταστάσεις. Και επίσης από νομική σκοπιά τι πρέπει να γίνει για να ε, βάλουμε ένα τέρμα σε αυτή την κατάσταση. Σε αυτές τις υποκλοπές, σε αυτές τις παρακολουθήσεις, σε αυτό το τεράστιο ζήτημα. Νομικά μπορούμε να κάνουμε τίποτα απέναντι σε αυτό. Αυτά. Ευχαριστώ. Υπόλοιποι τώρα. Έχουμε πολλούς βουλευτές που ζήτησαν το λόγο. Παρακαλώ δύο λεπτά έκαστος για να μπορέσουν να ε, ε, απαντήσουν οι προσκεκλημένοι μας. Ο κύριος Κόγιο, παρακαλώ. Euh, Τα γαλλικά, θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχάς τον κύριο Φολογού και την εφημερίδα Le Monde για όλο αυτό το έργο. Θέλω να κάνω συγκεκριμένες ερωτήσεις εγώ. Οι αποδέκτες ποιοι είναι αυτού του δικτύου που εσείς ε, αποκαλύψατε στο ρεπορτάζ. Είναι Γάλλοι πολίτες, Ευρωπαίοι πολίτες, πολίτες τρίτων χωρών. Όχι αποδέκτες, εννοώ τα θύματα ουσιαστικά, ποιους παρακολουθούν. Και μιλήσατε για συνεργασία μεταξύ διαφόρων γαλλικών υπηρεσιών και αστυνομίας. Αλλά υπάρχουν και άλλοι φορείς που έχουν πρόσβαση και μπορούν να φτάσουν στην υπηρεσία DGSE και να ζητήσουν ενημέρωση. Έχετε ενημέρωση εσείς για συνεργασία με μυστικές υπηρεσίες άλλων κρατών. Γνωρίζουμε ότι έχει θρηματιστεί ο εθνικός και κοινοβουλευτικός έλεγχος στις μυστικές υπηρεσίες. Όταν εξάγονται από κάθε χώρα ε, πληροφορίες από τις μυστικές υπηρεσίες προς άλλες χώρες, έχουμε ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Εξάγονται ε, σε όλο τον κόσμο αυτά τα στοιχεία και κανείς δεν τα ελέγχει. Και ε, θέλω να ρωτήσω τον κύριο Applebaum το εξή. Σας ευχαριστώ πολύ, πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε για τις νέες τεχνολογίες και τα νέα προγράμματα. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που τονίζετε ακριβώς ότι σήμερα παρακολουθούν τους πάντες. Ο Αλεξάνδερ Χέιγ νομίζω το είχε πει αυτό από τους ε, ε ψηλότερους Αμερικανούς αξιωματούχους που είπε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν παγκόσμιο συμφέρον και θα πρέπει να παρακολουθούν όλο τον κόσμο. Την υφήλη ολόκληρη. Πολύ ωραία παρουσιάσατε την κατάσταση και πώς μοιράζονται τα στοιχεία τελείως ασίδωτα ή μυστικές υπηρεσίες μεταξύ τους. Μιλήσατε όμως και για την ε, κρυπτογράφηση και εμείς το 2000-2001 εγκρίναμε τις ε, ε, συστάσεις για να διευρυνθεί η κρυπτογράφηση και να προστατεύονται οι πολίτες. Πώς μπορούμε εμείς να προστατεύουμε τους πολίτες ε, απέναντι σε αυτές τις παρακολουθήσεις και το ηλεκτρονικό φακέλωμα. Ε, δύο λεπτά παρακαλώ, η κυρία Ζίπελ. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω γερμανικά. Okay. Um, Αυτό το σκάνδαλο της NSA ουσιαστικά πρόκειται για τη μαζική παρακολούθηση, το μαζικό φακέλωμα, αλλά κυρίως για ποιο λόγο μαζεύονται όλα τα στοιχεία, για ποιο λόγο συλλέγονται και διατηρούνται και τι γίνεται με τα δεδομένα και τα στοιχεία που δεν έχω εγώ καμιά δυνατότητα ή δεν αποκαλύπτεται τίποτα αξιόπινο. Τι θα τα κάνουμε αυτά τα στοιχεία αυτών των πολίτων. Ε, ο κύριος Φολερό αναφέρθηκε σε ένα ζήτημα και μια κατάσταση που δεν ε, απαντά μόνο στη Γαλλία αλλά και αλλού. Ανεξάρτητα από το σκάνδαλο αυτό, ε, ε, συγχέονται διάφορες υπηρεσίες. Έχουμε τις υπηρεσίες μυστικών υπηρεσιών, κατασκοπία, αντικατασκοπία, αστυνομία, που καλώς ε, δουλεύουν ξεχωριστά και δεν είναι τυχαίο αυτό στις χώρες μας, αλλά από ό,τι φαίνεται τώρα έχουν γίνει όλα ένα συνοθήλευμα. Έχετε βρει στις ε, έρευνές σας ε, κάποιους ε, αρμοδίους που να έχουν προβληματιστεί όχι μόνο από την νομική σκοπιά αλλά και από την κοινωνική σκοπιά. Τι επιπτώσεις έχει αν όλες οι υπηρεσίες αυτές αναμειγνύονται και συγχέονται μεταξύ τους. Ο κύριος Άπελμπαουμ είπε ότι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρακολουθείται και όχι μόνο τα φάξ του και διερωτώμε. και σε αυτό το θέμα και σε άλλα θέματα. Εμείς πώς μπορούμε να ενημερώσουμε ε, το κοινό. Έχουμε συνεδριάσεις που είναι κυκλισμένων των θυρών και εδώ σε αίθουσες και στα γραφεία μας και ε, αναζητούμε ε, την αλήθεια, κάποιες πληροφορίες και ταυτόχρονα παρακολουθούμε. Θα ξέρω ότι δεν μπορείτε να το απαντήσετε αυτό. Ε, αναφερθήκατε και στα διάφορα προγράμματα που συλλέγονται πληροφορίες, παρακολουθούνται επικοινωνίες, ε, εκτός αυτών όμως υπάρχουν και άλλοι τρόποι συλλογή στοιχείων. Δείτε τις λίστες των επιβατών, το PNR και άλλα. Στα πλαίσια των δικών σας ερευνών έχετε βρει αποδείξεις ε, για άλλες πηγές συλλογή στοιχείων που να συνδυάζονται, να ε, συνενώνονται και να συγκρίνονται με άλλα στοιχεία και δεδομένα των πολιτών. Ο κύριος Ιακολίνο, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ήταν πάρα πολύ σημαντική η συνεισφορά των πυρογνωμόνων. Γι' αυτό άλλωστε έχει και σημασία η ερευνητική δημοσιογραφία. Ω υπεύθυνο για την έκθεση για το οργανωμένο έγκλημα γνωρίζω πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει δικαστική και αστυνομική συνεργασία για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε και τη ε, τρομοκρατία αλλά και το οργανωμένο έγκλημα. Αλλά δυστυχώ το επίπεδο εμπιστοσύνη στο οποίο αναφέρθηκε ο κύριο Άπολμπαουμ και η σχέση μεταξύ υπηρεσιών ε, πληροφοριών ε, κάπου χάθηκε. Ε, υπάρχει λιγότερη εμπιστοσύνη και συνδέθηκε περισσότερο με την κατασκοπία η οποία ήταν προς όλες τις κατευθύνσεις. Και ακούστηκαν και από τις προλαλήσαντες αρκετά προγράμματα, το πρόγραμμα πρίσμα έχει τα χαρακτηριστικά του, υπάρχουν κάποια άλλα προγράμματα τα οποία αναφέρθηκαν, το γαλλικό σύστημα της Γαλλικής Υπηρεσίας Περιοφοριών και υπάρχει και το Τέμπορα. Να περάσω στις ερωτήσεις. Την επόμενη εβδομάδα στην ε, Ρώμη θα γίνει το G6 των Υπουργών Εσωτερικών και κατά πάσα πιθανότητα θα είναι και μια ευκαιρία διότι θα υπάρχει και συμμετοχή από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να κατανοήσουμε εάν η ισορροπία μεταξύ ασφάλειας και θεμελιωδών δικαιωμάτων θα μπορούσε ίσως να διασφαλιστεί για το μέλλον. Η πρώτη ερώτηση λοιπόν αφορά την ύπαρξη αυτών των προγραμμάτων παρακολούθηση των κρατών μελών, τα οποία προέκυψαν και συζητήθηκαν πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα, είναι ίσως και μια ευκαιρία να ανακτήσουν την κυριαρχία τους στα κράτη-μέλη εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η άλλη ερώτηση ε, προς τον κύριο Applebaum. Πίσω από το Snowden ποιος κρύβεται, είναι ο Snowden ή υπάρχει κάτι ακόμα. Και κάτι ακόμα και ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε. Υπάρχει δυνατότητα να αξιολογήσουμε πόσο στοιχίζει αυτή η επιχείρηση πρίσμα; Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ σας ευχαριστώ. Ο κύριος, ε, η κυρία Ρομέρο, συγγνώμη, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η ερώτησή μου σχετίζεται με κάποιες από τις προηγούμενες ε, παρεμβάσεις. Επειδή υπάρχει αυτή η ροή πληροφοριών μεταξύ μυστικών υπηρεσιών, σε κάποιες περιπτώσεις ε, κάποια κράτη-μέλη μπορεί να έχουν και το καλύτερο μερίδιο. Πρόκειται για αγορά δεδομένων στην πραγματικότητα. Και η κρυπτογράφηση, όπως προκύπτει σαφώς, ε, φαίνεται ότι είναι κάτι το οποίο χρησιμοποιούν οι περισσότεροι πολίτες ατομικά, αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να είναι και ένα θεσμικό εργαλείο, διότι θα υπάρξει και άλλη αγορά κρυπτογράφηση στη συνέχεια. Αυτό λοιπόν που με ανησυχεί εμένα είναι ότι επειδή ακριβώς αυτή η είδηση προέκυψε από μία εφημερίδα, ο Guardian ήταν αυτή η οποία έκρουσε τον να του κινδύνου για το τι συνέβαινε, ε, δεν είδαμε να επεκτείνεται αυτό στη συνέχεια. Δηλαδή, αν όντω ε, αυτό είναι εξαίρεση, θα πρέπει να διασκεδάσουμε αυτή την αμφιβολία και να μην λέμε, να μην υπάρχει αυτή η ψευδής υπόθεση ότι όλα αυτά γίνονται για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Πρέπει να καταγγείλουμε ότι αυτό δεν βοηθά σε καμία περίπτωση την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, γίνεται για άλλους σκοπούς που προκύπτουν ακριβώς δεν υπάρχει έλεγχος. Και η μάχη κατά της τρομοκρατίας, προκειμένου να είναι αποτελεσματική, θα πρέπει ε, να ελέγχεται κατάλληλα από τα κοινοβούλια. Κυρία Σαρτζεντίνη για δύο λεπτά. Έχω δύο ερωτήσει κύριε Πρόεδρε. Ορίστε παρακαλώ. Πρώτα απ' την Applebaum. Εάν κατάλαβα καλά, αυτό το πρόγραμμα, τα πέντε μάτια στο οποίο αναφερθήκατε, είπατε εδώ εμπλέκονται διάφορε χώρες και η μία βοηθά την άλλη όσον αφορά την παρακολούθηση προσώπων από άλλες χώρες. Τι γίνεται, η νομοθεσία αυτών των χωρών το επιτρέπει, δεν το επιτρέπει, δεν ενδιαφέρει. Μπορείτε να μα ε, πείτε δύο λόγια παραπάνω στον με αυτή τη συνεργασία των ε, υπηρεσιών πληροφοριών. Αλλά για πετε μα τι γίνεται και με τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρατε τη Γερμανία Τώρα το, άλλο το οποίο είπατε έχουμε κάποιες άλλε ενδείξεις για την ΕΕΠ, την Αμερικανική, οι άλλε υπηρεσίε οι οποίε ε, έχουν διεισδύσει σε υπολογιστέ Ευρωπαίων. με ναι, διάφορες τεχνικές ή ιούς, οτιδήποτε, μποτνίξ. Ε, τι, τι, σε τι κατάσταση είναι τα πράγματα τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Λέει ο Πρόεδρος. Κύριε Μορβέ. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ όλες για αυτά τα, τα, το υπέροχο που έχει επιτελέσει. Εγώ να το εξή σας πω. Σε φιλελευθεροπολικό σε μια συνέντευξη. Ποιο Χόρβατ κάτι είπε, ο οποίος ήταν διαφωνών την εποχή του κομμουνισμού. Τώρα είναι σύμβουλος του κ. Μπαρόσο για το μέρο τη Βουλγική Ένωση. Και όταν ρωτήθηκε, τι γνώμη έχετε για το σκάνδαλο Σνόντεν, απάντησε, Ανησυχώ, ανησυχώ, γιατί συνέχεια παρακολουθούν το τηλεφωνό μου. Γινόταν αυτό συνέχεια στον κομμουνισμό. Ούτε αυτό ήταν σωστό, λέει ο δημοσιογράφος. Όχι, απάντησε. Δεν ήταν σωστό. Ούτε βέβαια όμω είναι σωστό να έχουμε ε, τρομοκρατικές επιθέσεις. Δηλαδή ήθελε να πει ότι δεν έχει τίποτα να κρύψει. Κλασική αντιμετώπιση, κλασικό επιχείρημα. Αυτό το έχω διαβάσει πολύ, το έχουμε ακούσει πολλές φορές. Είναι κλασική απάντηση το θέμα, όμως δεν είναι αν κανείς έχει να κρύψει κάτι ή όχι. Το θέμα είναι κατά πόσο μια κυβέρνηση ελέγχει τους ε, πολίτες, αντί να ελέγχουν οι πολίτες την κυβέρνηση. Εγώ να σας πω, εσείς τι λέτε, πώς το, τα μεν σχετίζονται με τα δε. Αυτή η μαζική παρακολούθηση, πώς επιδρά επί των ε, κινημάτων για κοινωνική δικαιοσύνη και βέβαια η προφανής ερώτηση τι τα κάνει αυτά τα δεδομένα ο μεγάλος αδελφός με τη βοήθεια αυτών των συστημάτων έχουν πει οι Αμερικανοί ότι μπορούν να, να, να αποτρέψουν καμιά εικοσαριά, πενταριά ξέρω εγώ πόσες επιθέσεις τρομοκρατικές. Τι λέτε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σα, πρόεδρε, θέλω να σου πω το εξή. Όταν κανείς ακούει τέτοια πράγματα αισθάνεται ανίσχυρος. Και ακριβώ είναι πάρα πολύ ευχάριστο το ότι έρχονται προσκεκλημένοι μας και μας προβληματίζουν σχετικά με το τι μπορεί το Κοινοβούλιο να κάνει για όλα αυτά, τι μπορεί να κάνει για αυτούς τους καταγγέλλοντες. Πώς τους αξιολογούμε αυτούς τους καταδότες, τους θεωρούμε κάτι σαν κατασκοπούς. Τι είναι αυτό, μια νέα εποχή για τα θεμελιώδη δικαιώματα. δεν θέλουμε αυτές οι δραστηριότητες να γίνονται παρά μόνο για την τρομοκρατία. Επομένως, αφού δεν ισχύει αυτό, τι γίνεται. Τέλος, για πέστε μας. Ποιο είναι το κόστος αυτών των προγραμμάτων. πιστεύω ότι η τεχνική άποψη είναι τεράστια αυτή η προσπάθεια που γίνεται και γι' αυτό και θέλω να μας πείτε ποιο είναι το κόστος που συνεπάγεται. Και με όλα αυτά τα συστήματα παρακολουθούσαμε ένα μήνα τον Άσαντ και παρόλα αυτά τις φαγές που διέπραξε εκεί γύρω γύρω από τη Δαμασκό δεν μπορούσαμε να τα αποτρέψουμε. Τι υπάρχει δηλαδή κάποιο είδους τέτοια ε, μόνιμη κατάσταση κατά την οποία υπάρχει αυτή η γενική, η μαζική συλλογή δεδομένων. Είπαμε, ξεκίνησε αυτό το Σεπτέμβριο του 2001. Αλλά βέβαια είχαμε κάποιο είδους αποφάσεις που όλοι τις ενέκριναν κάπως κάπου. επιχειρήσεις, διάφορες υπηρεσίες έχουν εδώ συνεργαστεί για να γίνονται αυτές τις παρακολουθήσεις. Ποια είναι η γεωγραφία αυτής της ε, συνεργασίας. Φτάνουμε από τη συνεργασία στον ανταγωνισμό μεταξύ του. Τι γίνεται με αυτές τις πληροφορίες και όσον αφορά του ελέγχου πότε δεν υπάρχει κοινοβουλευτικό. δεν υπάρχει κυβερνητικό έλεγχο. Ό,τι θέλει κάνει η κυβέρνηση. Οι υπηρεσίες συνταλλάσσουν τα δεδομένα, ε, κάθε κυβέρνηση ε, βρίσκει τις, ε, τα δεδομένα στην υπηρεσία πληροφοριών που κληρονομεί, τα χρησιμοποιεί όπως θέλει. Τι είναι αυτό το βαθύ κράτος. Είναι η, βαθιά καρδιά όπου εκεί χτυπάει <laughs> σαν η καρδιά της κυβέρνησης. Υπάρχει εδώ πέρα συνενοχή, οπωσδήποτε. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Σέντσιν. Το 70% των Ευρωπαίων έχουμε εδώ μια στατιστική που λέει ότι τα προσωπικά του δεδομένα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς διαφορετικού από αυτούς του οποίους η συλλογή του αρχικά εστόχευε. Φυσικά και είναι προφανής αυτονόητος ο φόβος για τέτοιες εξελίξεις. Ο κ. δεν έχουν λόγο οι Αμερικανοί να φοβούνται, διότι το πρόγραμμα αυτό δεν ισχύει για τους Αμερικανούς. Δεν εφαρμόζεται για τους Αμερικανούς. Και η Γαλλία δεν υπήρξε καμία αντίδραση όσον αφορά ε, την πληροφορία ότι υπάρχει παρακολούθηση. Τι τώρα προβληματίστηκαν οι Γάλλοι για την παρακολούθηση αυτή ε, ε, δεν αφορά μόνο τους ξένους. Και επίσης για τον κύριο Απλουδάου. Σε τι βαθμό θεωρείτε εσείς ότι αυτή η μαζική παρακολούθηση που επικαλείται γίνεται εξυπηρετεί την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και σε ποιο βαθμό εξυπηρετεί άλλους σκοπούς που είναι παντελώς άσχετοι με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Μήπως είναι απλώς κάτι σαν πρόφαση για να πάμε σε έναν κόσμο που θα είναι σαν το 1984 Orwell. Uh, we've heard from Mr. Applebaum that... Ο κύριος Μπρόντ, από τον κύριο Applebaum ακούσαμε ότι παρακολουθείται κόσμος και δεν έχουμε μόνο υπόπτους τρομοκράτες και παρακολουθείται και ο ίδιος απλώς και μόνο γιατί είναι δημοσιογράφος που κάνει έρευνα. Δεν ξέρω αν αυτό ισχύει και για ακτιβιστές. Με άλλα λόγια το ερώτημά μου είναι ποια είναι τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται. Και από εκεί και πέρα, τα στοιχεία αυτά διατηρούνται από τις υπηρεσίες ασφαλείας ή παραδίδονται στις κυβερνήσεις οι οποίες μπορούν κάλλιστα μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν για εσωτερικούς σκοπούς. Χρησιμοποιούνται για την ασφάλεια των θέσεων εργασίας του δημοσίου τομέα, που συνδέονται με οργανώσεις ή ε, ε, θέματα τα οποία δεν ε, θεωρούμε σημαντικά. Και τι γίνεται με τους ανθρώπους που γίνονται πληροφοριοδότες. Μπορεί να είναι και οι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να συνδέονται με, την, με οικογενειακούς δεσμούς ή για τυχαίου λόγου με του ανθρώπους οι οποίοι δίνουν πληροφορίες. Χρησιμοποιούνται τα στοιχεία λοιπόν για να χρησιμοποιηθούν κατά των αντιπάλων του όπως συνέβαινε στο παρελθόν ή συμβαίνει και σήμερα. Τα δεδομένα αυτά μήπως χρησιμοποιούνται όχι μόνο για να μελετούν άτομα και οργανώσεις οι οποίες δεν είναι και τόσο επικίνδυνες, αλλά μήπως χρησιμοποιούνται και για να παρενοχλήσουν ανθρώπους ή και τις ζωές τους και οργανώσεις. Ε, έχουμε κάποιες αποδείξεις για τα στοιχεία αυτά στις εφημερίδες. Μήπως οι υπηρεσίες ασφαλείας μιας χώρας, ε, και ίσως και αυτό είναι πολύ επίκαιρο, διαβιβάζουν εσκεμμένα, παραποιημένα στοιχεία για να μειώσουν ε, στρατιωτική δράση, όπως γίνεται για παράδειγμα με τα όπλα μαζικής καταστροφής στο Ιράκ. Και μία πιο ίσως ε, τολμήρη ερώτηση, πώς γνωρίζουν αυτοί που παρακολουθούνται ότι παρακολουθούνται. Και τέλος, πώς θα μπορούσαμε να διατυπώσουμε την νομοθεσία κατά τρόπον ώστε να επιτρέπεται νόμιμη παρακολούθηση για σοβαρά υπόπτους ε, τρομοκράτες και ε, ταυτόχρονα να μην επιτρέπει την παράνομη παρακολούθηση. Ο κύριος Τόρβαλτς για δύο λεπτά. Αυτή είναι μια ανεσυνήθιστη κατάσταση. Στην 11η Σεπτεμβρίου ήμουν δημοσιογράφος, ε, ήμουν στη Νέα Υόρκη και πήρα ένα ταξί και πήγα στο σημείο 0. Και μετά για τέσσερα περίπου χρόνια έγραφα άρθρα για το τι συνέβη. Κάποιες αντιδράσεις ε, ήταν πιο ήπιες, κάποιες άλλες ήταν μέχρι και ιστερικές. Και πρέπει να πω ότι μετά από αυτό το περιστατικό όλες οι υπηρεσίες πληροφοριών της δύση παρακολουθούν στο βαθμό που μπορούν με τα μέσα που διαθέτουν και χωρίς καμία νομοθεσία ε, που να μπορεί να του ελέγξει. Για παράδειγμα, στον κυβερνοχώρο δεν έχουμε εθνικά σύνορα. Δεν μπορεί κανεί να πει ότι αυτό είναι ο κυβερνοχώρο τη Σουηδία και αυτό των ΗΠΑ. Και φυσικά έγινε διότι είχαν τη δυνατότητα να το κάνουν. Έχουμε λοιπόν οι ε, μη ε, οργανώσεις πληροφοριών, υπηρεσίες πληροφοριών της Δύση, που ε, κάνουν παρακολουθήσεις. Θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας και να μου πείτε κατά πόσο θεωρείτε ότι το πρόβλημα είναι παρόν και τη σήμερα ημέρα. Ο κύριος Μποργέτσιο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι είμαστε λίγο υποκριτές εμείς οι πολιτικοί αλλά και οι υπηρεσίες πληροφορίας είναι υποκριτικές, διότι διότι αποκαλύπτονται αυτά τα σκάνδαλα, αποκαλύπτονται αυτές οι πληροφορίες με ανησυχητικούς τόνους και λένε ότι πρόκειται για κάτι το οποίο δεν μπορούμε να προβλέψουμε. Αυτή είναι η φιλοσοφία της νέας παγκόσμιας τάξης η οποία εκφράζεται ακόμα και φυσικά στα πλαίσια του πλήρους ελέγχου των πληροφοριών, των ατόμων και εγώ θα ήθελα να φτάσω και, δεν θα ήθελα να φτάσω και μέχρι και τις σκέψεις, ελέγχα εδώ αυτά που σκεφτόμαστε. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω ε, στους δύο μιλητές εάν από την εις και σοβαρή ανάλυση που έκαναν όχι μόνο από τεχνική σκοπιάς επί του ζητήματος, δημιουργήθηκε το εξής ερώτημα. Ποια στοιχεία ε, βρήκαν ως απάντηση σε αυτό που θα ρωτήσω. Το στοιχείο το οποίο χαρακτηρίζει όλα όσα ανακύπτουν από το σκάνδαλο το οποίο αποκαλύφθηκε από τις εφημερίδες και από τους ε, ερευνητέ δημοσιογράφους ε, είναι στην πραγματικότητα μια μυστική δύναμη διότι αυτό το οποίο προκύπτει κατ' επανάληψη είναι ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών ανταλλάζουν πληροφορίες η μία με την άλλη, αλλά τελικώς δεν ξέρουμε πού καταλήγουν αυτά τα στοιχεία και πώς χρησιμοποιούνται. Σίγουρα έχουν τεράστιες συνέπειες στην οικονομική και χρηματοπιστωτική πραγματικότητα, αλλά προς ποια κατεύθυνση και σε ποιες περιπτώσεις. Με ποιο στόχο ε, συνέβη όλο αυτό. Ποιος ήταν ο αντικειμενικός σκοπός. Και αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε ότι κάποιες πολύ σημαντικές αποφάσεις λαμβάνονται από οργανισμούς οι οποίοι είναι είτε εν μέρη είτε απόλυτα μυστικοί, από την Bilderberg μέχρι το άλλο άκρο. Ε, μήπως λοιπόν η αναλογία αυτού του παγκοσμιοποιημένου ελέγχου των πληροφοριών υπόκειται στα συμφέροντα μυστικών δυνάμεων που καθορίζουν τις αποφάσεις οι οποίες ε, ε, είναι κατεπίφαση δημοκρατικές. Ευχαριστώ. Όσο συμβαίνει συνήθως στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, οι συνάδελφοι που ζήτησαν το λόγο είναι πάρα πολλοί και εμείς έχουμε προγραμματίσει αυτή τη βιντεοδιάσκεψη με τον τρίτον ομιλητή μας ε, σήμερα, τον Άλαν Ρος Πρίτζερ, τον αρχισυντάκτη της Guardian, στις 4.30 και είναι πολύ συγκεκριμένος και ο χρόνος, η διάρκεια της ε, βιντεοδιάσκεψης αυτής θα διαρκέσει μόνο μισή ώρα. Γι' αυτό ακριβώς προτείνω να... Α, έχουμε ήδη τον ομιλητή μας. Ίσως θα μπορούσαμε να ακούσουμε κάποιες απαντήσεις πρώτα από τους προσκεκλημένους μας, ε, τον κύριο Φολορού και τον κύριο Άπελμπαουμ, αλλά όχι, να πάμε απευθείας στον ε, τρίτο ομιλητή μας, τον κύριο Ρόους Πρίτζερ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Σας ευχαριστούμε για αυτή τη μισή ώρα που θα μας αφιερώσετε και σας ευχαριστούμε που είστε διατεθειμένους να συζητήσετε μαζί μας. Ε, για να μας πείτε τις απόψεις σας με βάση τα όσα κάνετε και ως αρχισυντάκτης της Guardian. και να σας καλωσορίσω όπως έκανα και με τους προηγούμενους ομιλητές και να υπενθυμίσω σε όλα τα μέλη εδώ στην αίθουσα ότι η Guardian ήταν αυτή η οποία δημοσίευσε φέτος το καλοκαίρι ε, τη συνεργασία μεταξύ της NSA, της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφάλειας και της ε, ε, GCHQ, το πρόγραμμα Tempora, το PRIS και πιο πρόσφατα την υπόθεση Μιράντα, μάλιστα την υπόθεση Μιράντα 2, διότι υπήρχε και μια θρηλυκή Μιράντα 1 το, η δεκαετία του 60 ε, από το Αμερικανικό Ανώτατο Δικαστήριο. Έχουμε λοιπόν ε, τη μαρτυρία εδώ του κύριου Ρούς Πρίτζερ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Εκτιμούμε ιδιαίτερα το έργο σας. Θα λάβετε το λόγο. Σας παρακαλώ ένα τέταρτο ώστε να έχουμε και λίγο χρόνο να τεθούν κάποιες λίγες ερωτήσεις πριν δώσουμε το λόγο στους ε, υπόλοιπους ομιλητές, ε, τους κυρίους Φολεοχού και τον κύριο Άπελμπαουμ για να απαντήσουν ε, στις ερωτήσεις που τους ετέθησαν. Κύριε Ρος Πρίτζερ, έχετε το λόγο. Thank you and thank Ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ που με καλέσατε να συμμετάσχω στη συζήτηση αυτή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Θα προσπαθήσω να καλύψω τρεις τομείς. Πρώτον, πέρα από το ύφο τη φύση της συζήτησης, θα προσπαθήσω να σας ενημερώσω ε, για την ε, έρευνα αυτή και το ρεπορτάζ και το ρόλο που θεωρώ εγώ ότι θα πρέπει να διαδραματίζουν οι νομοθέτες και τα κοινοβούλια το συνολικό πλαίσιο, περί τίνος πρόκειται και γιατί είναι ε, σημαντικό αυτό. Κάτι που ερευνάτε κι εσείς, δηλαδή κάτι νέο που έχει ανακύψει στις υπηρεσίες πληροφοριών και αυτό είναι η μαζική παρακολούθηση ολόκληρων πληθυσμών, φακέλωμα ουσιαστικά, ε, πληθυσμών ολόκληρων. Αυτό είναι κάτι το καινοφανές κατά την άποψή μου. Δεν έχει συζητηθεί επαρκώς είναι κάτι το οποίο πρέπει να συζητηθεί και αυτό το λένε όλοι αρχής γενομένης από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτικών και των Πολιτιών και προς τα κάτω ε, οι υπόλοιποι πολιτικοί όλοι λέγουν ότι θα πρέπει να συζητηθεί και γι' αυτό κάναμε το ρεπορτάζ αυτό και είναι σημαντικό το γεγονός ότι ορισμένες χώρες προσπαθούν αυτό να το καταστήλουν, να το πνίξουν. Ε, να σας πω δύο λόγια για το πώς προέκυψε όλη αυτή η ιστορία και πώς προσπαθούμε εμείς να κάνουμε το ρεπορτάζ, να αναφέρουμε, να αποκαλύπτουμε αυτά τα πράγματα και ποιες είναι οι ευθύνες και οι προκλήσεις ε, που συνδέονται με αυτά. Μέσα Μαΐου περίπου, είναι γνωστό αυτό, μας προσέγγισε ο Έντουαρτ Σνόουντεν. Και είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι μας προσέγγισε διπλά, όχι μόνο το μεμονωμένο δημοσιογράφο, το Greenwald, το Glenn, ο οποίος, αν θέλετε, είναι τμήμα και του Guardian, αλλά και ε, γενικότερα της νέας ψηφιακής ε, ε, σφαίρας πληροφόρησης. Είναι blogger δηλαδή, δεν είναι κλασικός δημοσιογράφος. Ο Glenn Greenwald είναι δικηγόρος, δημοσιογράφος και blogger. Ε, έχει μια διπλή ιδιότητα λοιπόν και αυτόν προσέγγισε ο Σνόουντεν γιατί έγραφε ε, τόσο υπεύθυνα και τόσο έγκριτα και τόσο πληροφορημένα για το αντικείμενο αυτό. Και στο πρόσωπό του ο Σνόουντεν αναγνώρισε κάποιον που του είχε εμπιστοσύνη και ήξερε ότι θα τα αναφέρει σωστά. Ε, επίσης, απευθύνθηκε στην εφημερίδα The ε, Guardian που φτάνει σε 80 εκατομμύρια ε, υπολογιστές το μήνα. Ε, είναι ένα μεγάλο φόρουμ. Ο Glenn Greenwald είναι και τμήμα αυτού του νέου κόσμου και τμήμα της εφημερίδας Guardian. Το ρεπορτάζ λοιπόν και το άρθρο ήταν περίπλοκο να γραφεί ακριβώς λόγω ε, του αντικειμένου για το πώς παρακολουθούνται οι επικοινωνίες και πώς μπορούν οι υπηρεσίες και τα κράτη να μπαίνουν πραγματικά μέσα στα email, στις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, σε μηνύματα, σε κείμενα. Και αυτό είναι πρόβλημα για τους δημοσιογράφους και είναι από τα θέματα που εμείς διερευνήσαμε, εάν και κατά πόσον η ίδια η δημοσιογραφία ε, και η εμπιστευτικότητα των πηγών ε, μπορεί να είναι δεδομένη σε αυτή τη νέα εποχή. Ο Greenwald είναι Αμερικανός πολίτης, ζει στο Ρίο και η εκδοτική ομάδα είναι στη Νέα Υόρκη, στο Ρίο Ιανέρο, στο Χονγκ στη Ρωσία ε, και στο Λονδίνο συγκεντρώνονται πληροφορίες και η κατάσταση αυτή γεννά πολλά προβλήματα μεταξύ αυτών και νομικά. Δηλαδή υπάρχουν διαφορετικές νομοθεσίες στις Ηνωμένες Πολιτείες και διαφορετική νομοθεσία στο Λονδίνο για παράδειγμα. Εξετάσαμε το υλικό, αλλά και αυτό είχε να κάνει με προβλήματα ασφαλείας. Δηλαδή πώς μπορεί κανείς με τρόπο ασφαλή να εξετάσει αυτό το υλικό χρειαζόταν και υψηλή κρίση ε, από την εκδοτική ομάδα ε, ως προς την ευθύνη που έχουμε γι' αυτό και θέλω να πω κάτι σχετικά. Από την αρχή καταλάβαμε ότι δεν θα κάναμε τίποτα, δεν είναι πρόκειτο να κάνει τίποτα που να αποκαλύπτει ονόματα πρακτόρων, ε, που να φέρνει και να διακυβεύει κάποιες επιχειρήσεις, ούτε θα χρησιμοποιούσαμε αυτό το υλικό ως ένα ε, δόλο μας πούμε, για να ψάξουμε να βρούμε νέες ε, ιστορίες και νέες έρευνες. Το ξέρει και η Βρετανική κυβέρνηση. Ε, δράσαμε με μεγάλη ευθύνη και κατά 90% του ρεπορτάζ είχαμε ειδοποιήσει τις κυβερνήσεις και τις αλόγου υπηρεσίες. Ακούσαμε και την απάντησή τους και νομίζω ότι πραγματικά μας διέκρινε πολύ μεγάλη ευθύνη στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάσαμε την ιστορία αυτή. Κάποια στιγμή προσκρούσαμε σε νόμους. Το είπα και προηγουμένως. Η νομοθεσία των διαφόρων κρατών κάνει αυτό του είδους το ρεπορτάζ είτε δύσκολο είτε ανέφικτο είτε επιτρεπτό ανάλογος. Και είναι προφανές ότι οι νομοθέτες που κάθονται και ακούνε τώρα αυτά τα πράγματα τουλάχιστον δεν μας βρήκαν σύμφωνους. Ε, σε δύο τουλάχιστον περιπτώσεις συγκρουστήκαμε ε, πάρα πολύ γιατί χρησιμοποίησαν την ε, νομοθεσία κατά της τρομοκρατίας για να συλλάβουν και να κρατήσουν τον David Miranda που ήταν ένα τμήμα της ομάδας του Guardian ε, και η άλλη δυσκολία ήταν η άμεση απειλή ε, που εξαπέλυσε η Βρετανική κυβέρνηση ότι θα χρησιμοποιήσουν τον νόμο για να μας εμποδίσουν να ε, το δημοσιεύσουμε και μας απείλησαν μέχρι ότι θα μας καταστρέψουν το υλικό. Γι' αυτό τώρα συνεργαζόμαστε με Αμερικανούς εταίρους διότι η Αμερικανική νομοθεσία και μάλιστα η πρώτη το πρώτο εδάφιο του συντάγματος ε, δίνει προστασία πολύ μεγαλύτερη από ό,τι ε, στη Βρετανία ή στην Ευρώπη. Το άρθρο 10 ε, το, το δικό μας δεν είναι το ίδιο με το πρώτο άρθρο του Αμερικανικού συντάγματος, First Amendment. Δεν μπορεί κανείς εκ των προτέρων να κάνει λογοκρισία στην Αμερική, να εμποδίζει να δημοσιεύεται κάποιο υλικό. Έχουμε λοιπόν ένα νέο περιβάλλον στο οποίο πρέπει να εργαζόμαστε ως δημοσιογράφοι και ε, προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε την καλύτερη νομική ε, κατάσταση και το καλύτερο νομικό καθεστώς. Όταν ε, τα κράτη θέλουν να μας αποτρέψουν και να μας εμποδίσουν να αποκαλύπτουμε κάποιες καταστάσεις στην Ευρώπη. Έτσι λοιπόν προέκυψε αυτό το ρεπορτάζ, έτσι προσπαθούμε να εργαστούμε με βάση το υλικό που έχουμε Υπήρξαν ζητήματα ασφάλειας των επικοινωνιών και των τηλεπικοινωνιών, ασφάλειας του υλικού. Όπως προσπάθησα να τονίσω, ήταν ομαδική αυτή η δουλειά, συλλογικό το εγχείρημα. Πολλοί οι ρεπόρτερ, οι δημοσιογράφοι, οι συντάκτες που συνεργάστηκαν με τον Glenn Greenwald και χρησιμοποίησαν τις γνώσεις του και την πραγματογνωμοσύνη του μαζί με τις ε, συντακτικές εκδοτικές ε, ε, δυνατότητες. Είχαμε υποστήριξη τεχνολογική, είχαμε υποστήριξη νομική για να κάνουμε σωστή δημοσιογραφία προς το όφελος του κοινού. Και σε τελική ανάλυση <laughs> θα έχουμε πολύ μεγάλες ε, οικονομικές υποχρεώσεις και πολύ μεγάλα έξοδα απέναντι σε δικηγόρους που πρέπει να πληρώσουμε για να ε, υποστηρίξουμε όλη αυτή την προσπάθεια. Η New York Times και η Republica συνεργάζονται για να μπορέσουμε να βγάλουμε όλο αυτό το υλικό και να το δημοσιεύσουμε. Αλλιώς στο Ηνωμένο Βασίλειο κάτι τέτοιο είναι αδύνατο. Να σας πω για ποιο λόγο Αξίζει όλη αυτή η υπόθεση, αυτή την προσπάθεια, με όλες αυτές τις δυσκολίες, όλες αυτές τις προκλήσεις και τα προβλήματα. Γιατί είναι σημαντικό πραγματικά μια εφημερίδα να κάνει ένα τέτοιο ρεπορτάζ με τρόπο υπεύθυνο πάντα. Επανέρχομαι ε, εκεί από όπου ξεκίνησα. Στον παλιό κόσμο, το προηγούμενο κόσμο, κατασκοπία έκανε μια χώρα κατά της άλλη. Ήταν μια στοχευμένη δραστηριότητα με πολύ στοχευμένες και υψηλές ε, τεχνολογίες και τεχνικές για να κατασκοπεύει μία χώρα την άλλη. Τι συνέβη όμως το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία 10-15 χρόνια. Έχουμε περάσει σε έναν άλλο κόσμο όπου συνεργάζονται ε, χώρες και εταιρείες... και αρχίζουμε να τα αντιλαμβανόμαστε αυτά, να τα υποψιαζόμαστε μέσω των ε, γράφων του Σνόντεν. Υπάρχει μαζική επιδρομή ε, και παρακολούθηση οποιοδήποτε πολίτη που χρησιμοποιεί ψηφιακή τεχνολογία. Υφίσταται κάποιο είδους παρακολούθηση. Αυτό πιστεύω ότι δεν επιτρέπεται να συμβαίνει χωρίς προότερη συνένεση του ενδιαφερομένου και των πληθυσμών αυτών. Δεν μπορεί κανείς να συνενεί ε, χωρίς να έχει την απαραίτητη πληροφόρηση. Χωρίς τη σημερινή συζήτηση που κάνετε εσείς στο κοινοβούλιο σας. Θα πρέπει να έχετε ε, πληροφορίες για να βασιστείτε σε αυτή τη συζήτηση. Δεν μπορεί ταυτόχρονα οι κυβερνήσεις να προσπαθούν ε, να εμποδίζουν τις εφημερίδες να δημοσιεύουν και ταυτόχρονα να γίνεται και η συζήτηση. Χαίρομαι που ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο κύριος Ομπάμα, και χτες μάλιστα, είπε ότι είναι απαραίτητη η συζήτηση αυτή επειδή δεν μπορεί να ε, κάνει κάποιο κάποια πράγματα, δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να προσπαθήσει να τα κάνει. Όταν κάποια πράγματα έχουν πάει στραβά, θα πρέπει αυτό να καταδεικνύεται. Δεν μπορεί να γίνει αυτή η συζήτηση χωρίς γνώση και πληροφόρηση όμως. Ξέρω ότι πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Μεταξύ της ασφάλειας, του του ιδιωτικού βίου και τη ελευθερίας του λόγου, αλλά και τη ελευθερίας του συνεταιρίζεστε, αλλά και της δυνατότητας να καταγγέλει κανεί. Όλα αυτά όμως θα πρέπει να σταθμιστούν. Και αυτό το οποίο τελικά γίνεται είναι ότι η πτυχή ασφάλεια αυτή κατησχύει. Οπότε στι συζητήσει και επαφές που με τις κυβερνήσεις βεβαίως ο παράγων ασφάλεια λέω δεν θα έπρεπε να το δημοσιεύσετε αυτό Έχουμε κάποιους κορυφαίους παλιού που είπαν ότι εντάξει έγινε κουβέντα, τώρα κόφτε το, βουλώστε το. Για μένα όμως το θέμα δεν είναι το κράτος. Δεν μπορεί το κράτος να λέει στον δημοσιογράφο πότε να το βουλώσει. Ε, αυτή η προβληματική θα πρέπει να ξεκινήσει τώρα. Αυτή η προβληματική η οποία είναι αναγκαία ούτως ώστε να μπορέσουμε να ελκύσουμε τη συνένεση του κόσμου για το εάν θα χρησιμοποιούνται αυτά τα νέα μέσα παρακολούθησης όλα αυτά τα οποία επηρεάζουν ε, ό,τι ηλεκτρονικό κάνει κανείς. Δεν μπορεί να σε να το, τον τύπο, οπότε και εγώ δεν μπορώ παρά να χαιρετήσω τη σημερινή συνάντηση. Να τη θεωρήσω κάτι πάρα πολύ θετικό. Και πέρα θα πρέπει πας νομοθέτης εις πάσα χώρα στον ελεύθερο κόσμο, όλοι αυτοί οι οποίοι πρόκειται να είναι στόχος αυτών των ε, τόσο επιθετικών μορφών ε, παρακολούθηση να το λάβουν υπόψη. Γιατί υπάρχουν ε, οι μηχανικοί οι οποίοι τα φτιάχνουν αυτά τα gadget και αυτοί πάντοτε θα είναι μπροστά ε, από τον νομοθέτη. Άρα είναι δουλειά του Κοινοβουλίου να κάτσει και να σταθμίσει όλους αυτούς τους παράγοντες και να δει κατά πόσο αυτή η εποπτεία, η παρακολούθηση ε, έχει νόημα, πώς γίνεται, εγκριτό και παραβίστο κλπ. και να δούμε και το κατά πόσο όλα αυτά έχουν γίνει, έχουν κηρυθεί στο παρελθόν, αν έχουν νόημα, αν είναι χρήσιμο. Οπότε σας, παρα... ευχαριστώ που με καλέσατε να μιλήσω και ε, ήθελα αυτά να ξεκαθαρίσω για την προβληματική. Το ότι θα πρέπει να υπάρχει υπεύθυνη δημοσιογραφία και επίσης ότι θα πρέπει ε, ο κάθε νομοθέτης να προστατεύει τέτοιου είδους ε, δημοσιογραφία και ούτως ώστε να μπορούμε να συζητούμε αυτό το υλικό, το υλικό αυτό το οποίο εκθέτουμε ε, το, και το εκθέτουμε σε το, το ξυμπροστιάζουμε παρά το ότι υπάρχουν προβλήματα από τον νόμο, ε, ότι ρισκάρουμε, αλλά θα πρέπει ο νομοθέτης να προστατεύσει την υπεύθυνη δημοσιογραφία και να ενθαρρύνει τέτοιου είδους προβληματική. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, κύριε. Σας ευχαριστούμε για το έργο σας εκεί για, για, για τον πρωτοπόρο ρόλο που παίζεται ή στον Guardian που προβάλλεται αυτές τις αξίες που και εμείς α, ασπαζόμεθα και ακριβώ ξεμπροστιάζεται αυτή η κατάσταση που τώρα συζητούμε και σας ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ σε αυτή την τηλεδιάσκεψη σας ευχαριστούμε για την εισφορά σας ή σε αυτήν την έρευνα ή σε αυτήν την συζήτηση οπότε δεν μπορώ παρά να σας συνεχίσω τώρα ότι θα έχουμε και ένα δεύτερο δεύτερο, δεύτερο πάνελ άλλους τρεις ε, προσκεκλημένου στι 5 ώρα που θα συζητήσουμε τι γίνεται με το σύστημα Ε, Και επίση έχουμε ε, εισηγητή τον Σμιτ, τον Κοέλιο και τον Ντάνκαν Κάμελ που είναι και εκείνο ένα ε, προσκεκλημένος εκπροσωπή ΜΜΕ. Σα προτείνω τώρα να λάβουμε υπόψη το ότι έχουμε πίεση χρόνου και επίσης η τηλεδιάσκεψη έχει συγκεκριμένο χρόνο που μπορεί να ε, έχει τη σύνδεση. Άρα να πούμε στον κύριο Ράσμπετζερ ε, τις ερωτήσεις που έχουμε και κατόπιν να απευθυνθούμε στους ε, άλλους ομιλητές μας, τον κύριο Φολερού και τον κύριο Απελμπαμ και εκείνοι μετά να απαντήσουν πριν αρχίσει το δεύτερο πάνελ. And we will be thanking you for being here and moving on to our previous guests for them to react to the questions that we already... Πρώτα επομένως με τηλεδιάσκεψη και κατόπιν στους λοιπούς. Οπότε πάμε πρώτα στον κύριο Μωράες. Σας ευχαριστώ κύριε που ήρθατε εδώ. Όλοι γνωρίζουμε ότι ήταν πρωταγωνιστής η εφημερίδα Guardian για την ιστορία με αυτόν τον καταδότη. Και βέβαια φυσικά και όλα αυτά γίνανε με ρίσκο για την εφημερίδα. Έχω μια σύντομη ερώτηση. Στο Στρασβούργο θα υπάρξει δήλωση όσον αφορά την υπόθεση Μιράντα. Ήλκησε την προσοχή όλου του κόσμου. Πρόκειται για την αντιτρομοκρατική νομοθεσία της Αγγλίας. Έγινε λάθος χρονή της νομοθεσίας εις βάρος κάποιου που κατήχε πληροφορίες. Πληροφορίες που σχετιζόντουσαν με την εφημερίδα σας. Επίσης είχαμε και την κατάσχεση και των σκληρών τη της εφημερίδας που τα είπατε όλα αυτά. Εγώ σα ερωτώ, ω διευθυντή τη εφημερίδα, ω υπεύθυνο του τα είπατε όλα αυτά. Είπατε τι έπαθε η εφημερίδα σα. Αλλά για πετε μα, ποιε είναι οι επιπτώσει επί τη δημοσιογραφία γενικώ ή συγκεκριμένα επί ημών, συγκεκριμένα επί τη ελευθερία του τύπου. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση είναι. Είπατε, αναρωτηθήκατε ποιο θα είναι το επόμενο βήμα. Είπατε ότι σας είπαν. Εντάξει, το κουβεντιάσατε, τώρα σκάστε. Ναι, θα πρέπει όμως να πιεστεί ο νομοθέτης κάτι να κάνει. Τι θα κάνουμε, να αλλάξουμε την νομοθεσία ή να αναζητήσουμε ή να, να, να, να, προσδοκώ, να προσδοκάμε περισσότερους καταδότες. Και τώρα θα είναι να δώσω λόγο στον κύριο Φως, Άλμπρεχτ, παρακαλώ, ένα λεπτό έκαστος, ούτως ώστε ο προσεκλημένος μας να μπορέσει να απαντήσει και κατόπιν οι άλλοι δύο μιλητές. Σύντομα παρακαλώ, αλλιώς δεν θα τα καταφέρουμε. Σύντομα. we, are our schedule. make it short. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Ακούστηκε και αναφέρθηκε η ελευθερία του τύπου, η ελευθεροτυπία. Δεν έχετε την αίσθηση ότι και η ελευθεροτυπία έχει κάποια όρια και σταματά εκεί που αρχίζει η γενική ασφάλεια. Ε, και επίσης θα ήθελα να μου πείτε αν έχετε την αίσθηση ότι ο εσωτερικό έλεγχος των μυστικών υπηρεσιών ή ο κοινοβουλευτικός ή ακόμα και ο δικαστικός έλεγχος δεν υπάρχει καθόλου στις μυστικές υπηρεσίες. Και επίση θα με ενδιέφερε να μάθω αν η εφημερίδα Guardian για την πληροφόρηση αυτή χρειάστηκε να πληρώσει για να αποκτήσει αυτές τις πληροφορίες. Ευχαριστώ πολύ. Ένα λεπτό. Η κυρία Νετβέλτ. Ευχαριστώ και σας ευχαριστώ κύριε Ροζ για την πολύ ενδιαφέρουσα συνεισφορά σας αναφερθήκατε σε νομικές κατηγορίες ε, θα ε, ζητήσετε αποζημίωση από την ε, κυβέρνηση που σας υποχρέωσε να καταστρέψετε τους σκληρούς σας δίσκους ή κατέστρεψαν οι ίδιοι τους σκληρούς σας δίσκους. Και επίση υπάρχει ανησυχία μεταξύ των συναδέλφων σας στην Ευρώπη. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι ανησυχούν παρά το γεγονός ότι είναι μικρή αυτή η ανησυχία. Γιατί υπάρχει αυτή η ανάγκη οι δημοσιογράφοι να προστατεύσουν τα δικαιώματά τους. Και τρίτη μου ερώτηση. Θεωρείτε ότι υπάρχει ανάγκη για ευρωπαϊκές ε, νομικές διασφαλίσεις για την ελευθεροτυπία. Όπως είπατε, στις Ηνωμένε Πολιτείε αυτές οι ε, ε, διασφαλίσεις είναι πολύ πιο εύρωστες. Και επίσης μου φαίνεται ότι οι ίδιοι άνθρωποι που είναι αντίθετοι στις συστάσεις της έρευνας Λέβερσον για τους ε, μεγαλύτερους ελέγχους προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ζήτησαν να καταστραφούν οι σκληροί σας δίσκοι. Τι σημαίνει αυτό για τη συζήτηση στις ΗΠΑ. Ε, για ένα λεπτό σας παρακαλώ γιατί καθυστερούμε ο επόμενος ομιλητής και πρέπει να ακούσουμε και τους ε, προλαλήσαντες. Ευχαριστώ. Κύριε Ροσπρίτζερ, μία ερώτηση έχω κι εγώ, ο κύριος Άλμπρεχτ. Αναφερθήκατε σε ένα σύστημα το οποίο δεν θα έπρεπε να επιτρέπει ό,τι επιτρέπει η τεχνολογία να κάνουμε δεν θα έπρεπε να λαμβάνονται όλες οι πληροφορίες από τις τηλεπικοινωνίες. Υπάρχει δυνατότητα να τευθυγραμμίσουμε αυτά με μια ελεύθερη δημοκρατική κοινωνία και την ελευθεροτυπία. Η κυρία Βερζιά, σύντομα σας παρακαλώ. Ναι, κύριε Πρόεδρε, θα είμαι πολύ σύντομη, διότι η ερώτησή μου είναι αντίστοιχη με την ερώτηση της Σοφίνεντβελτ. Είπατε ότι το σύστημα προστασίας των δημοσιογράφων στις ΗΠΑ είναι πιο αποτελεσματικό και το αποδεικνύεται διότι μπορείτε να δημοσιεύσετε στις ε, ΗΠΑ Πολιτείες κάποιες πληροφορίες που δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε στη Μεγάλη Βρετανία και προστατεύονται από πιο αποτελεσματικά μέτρα οι δημοσιογράφοι. Και θα έπρεπε να προστατεύονται οι δημοσιογράφοι. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν έχετε κάποια πρόταση να μας κάνετε ως προς την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, ποια θα έπρεπε να είναι κατά την άποψή σας η προτεραιότητα και πού θα πρέπει να δώσουμε έμφαση. Ευχαριστούμε κυρία Βερσιά. Κύριε Ροσπρίτσερ, σας ευχαριστούμε πολύ και για το χρόνο σας και για τις απαντήσεις που θα μας δώσετε. Καταρχάς θα πρέπει να με συγχωρήσετε. Θα απαντήσω όλες τις ερωτήσεις ε, στα αγγλικά για τις δύο ερωτήσεις που δεν ήταν στα αγγλικά θα μπορούσε κάποιος να με βοηθήσει διότι δεν είχα μετάφραση. Mm. Θα απαντήσω λοιπόν στις ερωτήσεις οι οποίες ετέθησαν στα αγγλικά. Η πρώτη ερώτηση για το τι συνέπεια έχουν για τη δημοσιογραφία αυτές οι ε, παρεμβάσεις. Το γεγονός ότι χρησιμοποιείται ε, η απειλή των κυρώσεων και ε, νομοθεσία τρομοκρατίας. Να σας πω ότι αυτό πραγματικά θα ήταν ανατριχιαστικό. Ε, θα παρακολύσει τη δημοσιογραφία. Υπάρχει ένα ιστολόγιο το οποίο γράφει ένας πρώην πράκτορας της CIA, ε, μπορώ να σας δώσω και τη σχετική διεύθυνση και έλεγε ότι ουσιαστικά ε, προσπαθούν να μας εκφοβήσουν, να σταματήσουν τη δημοσιογραφία αλλά είναι σαν να ρίχνουν άμμο στους τροχούς μας. Αλλά το να μην χρησιμοποιείται η κατάλληλη νομοθεσία και να μας απειλούν για κυρώσεις αναπόφευκτα θα είναι ανατριχιαστικό για τη δημοσιογραφία τώρα. Το τι θα σημαίνει αυτό ε, για τους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν καταγγελίες, τους πληροφοριοδότες, δεν ξέρω ποιους θα θέλαμε να ενθαρρύνει η Δύση να δώσουν πληροφορίες αν υπάρχει κάποιος ο οποίος μπορεί να μας πει ότι υπάρχει μια συμμετρία και μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε να αποκαλύψουμε τα μυστικά του Σνόντεν αλλά όχι των Κινέζων και ότι θα έχουμε Γερμανούς και Ιρανούς πληροφοριοδότες αλλά θα πρέπει να δούμε και τι μήνυμα στέλνουμε. Δηλαδή, εάν δεν επιτρέψουμε για 60 χρόνια στη Δύση να γίνονται καταγγελίες από πληροφοριοδότες γιατί δεν θεωρούμε ότι είναι σωστό, πώς θα ενθαρρύνουμε Κινέζους, Ρώσους, Ιρανούς πληροφοριοδότες να έρθουν να μιλήσουν στην Guardian και να χρησιμοποιήσουν την προστασία που τους προσφέρει, ε, το άρθρο 10 στην Ευρώπη και το πρώτο ε, εδάφιο του Συντάγματος των ΗΠΑ. υπάρχουν κάποιες καταγγελίες για δημοσιογράφους και πληροφοριοδότες οι οποίοι θανατώθηκαν στην Ινδία. Για μένα το γεγονός ότι κάποιος αποφασίζει να δώσει πληροφορίες σημαίνει ότι πρέπει αυτόματα να προστατεύεται. Το να υπάρχει νομοθεσία που μόνο τιμωρεί αυτούς τους ανθρώπους και ε, ακατάλληλη νομοθεσία για να σιωπήσει το έργο της δημοσιογραφίας σημαίνει ότι οι δυτικέ κυβερνήσει θα πρέπει να σκεφτούν τι μήνυμα στέλνουμε με αυτέ τι συμπεριφορέ. Αυτή είναι η απάντηση προ την πρώτη ερώτηση. Τώρα, η επόμενη ερώτηση η οποία τέθηκε στα αγγλικά ήταν κατά πόσον η Guardian θα ε, μηνύσει για την καταστροφή των σκληρών δίσκων. Η απάντηση είναι όχι, διότι αυτό είναι κάτι το οποίο έκανα εγώ ο ίδιος, ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα να μου επιβληθεί μια ποινή η οποία δεν θα μου επιτρέπει να δημοσιογραφώ και, να γνωρίζω ότι, ε, και επειδή γνώριζα ότι δεν πρόκειται να σταματήσει διότι υπάρχουν αντίγραφα όπως ε, έχω ζητήσει από τη Βρετανική κυβέρνηση αλλού ανά τον κόσμο. Επομένως δεν θεωρώ ότι το να καταθέσω μια αγωγή είναι η σωστή λύση. Τώρα, γιατί δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανησυχία για το θέμα αυτό στην Ευρώπη, νομίζω ότι αυτό όλο είναι λίγο ε, διάσπαρτο. Σε κάποιες περιπτώσεις άκουσα στην Ευρώπη συντάκτες ε, και οργανώσεις ελευθερίας ε, του τύπου κάποιες φωνές υποστήριξής μας, αλλά νομίζω ότι αυτό σχετίζεται και με την απάντηση για την ερώτηση για το Ηνωμένο Βασίλειο και τι σχέση έχει το θέμα. Βασικά σημαίνει ότι ο κόσμος δεν ε, σκέφτεται λίγο το ευρύτερη εικόνα. Τα όσα κάνει η δημοσιογραφία σχετίζονται άμεσα και με τη δυνατότητα να μπορέσουμε να έχουμε μια συζήτηση επί του θέματος. Και αυτό μπορεί να έχει σχέση και με την οτροπία μας σε εθνικό επίπεδο και την εμπειρία που έχουμε για την ε, ε, τον έλεγχο που γίνεται στις υπηρεσίες πληροφοριών και τα όσα θα μπορούσαν να συμβούν, τα άσχημα τα οποία θα μπορούσαν να συμβούν, εάν υπάρχει και αυτή η κακή πτυχή της ε, παρακολούθησης. Και νομίζω ότι είναι θέμα νοοτροπίας του κάθε λαού ε, και αυτό διέπει το βαθμό ανησυχίας τους κάθε φορά. Σε κάποιες χώρες έχουν ακουστεί φωνές υποστήριξης, μεγάλη υποστήριξη για τα όσα κάνει η Guardian, για τα όσα κάνει ο Snowden ε, και ο, ο blogger μας. Ε, νομίζω όμως ότι ήταν ε, λίγο διάσπαρτες οι, οι φωνές υποστηρικτικές. Και φυσικά υπάρχει και συγκεκριμένος τρόπος με τον οποίο ανταποκρίνεται το Ηνωμένο Βασίλειο. Τώρα, για τις δικλείδες ασφαλείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ερώτηση που τέθηκε για το θέμα αυτό. Η απάντησή μου είναι ότι εγώ δεν είμαι νομικός. Γνωρίζω ότι υπάρχει το άρθρο 10 στην Ευρώπη, το οποίο έχει ε, ενσωματωθεί και στο Βρετανικό δίκαιο και Το ερώτημα είναι γιατί κατά την άποψη των περισσότερων δημοσιογράφων που γνωρίζω το άρθρο 10 δεν έχει την ίδια βαρύτητα με, την, με το πρώτο εδάφιο του Αμερικανικού Συντάγματος. Ίσως η απάντηση να είναι ότι εμείς δεν έχουμε την ίδια προστασία κατά ε, αυτών των δράσεων και δεν έχουμε την ίδια ελευθερία έκφρασης που υπάρχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως σας είπα, εγώ δεν είμαι νομικός, εκφράζω απλώς την προσωπική μου άποψη ως δημοσιογράφος. Και ένας από τους λόγους για τους οποίους θεωρώ ότι οι δημοσιογράφοι θα πρέπει να ανησυχούν λίγο περισσότερο για τα όσα προκύπτουν από τα ε, ε, έγγραφα του Σνόντεν είναι ότι η δημοσιογραφία αυτή καθεαυτή ε, είναι δυνατικά υπό από αυτές τις αποκαλύψεις. Οποιοςδήποτε λοιπόν έχει τον όλοχο αυτού του υλικού ε, δεν έχει σχέση με το περιεχόμενο των ε, ε, μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αλλά αυτά τα μεταστοιχεία. Ποιος στέλνει email σε ποιον και γιατί. Ποιος είναι αυτός ο οποίος αναζητά κάτι σε ποια μηχανή αναζήτησης. Αυτό είναι τα μεταστοιχεία τα οποία εξόψεως είναι ε, αυλαβή, συλλέγονται σοριδών, αλλά στην πραγματικότητα ε, σου λένε ποιοι δημοσιογράφοι έρχονται σε επαφή με ποιον και ποιες είναι οι πηγές τους. Επομένως η δημοσιογραφία απελείται ε, βαθύτατα από αυτές τις ε, τεχνικές μαζικής παρακολούθησης και έχουμε διαπιστώσει ότι όλα αυτά τα συστήματα μαζικής παρακολούθησης ε, σίγουρα δεν είναι και τα ίδια ασφαλή. Αυτή είναι η ηρωνία αυτού του συστήματος ε, άκουσα ανθρώπους να μου κάνουν κήρυγμα για την ασφάλειά τους όταν οι ίδιοι άνθρωποι που μέχρι τώρα έχουν διαρρεύσει υλικό είναι οι ίδιες οι υπηρεσίες οι οποίες υποτίθεται ότι κρατούν ασφαλή αυτά τα στοιχεία. Όσον αφορά τώρα την ε, τελευταία ερώτηση η οποία τέθηκε στα αγγλικά και ζητώ συγγνώμη που δεν θα απαντήσω τις ερωτήσεις που ήταν σε άλλη γλώσσα, ε, δυστυχώς ε, είναι η Βρετανική μονατροφή, αυτές είναι οι γλυσικές μου δεξιότητες, οι οποίες γνωρίζετε φαντάζομαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το σύστημα του ελέγχου, της εποπτείας στο οποίο αναφέρθηκε κάποιος. Κάποιος ρώτησε αν αυτή η συλλογή δεδομένων σε μαζικό επίπεδο ε, συμφιλιώνεται με την ελεύθερη κοινωνία. Νομίζω ότι η απάντηση αφορά τα συστήματα εποπτείας ε, και κατά πόσον υπάρχει ένας κατάλληλος μηχανισμός για να αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά ή είναι ένας απλός μηχανισμός ο οποίος ε, μας δείχνει λίγο πολύ πώς λειτουργούν τα πράγματα στις ΗΠΑ και σε ποιο βαθμό έχουν δίκιο οι επικροτές τους όταν τους λένε ότι είναι μονόπλευρη η στάση τους ή όταν ε, ε, κάνουν κάποιες πιο αυστηρές επιλογές. Και εγώ πραγματικά δεν γνωρίζω σε ποιο βαθμό η εποπτεία του Κογκρέσου και του Κοινοβουλίου είναι αποτελεσματικές. Ο έλεγχος ε, από αυτή την πλευρά είναι οι νομοθέτες ή είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι δέσμοι των κοινωνιών στις οποίες υποτίθεται ότι ε, προστατεύουν. Δεν ξέρω και τι έγγραφα βλέπουν. Έχουν δει όλα αυτά που έχουμε δει εμείς ή ένα μικρό ποσοστό τους και μόνον. Και το θέμα είναι ότι όλα αυτά τα στοιχεία δεν μας είναι γνωστά. Αυτό το οποίο θα ήθελα λοιπόν να πω στους νομοθέτες, όπως είπα και προηγουμένως, είναι σας παρακαλώ βρείτε τρόπους να προστατεύσετε τη δημοσιογραφία, γιατί η δημοσιογραφία είναι ο μόνος τρόπος για να διεξαχθεί αυτή η συζήτηση, αυτή τη συζήτηση που όλοι θεωρούν πλέον απαραίτητη, αλλά οι κυβερνήσεις οι ίδιες δεν θα ενθαρρύνουν και οι υπηρεσίες πληροφοριών δεν θα θεωρήσουν ότι είναι ευπρόσδεκτη, επομένως μόνο η δημοσιογραφία θα σας δώσει... Ε, μια κατάλληλη και αμερόληπτη εικόνα του, κόνου, του κόσμου αυτού βάσει των στοιχείων που μας δίνουν οι πληροφοριαδόντες. Σας παρακαλώ προστατεύσε μας ως δημοσιογράφους και θεωρήστε ότι αυτοί οι μηχανισμοί ελέγχου ε, θα πρέπει ε, να ε, επανεξεταστούν και να δούνε πώς μπορούν να έχουν κάποια ουσία όπως θα έπρεπε να είναι ουσιαστικοί. Δεν ξέρω ποιο είναι αυτό ο οποίο θα πρέπει να το κάνει. Κατά την άποψή μου, οι νομοθέτε είναι αυτοί και θα πρέπει να βρουν έναν τρόπο να συγκρίνουν το υλικό το οποίο διαθέτουμε εμεί και ε, θα ήθελα να ακούσω και την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το τι θα πρέπει να γίνει με αυτό το υλικό και να το συγκρίνουν με ε, τα στοιχεία τα οποία διαθέτουν και τα στοιχεία τα οποία έχουν δει οι επιτροπές ελέγχου. Διότι έτσι θα έχετε μία αίσθηση του ε, πώς ακριβώς δραστηριοποιούνται οι ελεγκτικοί μηχανισμοί ε, εάν δρούν ανεξάρτητα ή αν και οι ίδιοι έχουν απλώς μια πολύ μεροληπτική εικόνα του τι συμβαίνει. Ευχαριστούμε κύριε Ρώσπιν, Ευχαριστούμε για το χρόνο σας. Τώρα, εάν έχετε την υπομονή να μας ακούσει λίγο παραπάνω, ένα, ένα λεπτάκι μόνο, γιατί δεν θα πρέπει να αφήσουμε απ' έξω τις ερωτήσεις που δεν διατυπώθηκαν ή σε άλλη γλώσσα. Γιατί έχουμε την ερώτηση κύριε κ. που είπε εσείς θα συμβουλεύατε να γίνει ένα βήμα προς το εμπρός από το ευρωπαϊκό επίπεδο του ευρωπαϊκή σκοπιά ώστε να προστατεύσουμε καλύτερα την ελευθερία των ΜΜΕ, την ελευθερία της για την πληροφόρηση αλλά και ο κύριο Αξελφός από τη Γερμανία είπε κάτι συγκεκριμένο ότι έχετε ποτέ αμύψει κάποιον καταδότη πληροφορίε Οπότε, ε, αν δεν έχουμε αντίρρηση, ε, λεφτά για να τα ξαναδιατυπώσουμε αυτά στα αγγλικά. Σα ευχαριστώ. Τρει ερωτήσει είχα κάνει, λέει ο κύριο Βό, στα αγγλικά τώρα. Για τη δημοσιογραφία θεωρείτε ότι δεν θα πρέπει να έχει όρια, ακόμα και αν ζητήματα εθνική ασφαλείας. Θα πρέπει να είναι απεριόριστη η δημοκρατία και ανεξέλεγκτα όλα για τα στοιχεία. Εσωτερικά θεωρείτε δεν θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος ε, στις μυστικές υπηρεσίες από πλευράς κοινοβουλίου ή της δικαιοσύνης. Και το τελευταίο νομίζω απαντήθηκε, ε, ε, χρειάστηκε να πληρώσετε για αυτές τις πληροφορίες. τελευταία απάντηση και σας ευχαριστώ που ήρθατε. Όχι, δεν πληρώσαμε για την παροχή των πληροφοριών. Τώρα το θέμα ελέγχου από το Κοινοβούλιο και από τις δικαστικές αρχές απήντησα προηγουμένως και σε σχέση με το κατά πόσον θεωρούμε ότι υπάρχουν όρια προς όφελος της ασφαλείας και αυτό το είπα στην πρώτη απάντηση ότι εδώ πέρα είναι δυσδιάκριτα τα όρια μεταξύ των διαφορετικών αυτών πτυχών. Αλλά και όταν δημοσιεύουμε κάτι, κάνουμε τη διάκριση μεταξύ του τι είναι απειλητικό, κακό για την εθνική ασφάλεια. Δεν νομίζω ότι περάσαμε τα όρια. Γιατί από την άλλη μεριά υπάρχει και το θέμα της ζωής, της θετικής ζωής αυτών που χρησιμοποιούν την ψηφιακή τεχνολογία και επικοινωνία. Στάθμιση των πτυχών αυτών. Αυτό όμως δεν το κάνουν οι, οι υπηρεσίες πληροφοριών. Λένε δεν θα δημοσιεύσετε τίποτα. Γιατί αν δημοσιεύσετε δεν θα ξέρετε τι να σταθμίσετε γιατί δεν ξέρετε τα θέματα της ε, εθνικής ασφαλείας. Όντως τα θέματα αυτά είναι ε, δύσκολα, είναι δυσδιάκριτη, στάφηση και θα πρέπει κάποιος, όπως η New York Times, όπως ο Guardian και η Washington Post, είναι να είναι υπεύθυνοι κριτές για να μπορέσουν να τα σταθμίσουν. Και θα πρέπει να έχουν σε συνέντευξη με τις υπηρεσίες πληροφοριών, αλλά όχι μόνο με αυτές. Γιατί υπάρχει και η πτυχή των δημοκρατικών ελευθεριών, της δημοκρατίας. Γιατί ε, δεν θα πρέπει να ακούγεται μόνο φωνή των υπηρεσιών πληροφοριών τώρα για τον ε, Βρετανό συνάδελφο. Τον Γάλλο, συγγνώμη, τον Γάλλο. Ή την Γαλλίδα τέλο πάντων. Σας είπα, δεν καταλαβαίνω γιατί το άρθρο 10 δεν θα πρέπει να έχει το ίδιο ειδικό βάρος, τις ίδιες επιπτώσεις ε, θετικές, της προστασίας που θα οραματιζόμαστε. Γιατί στα Βρετανικά δικαστήρια είπαμε ότι είναι πάρα πολύ θετικό το άρθρο 10. Απέβει ένα επιχείρημα πολύ αποτελεσματικό. Έχουμε βέβαια προς σύμφωνα με την οποία περισσότεροι δημοσιογράφοι στην Αγγλία δεν θεωρούμε ότι συμβαίνει τόσο πολύ στην προστασία τη ελευθερία του λόγου. Σα πάρα πολύ, κύριε. Είστε ένα εκ των διευθυντών τη ε, Guardian. Σα ευχαριστούμε, μα διαφωτίσατε πάρα πολύ. Πάρα πολύ χρήσιμο αυτό για το έργο που έχουμε περίσουμε στο μέλλον. Ε, Σα ευχόμαστε καλή συνέχεια και γυρνάμε ή στο πάνελ μας. Thank you. Opening time for the answers, we thank you for your patience and cooperation for this video conference. Now we're turning back to you. Λοιπόν, επανερχόμεθα στο πάνελ. Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία σας και για αυτή την τηλεδιάσκεψη. Ο κύριος Φολγού να απαντήσει λοιπόν σε ερωτήσεις που έγιναν. Ίσως θα έπρεπε να ξεκινήσω από τις ερωτήσεις που προσπαθούν να δώσουν μια προοπτική σε όλο αυτό το θέμα. Ε, Θα επικεντρωθώ στη γαλλική περίπτωση, αλλά νομίζω οι αντίστοιχε είναι οι πραγματικότητε και οι προβληματικέ σε άλλε χώρε. Αυτή η επανάσταση τη τεχνολογία προφορίας άρχισε πριν την 11η Σεπτεμβρίου από το διαδίκτυο και την εμφάνισή του και κυρίως ένα άλλο στοιχείο το οποίο δεν αναφέρεται αρκετά συχνά δημοσίως, που είναι ότι πέρασε η κρυπτογράφηση στο δημόσιο χώρο. Ε, και αυτό πραγματικά έκανε τις μυστικές υπηρεσίες να φρίξουν. Και μάλιστα στη Γαλλία ε, ε, κάποιοι πράκτορες το έλεγαν έτσι μηδιώντες ότι τώρα που άνοιξε η κρυπτογράφηση και είναι ε, στη διάθεση όλων θα μας βγάλουν όλους στην ανεργία μας των μυστικών υπηρεσιών. Το έλεγαν έτσι χαμογελώντας αλλά μεταξύ αστείου και σοβαρού το εννοούσαν. Δηλαδή τους εξέφυγε από τα χέρια αυτή η δουλειά. Υπήρχε πολύ μεγάλη δουλειά, πολύ λόμπι ε, στους βουλευτές και στις δημόσιες υπηρεσίες για να καθυστερήσει όσο γίνεται ε, η διάθεση στο κοινό αυτών των δυνατοτήτων κρυπτογράφησης και της τεχνολογίας. Στη Γαλλία τώρα, ε, οι υπηρεσίες πληροφοριών Έχω την αίσθηση ότι ακριβώς λόγω αυτής της τεχνολογικής επανάστασης και της διάστασης που πήρε, έτσι και της ε, μαζικής παρακολούθησης και φακελώματος, είναι ένα στοιχείο κυριαρχίας και οι μυστικές ε, υπηρεσίες και οι πληροφορίε. Ε, αυτό που ενδιέφερε τους Γάλλους είναι να είναι αυτόνομοι, να έχουν τη δυνατότητα μόνοι τους να τα κάνουν όλα αυτά. Ε, οι πολιτικοί, ας πούμε, να ε, έχουν μία ίδια γνώμη και να μην εξαρτώνται από πληροφορίες που τους δίνουν κάποιοι σύμμαχοι ή φίλοι ως κράτη. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν με αυτά τα μεταστοιχεία και ποιοι φύγονται, ποιοι είναι οι στόχοι ας πούμε ή τα θύματα πώς να το πω, είναι οι πάντες. Δηλαδή αυτά τα λεγόμενα στοιχεία, τι είναι. Το είπε και ο Λαν Ρασπρίτσερ, ποια είναι αυτά τα στοιχεία. Ε, Ορισμένοι προσπαθούν να ελεγχιστοποιήσουν, αλλά σήμερα για τις μυστικές υπηρεσίες η πληροφορία η πιο σημαντική δεν είναι να ακούνε τα τηλεφωνήματα, να υποκλέπτουν τις τηλεφωνικές συνομιλίες, γιατί ο κόσμος τώρα δεν λέει τίποτα στο τηλέφωνο σοβαρό. Ε, αλλά με αυτά τα μεταστοιχεία μπορεί με λεπτομέρειες ε, κάποιος ε, να δει όλη τη ζωή ε, ενός ανθρώπου, ε, με ποιον επικοινωνεί, πώς μετακινείται, πού πηγαίνει, με ποια συχνότητα κτλ. Δηλαδή πλήρης παρακολουθία παρακολούθηση και πλήρης γνώση για τη ζωή του. Λοιπόν, όταν ε, ζητούν τεχνικές ε, πληροφορίες και βοήθεια, τι γίνεται. Έχει το όνομα κάποιου ή ε, μια ομάδα ή μια εταιρεία ή μια διεύθυνση. Η DGS βάζει μπρο το σούπερ κοριό, το σούπερ υπολογιστή, βγάζει κάποια στοιχεία χίδιν, εκ των υστέρων για μια συγκεκριμένη περίοδο που έχει ζητηθεί και δεν διαβιβάζει ε, στον ενδιαφερόμενο, στην άλλη υπηρεσία ή στην αντικατασκοπία, τη γαλλική στο ε, τελωνίο ή στην αρμόδια αρχή. Δεν διαβιβάζει αυτά τα στοιχεία ε, χωρίς επεξεργασία. Δίνει αυτά τα λεγόμενα μεταστοιχεία, τα οποία είναι επεξεργασμένα με υπεραξία και επανέρχονται αυτά ε, στα χέρια των γαλλικών υπηρεσιών που είναι άλλες απομυστικές ε, ενδεχομένω και υπόκεινται στη γαλλική νομοθεσία. Οι στόχοι ποιοι είναι. Οι πάντες μπορεί να είναι. Μπορεί με να είναι και τρομοκράτες ή άτομα που συνδέονται με την τρομοκρατία, αλλά στα πλαίσια του δικού μας ρεπορτάζ και της έρευνας ακούσαμε ότι ερευνούν και άλλους, όπως αυτές οι μυστικές υπηρεσίες η Γενική Διεύθυνση ε, ε, Πληροφοριών του εσωτερικού της χώρας για κάποιους ας πούμε που ήταν απειλή για τον πρόεδρο της χώρας. Ναι, ενδεχόμενη απειλή, μπορεί να είναι οποιοδήποτε. Ε. Ένας δικηγόρος μπορεί να είναι, ας πούμε, ένας δημοσιογράφος, ένας πολιτικός, ένας ερετός, ένας ευρωβουλευτής. Ε, αν θεωρούν ότι είναι απειλή ε, για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και την ασφάλειά του και την εθνική ασφάλεια γενικά, η δικαιολόγια θα βρεθεί, εν πάση περιπτώσει. Και είναι πολύ γενικόλογοι συνήθως και αόριστη, και ε, θα γίνει το αίτημα και θα δοθούν τα στοιχεία χωρίς να υπάρξει κανένας έλεγχος και χωρίς να εμποδίσει κανείς τίποτα. Έγινε μια ερώτηση σχετικά με την νομιμότητα, πώς νομιμοποιείται ε, η ηγεσία αυτών των υπηρεσιών. Το είπα και προηγουμένως σε συντομία. Οι άνθρωποι αυτοί λένε ότι είναι του κράτους, έμπιστοι, ότι είναι καλοί πατριώτες. Εγνωρίζουν και αυτοί ε, σε ποια θολή κατάσταση κινούνται και σε ποια παρανομία. Δεν είναι παράνομο, είναι άνομο όπως είπε ένας ε, διευθυντής ε, που χρησιμοποιεί τα στοιχεία της ΔΕΖΕΣΕ και κάποια άλλα εκτός νόμου. Οι άνθρωποι αυτοί λένε ότι κάποια στιγμή θα βρεθούμε μοιραία μπροστά σε ένα δικαστή. Ορισμένοι φοβούνται, άλλοι καθόλου από το γεγονός αυτό. Αλλά πώς να το πω, το επάγγελμά τους το ίδιο και η δουλειά τους έχει να κάνει με αυτό, έτσι δουλεύουν. Δεν, δεν ε, σκέφτονται ότι υπάρχουν δικαστές στον κόσμο. Και η εκτελεστική εξουσία εδώ και χρόνια έχει φροντίσει ακριβώς οι δικαστές να μην πλησιάζουν αυτό τον κόσμο, τον εφέλωμα των μυστικών υπηρεσιών. Και υπάρχει και ένα θέμα μαζικής και αδιάκριτης ε, διαβίβασης αυτών των στοιχείων. Ε, υπάρχει και μια λογική αναπόφευκτα εδώ αποτελεσματικότητας. Ξέρετε η Γαλλία ότι θέλει να είναι και αυτή στο ύψος άλλων κρατών στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, να είναι εξίσου ε, αποτελεσματική και ισχυρή με κάποιους γείτονες. Αυτά τα στοιχεία που διαχειρίζονται ορισμένοι εκεί και τα επεξεργάζονται δίδονται και στην αστυνομία ιδιαίτερα στην αντιτρομοκρατική. Ξέρετε ότι έχουμε υπηρεσίες που ασχολούνται με τη διεθνή τρομοκρατία στην αστυνομία και εκτός των γαλλικών συνόρων, βέβαια η βάση του είναι η Γαλλία. Σε αυτή την περίπτωση έχουν και άμεσες σχέσεις και συνδέσμους ε, οι ε, τεχνικές υπηρεσίες των μυστικών υπηρεσιών με τις αστυνομικέ αυτέ υπηρεσίε, για πληροφορίε σε σχέση με κάποιου που μπορούν να ταξιδεύουν, να φεύγουν από τη Γαλλία, να πηγαίνουν σε άλλες χώρες και να επιστρέφουν. Και υπάρχει μια συμμαχία μετά και ένα κράμα με διάφορες τεχνικές και στα πρακτικά της δικαιοσύνης μπορείτε να βρείτε ε, βάσει μια ανώνυμης πληροφορίας ε, συγκεκριμένες εκφράσεις που κρύβουν την προέλευση της πληροφορίας και την πηγή που έρχεται να θρέψει μια δικαστική ε, διαδικασία και μπορεί να συνδέεται με κάποια νομικά προβλήματα. Γιατί όλες αυτές οι πληροφορίες δεν προήλθαν από πηγές τέτοιες αντιπαράστασης, αντιπαράθεσης μαρτύρων κτλ. και με τον τρόπο που είναι σύνομος σε πάση περιπτώσει. Αυτή η λογική της κυριαρχίας και το να είμαστε αυτόνομοι από πλευράς πληροφοριών δεν αποκλείει βέβαια Ανταλλαγέ πληροφοριών και η μαζική αυτή παρακολούθηση που ήρθε να ενισχυθεί από την 11η Σεπτεμβρίου πολλές φορές ε, χρησιμοποιείται ε, πραγματικά ως πολιτική δικαιολογία, όπως είπε προηγουμένως ένας βουλευτής. Έρχονται να τα δικαιολογήσουν όλα αυτά τα τεχνικά. Ε, υπάρχουν ανταλλαγές και στη Γαλλία έγινε μια ακρόαση στη Γερουσία. Ο πρώην ε, διοικητή της ΔΕΖΕΣΟ είχε πει ότι υπάρχει κοινή βάση δεδομένων σε ένα κλειστό κύκλο των βασικών δυτικών μυστικών υπηρεσιών ε, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και όλοι αντλούν από εκεί στοιχεία, όλοι βάζουν στοιχεία. Για παράδειγμα στις Ηνωμένε Πολιτείε. Οι Ηνωμένε Πολιτείε απευθύνονται πολύ συχνά στη Γαλλία που ξέρει πάρα πολύ κατεκάτασταση στο Σαχέλ και πολύ συγκεκριμένα πράγματα ζητούν οι Αμερικανοί. Και η NSA τηλεφωνεί στην DGSE και τους λέει δώστε μας σας παρακαλώ την παραγωγή ενός μηνός υποκλοπών στο Σαχέλ. είναι όχι μόνο τα τεχνικά μηνύματα που περνούν, αλλά και τα ηλεκτρονικά από τη Γαλλία στο Σαχέλ, από το Σαχέλ προς τη Γαλλία. Euh, είναι μια τεράστια βάση δεδομένων που χωρίς κανέναν έλεγχο διαβιβάζεται από τις γαλλικές υπηρεσίες τις αμερικανικές οι οποίες ε, τα επεξεργάζονται με τα δικά τους ε, ε, μέσα και δυνατότητες. Δεν ξέρω αν μου διέφυγε κάτι, αλλά υπάρχει μια μεγάλη διαφορά ανάμεσα ε, στην τακτική του Edward Snowden και εκείνη που υιοθέτησαν ε, στα Wikileaks. Απευθύθηκα στον τύπο, σε εφημερίδες και υπάρχει μια δημοσίευση υπεύθυνη. Δηλαδή, αυτό που ενδιαφέρει εδώ δεν είναι πλήρης διαφάνεια δεν τα ρίχνουν όλα στο φως αδιάκριτα, ε, δεν τα δημοσιοποιούν όλα τα στοιχεία. Αυτή η τακτική προσέγγιση, δεν ξέρω αν είναι πραγματικότητα, αυτό ακούμε, αλλά για μας αυτό νομιμοποιεί τη δράση μας και τις αποκαλύψεις και τη συμμετοχή στη συζήτηση για τις ελευθερίες. Έτσι ο Έντουαρτ Σνόντεν γίνεται πιστευτός, αξιόπιστο. Συχνά υπάρχει το επιχείρημα που λέει πήγε στο Χονγκ Κονγκ και μετά διέφυγε στη Μόσχα. Στο Χονγκ Κονγκ πήγε γιατί μπορούσε να έχει κάποια ελευθερία για να δώσει αυτά τα στοιχεία, να έχει επαφές με τους συνδέσμους εκεί, με τον ε, Green Wall ή τους άλλους, ενώ σε ό,τι αφορά τη Ρωσία δεν την επέλεξε. Η χώρα δέχτηκε να τον ε, υποδεχτεί. Για την ελευθεροτυπία και θα τελειώσουμε αυτό. Είναι προφανές ότι υπάρχει μια ενδεχόμενη απειλή, δεν το αφισβητώ. Αλλά ακριβώς επειδή είναι τέτοια τα προγράμματα παρακολούθησης και φακελώματος και στη Γαλλία και στις Ηνωμένε Πολιτείες, βρισκόμαστε μόνο στην αρχή. Δεν έχουμε, τώρα αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε το σύστημα, πόσο διεισδυτικό είναι και πόσο ευρεία είναι η παρακολούθηση και διαδεδομένη. Βέβαια, οι βασικές χώρες αυτές δεν περιορίστηκαν να χρησιμοποιούν αυτό το ηλεκτρονικό εργαλείο μόνο για την τρομοκρατία. Το χρησιμοποίησαν και για άλλους πολέμους, οικονομικούς, πολιτικούς και πάει λέγοντας όλους τους πολέμους. Τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια θα δούμε ε, τι θα προκύψει, γιατί οι εφημερίδες θα συνεχίσουν να κάνουν τη δουλειά τους και θα δούμε και τις ε, κυβερνήσεις και τις χώρες να εκτίθενται. Έλεγα λοιπόν ότι θα ασκηθούν όλο και μεγαλύτερες πιέσεις στους δημοσιογράφους με εκφοβισμό ε, και με απειλές και με διώξεις, αλλά αυτό θα είναι όντως οδυνηρό για τους δημοσιογράφους τα επόμενα έτη. Σας ευχαριστούμε κύριε Φολογού. And now again, again, as... Και τώρα, way behind επειδή έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ, θα ήθελα να προτείνω να χειριστούμε λίγο διαφορετικά την ημερήσια διάταξη. Mm. Ως εξής, Υποτίθεται ότι πρέπει να φτάσουμε στο δεύτερο τμήμα που είναι η παρακολούθηση της ε, μόνιμης επιτροπής ε, για το σύστημα ε, παρακολουθήσεων του ΕΣΕΛΟΝ και εδώ έχουμε τρεις ομιλητές, τον Κάρλος Κοέγιο, τον κύριο Ντάνκιαν Κάμπελ ο οποίος και αυτός κάνει ερευνητική δημοσιογραφία και τον πρώην συνάδελφο, τον κύριο Γκέρχαρ Σμίτζ, πρώην Ευρωβουλευτή, ο οποίος ήταν εισηγητής για την έκθεση ΕΣΕΛΟΝ του 2001. Και επειδή πρέπει στις 5.30 να φύγει. Ε, ευχαριστούμε καταρχάς τον κύριο Applebaum που ε, δέχτηκε να παραχωρήσει τη θέση του. Να δώσουμε το λόγο στον πρώην συνάδελφο, τον κύριο Γέρχαρτ Σμιθ και μετά θα ακούσουμε τις απαντήσεις ε, του κυρίου Applebaum για να μπορέσει να συνεχίσει το πρόγραμμά του απρόσκοπτα. Κύριε Σμιθ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Συμφώνησα με τον συνάδελφο Κοέγιο να μιλήσει εκείνος για τα αποτελέσματα της έρευνας για το ΕΣΕΛΟΝ και εγώ ουσιαστικά θα περιοριστώ σε κάποιες σκέψεις που έχουν να κάνουν με την εμπειρία που είχαμε από την έρευνα αυτή. Εάν έχετε ερωτήσει, είπε ο κύριος Κοαΐ ότι θα απαντήσει και εκ μέρου μου, γιατί ξέρει με βάση την έρευνα όλες τις λεπτομέρειες. Τα διαδικαστικά. Σε αντίθεση με το έσελον, για το πρίσμ ή το τέμπορα δεν χρειάστηκε να γίνει έργο detective για να το αποδείξουμε. Υπάρχουν τα έγγραφα. Αυτό είναι σημαντική διαφορά σε σχέση με το έσελον. Αλλά παρόλα αυτά ε, θα πρέπει να διερευνηθεί πραγματικά αυτό. Αν δούμε τα έγγραφα που δημοσίευσε ο Σνόουντεν, χρειάζεται μεγάλη μελέτη για να καταλάβουμε τι εννοεί πολλές φορές και οι ορισμοί δεν είναι κοινοί, δεν είναι κοινό αγαθό ας πούμε, δεν καταλαβαίνει ο καθένας τι σημαίνει. Και θα παρακαλούσα ε, να ε, μπορέσουμε για να ε, καταλάβουμε απολύτως τι μπορούν να κάνουν αυτά τα συστήματα, μόνο αν τα καταλάβουμε θα βγάλουμε πολιτικά συμπεράσματα. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε τι ακριβώς κάνουν αυτά τα συστήματα και τι είναι σε θέση να κάνουν από την αρχή. Ένα δεύτερο, από την εμπειρία μου και πάλι, είναι πολύ αποφασιστικό για την αξία αυτής της έκθεσης, η σοβαρότητα με την οποία θα πρέπει να εργαστείτε. Γι' αυτό θα σας συνιστούσα να μην υιοθετείτε όλα τα στοιχεία που σας δίνουν αγόγγιστα και ανεξέλεγκτα, αλλά να ελέγχετε πάντα τις ε, πηγές ως προς τη σοβαρότητα. Γιατί έτσι γίνεται σε κάθε επιστημονική εργασία. Αυτό θα αυξήσει σημαντικά αργότερα την αξία της μελέτης σας και της έκθεσής σας. Ένα άλλο τεχνικό επίσης για την εργασία και μεθοδολογικό. Έχετε χρόνο μέχρι το Δεκέμβριο και καλό θα ήταν να ε, περιοριστείτε σε επίπεδο συντονιστών επί της ουσίας τι θέλετε ακριβώς να κάνετε κατά τη διάρκεια των εργασιών σας να μην χάσετε χρόνο γιατί είναι αντιπαραγωγικό. Και επίσης ε, θα πρέπει να αξιοποιήσετε τις επιστημονικές υπηρεσίες άλλων κοινοβουλίων όπως είναι το Αμερικανικό Κογκρέσο ή της Βουλής των Κοινοτήτων. Έχουν καταπληκτικό υλικό ήδη και μπορούν να σας βοηθήσουν. Υπάρχει αυτό το υλικό, δεν χρειάζεται να το ψάξετε από την αρχή. Στη συνέχεια, τι θα πρέπει τώρα να διερευνηθεί. Το ΕΣΕΛΟΝ, τι έδειξε, ότι μια υπηρεσία πληροφοριών παρακολουθούσε τις επικοινωνίες και έκανε τα πάντα και μπορεί πραγματικά να κάνει τα πάντα. Ό,τι υπάρχει τεχνικά και ε, ό,τι μπορεί να πληρωθεί, ό,τι είναι προς το συμφέρον της χώρας, το κάνουν. Και επίσης ό,τι τους επιτρέπει ο νόμος. Δεν ξέρουμε εάν οι υπηρεσίες κάνουν και πράγματα που τους απαγορεύει ο νόμος. Αλλά μπορεί κανείς να δει από τις λεπτομέρειες το τι επιτρέπεται για τις υπηρεσίες πληροφοριών θα καταλάβετε τουλάχιστον τι κάνουν, γιατί ό,τι επιτρέπεται το κάνουν. Και αυτό μπορεί να είναι για σας πολύ χρήσιμο. Επίσης θα πρέπει να αφιερώσετε χρόνο στο να καταλάβετε τεχνικά πώς γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Πώς παρακολουθούνται οι τηλεπικοινωνίες, πώς γίνονται οι υποκλοπές, για να το καταλάβετε ποια είναι τα μηχανήματα. Γιατί δεν είναι τίποτα ε, ερασιτέχνες ε, των μυστικών υπηρεσιών μαστροχαλαστής ας πούμε που παίρνει ένα ραδιόφωνο και φτιάχνει ένα πομπό. Είναι εταιρείε που είναι δουλειά τους και βγάζουν λεφτά γιατί τους τα πουλάνε αυτά τα μηχανήματα. Και υπάρχουν και εταιρείε επίσης που επεξεργάζονται δεδομένα. Καλέστε μια τέτοια εταιρεία για να δείτε ακριβώς πού δραστηριοποιούνται και τι δυνατότητες υπάρχουν τεχνικές. Ένας άλλος τομέας και ένα πρόβλημα που δεν υπήρχε επί έσελον, υπάρχει τώρα, είναι το εξής γεγονός. Η Υπηρεσία Εθνικής Ασφαλείας, η NSA, έχει αναθέσει 70% των εργασιών ε, και του προπολογισμού σε εξωτερική ανάθεση, σε υπεργολαβίες. Αυτό έχει να κάνει με την ασφάλεια. Το είδαμε και με τον Σνόουντεν. Πόσο μεγάλη είναι η ασφάλεια της ίδιας της υπηρεσίας εθνικής ασφάλειας. Η NSA δεν έχει στην κυριότητά της ούτε τα ίδια τα τηλέφωνα τα οποία χρησιμοποιεί. Δηλαδή οι άνθρωποι παρακολουθούν τα τηλέφωνα και τα ίδια τους τα τηλέφωνα ανήκουν σε ιδιωτικές εταιρείε. Καταλαβαίνετε αυτό τι σημαίνει και θα πρέπει να σας απασχολήσει στη διάρκεια των ερευνών σας. Ποιος μπορεί να σας βοηθήσει σε αυτή την προσπάθεια, πάντα σύμφωνα με τις δικές μας εμπειρίες. Οι κυβερνήσεις και οι δικές μας κυβερνήσεις δεν έχουν κανένα συμφέρον να σας βοηθήσουν και επί τα ίδια είδαμε. Αντίθετα, πολλές φορές μπορεί να σας λένε και ψέματα οι κυβερνήσεις. Εμάς μας φλόμωσαν στο ψέμα. Και η Αμερικανική κυβέρνηση και η Βρετανική μας έλεγαν ότι δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα έσελων, δεν έχουμε τέτοιες ε, συμφωνίες. Έκτοτε ε, δεν είναι πλέον απόρριτα, έχουν δημοσιευτεί αυτά τα έγγραφα ε, και έχουν αποχαρακτηριστεί και φυσικά υπήρχαν. Αν απευθυνθείτε σε εθνικά κοινοβούλια είτε δεν επιτρέπετε να σας πούνε τίποτα, είτε αποδυναμώνονται και, και έχουν αδυναμίες και δεν θέλουν να τις ομολογήσουν και να ξεμπροστιαστούν και δεν θα σας βοηθήσει κανείς εάν καλέσετε κάποιον από την Ευρωπαϊκή... Μάλλον δεν θέλουν τα Εθνικά Κοινοβούλια να ανακατεύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση στις ειδικέ σας ε, υποθέσεις. Άρα, ποιος θα σας βοηθήσει. Η ερευνητική δημοσιογραφία μπορεί να βοηθήσει και ό,τι σας δίνουν οι δημοσιογράφοι όμως να το μελετάτε πάρα πολύ προσεκτικά. Πάρα πολύ προσεκτικά σημαίνει ότι θα πρέπει να δείτε κατά πόσο οι πηγές είναι αξιόπιστες, γιατί υπάρχει μαχόμενη και ερευνητική δημοσιογραφία, αλλά είναι δύο είδους δημοσιογράφοι. Είναι η ερευνητική και κάποιοι άλλοι είναι οι δημιουργικοί δημοσιογράφοι. Παρακαλώ, ε, μην πιστέψετε αυτούς που θέλουν να σας πουλήσουν μια ιστορία. Θα πρέπει πάντα να ψάχνετε την ιστορία. Δεν κατηγορώ κανέναν, απλώς μην πιστεύετε ότι σας λένε, όπως και οι κυβερνήσεις και οι δημοσιογράφοι δεν είναι όλοι καθώ περιστερές. Πρέπει να τα κοιτάτε μόνοι σας αυτά και να τα ελέγχετε. Επόμενο θέμα, η ασφάλεια στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, γιατί και αυτό ανέκυψε. Ακούνε την, αντιπροσωπεία μας στην Ουάσιγκτον και τις Βρυξέλλες επίσης, κοριούς και κυβερνήσεις. Κοιτάξτε, κυβερνήσεις και τα κράτη δεν έχουν φίλους, τα κράτη έχουν συμφέροντα. Μπορεί να έχουν συμμάχους για τα συμφέροντά τους ενίοτε, το πολύ πολύ, αλλά δεν έχουν φίλους ποτέ. Για μας είναι σημαντικό το εξή. Και από τότε το είχαμε επικρίνει επί έσελον, ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουμε σύστημα προστασίας από κατασκοπία. Δεν έχουμε αυτό που έχουν οι μεγάλες εταιρείες, ασφάλεια των εταιριών. Ούτε καν. Και αυτό θα πρέπει να το συζητήσουμε. Δεν μιλώ για το Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο έτσι κι αλλιώς είναι όλα δημόσια. Αλλά μιλώ για Κομισιόν και Συμβούλιο. Δεν μπορώ να το δεχτώ εγώ αυτό. Η εκπρόσωπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στην Ουάσιγκτον να μην έχει μέχρι σήμερα αίθουσα, γραφείο που να είναι ασφαλές από παρακολουθήσεις. Και οι φίλοι μεταξύ τους κατασκοπεύονται. Η κάθε πρεσβεία έχει τέτοια ασφαλή δωμάτια. Εμείς δεν έχουμε. Επίσης, θα πρέπει να ελέγξετε τις δυνατότητες, τις νομικές, αν όλα αυτά που κάνετε συνάδουν με το ε, κοινοτικό δίκαιο ή με το εθνικό δίκαιο ή πώς μπορεί κανείς να προστατεύσει τις εθνικές επικοινωνίες. Τι εννοώ. Στο παρελθόν όταν τηλεφωνούσα ή έστειλε ένα email από μία χώρα σε μια άλλη χώρα, ε, πήγαινε ε, από το πιο σύντομο δρόμο. Σήμερα δεν ξέρουμε που πάει το email. Μπορεί να πάει μέσω Αμερικής, μέσω Κίνας ή μέσω Κολοπετινίτσας. Ε, ανάλογα με το ποιο είναι πιο φτηνό. Αλλά θα πρέπει να δούμε, ε, δεν μιλάω για το Facebook, δεν μιλάω για διεθνείς επικοινωνίες, αλλά μέσα στην ίδια χώρα θα πρέπει να ελέγχεται αυτό. Ορισμένοι όταν κάποιος έχει ε, ε, και πληρώνει ένα ποσό κατά αποκοπή, ένα flat rate, θεωρεί ότι δεν παρακολουθείτε. Νομίζετε ότι δεν παρακολουθείστε σήμερα, ε, μπορεί να παρακολουθείτε και αυτό και οι αμερικανικές εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν και βάσει του αμερικανικού δικαίου μπορούν να φτάσουν σε αυτά τα μεταστοιχεία και, ε, ε, στην τιμολόγηση υπάρχει η δυνατότητα ε, να έχει ο πάροχος κάποια στοιχεία να τα διατηρεί, να τα αποθηκεύει, αλλά να μην τα εξάγει. Αυτά σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και να με συμπαθάτε γιατί πρέπει να φύγω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε αγαπητοί συνάδελφοι Χερ Σμιτ. Okay. Yes. Now. Και τώρα. να περάσουμε στο πρώτο τμήμα της ε, συνεδρίασής μας να δώσουμε και πάλι το λόγο στον κύριο Applebaum για να μας απαντήσει τις ερωτήσεις ε, που του απευθύνθηκαν και μετά θα περάσουμε και πάλι στο δεύτερο τμήμα της συνεδρίασης με τους συναδέλφους, τον κύριο Κοέγιο και τον ε, προσκεκλημένο μας, τον κύριο Κάμπελ. Κύριε Applebaum, έχετε το λόγο. Ο Ντάνκαν Κάμπελ συμμετείχε στην περίπτωση της Έσελον και ήταν πολύ σημαντικά διότι με βοήθησε να μάθει για την κρυπτογραφία και για το τι γίνεται με την παρακολούθηση ε, και μάλιστα σε μια εποχή που οι νομοθέτες ενδιαφέρονταν για την παρακολούθηση και δεν θεωρούσαν ότι έπρεπε να είναι όλα μυστικά. Ένα-δύο πράγματα λοιπόν τα οποία θα ήθελα να θίξω. Καταρχάς να πω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός των ερωτήσεων που μου θέσατε. Θα προσπαθήσω να απαντήσω όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Καταρχάς να πω ότι το θέμα αυτό είναι ιδιαίτερα πυκνό και εμείς στις Ηνωμένε Πολιτείε έχουμε ε, τη λεγόμενη Church Committee. Χρειαζόμαστε μια τέτοια στις ε, Ηνωμένε Πολιτείε, διότι χρειαζόμαστε να έχουμε τη δυνατότητα να στείλουμε ε, ένταλμα, κλίση σε κάποιον να έρθει να μιλήσει και να μιλήσουμε με τους υπευθύνου και να ρωτήσουμε ποιοι είναι οι υπεύθυνοι και θα ήθελα να βοηθήσω ή τον εαυτό μου ή τον Ντάνκαλ Κάμπελ να πάρουμε τους φακέλους μας από όλες τις μυστικές υπηρεσίες παγκοσμίω για να δείτε έτσι τι δυνατότητες έχουν αυτά τα συστήματα. Νομίζω ότι εμείς οι δύο έχουμε φακέλους τους οποίους θα αξίζει τον κόπο να διαβάσετε. Και μπορώ να σας πω βάλτε τους και αναρτήστε τους κάλλιστα στο διαδίκτυο. Αναφερθήκατε στο σκοπό, κύριε Μωράς. Ο σκοπός είναι αυτός ο οποίος δηλώσαμε. Ο ρόλος μιας υπηρεσίας πληροφοριών είναι να βοηθά τον έλεγχο και να επιβραδύνει κάποια πράγματα, όπως είπε και ο Άλλεν, διότι αυτό είναι ένας από τους θεμελιώδους τρόπους με τον οποίο μπορούμε να βοηθήσουμε και τους πολιτικούς, αλλά μπορεί να βοηθήσει και πολλές άλλες ομάδες να έχουν μια κάποια μορφή έλεγχο. Να σταματήσει η διάδοση, να καθυστερήσει η διάδοση των πληροφοριών για να μπορέσουμε να ελέγξουμε τι συμβαίνει, να μπορέσουμε να ε, καταστρέψουμε στοιχεία, να αλλάξουμε πληροφορίες, να δούμε αν κάποιος εκ των έσω προσπαθεί να διαρρεύσει κάποιου, να τους περάσουμε από έναν ανοιχνευτή ψεύδους, να δούμε τι γίνεται. Αυτός είναι ο στόχος των ε, συστημάτων παρακολούθησης ο έλεγχος. Και γι' αυτό ακριβώς χρησιμοποιούνται αυτά τα συστήματα. Η παρακολούθηση λοιπόν δεν είναι ο στόχος προς τον ολοκληρωτισμό, είναι ο ολοκληρωτισμός αυτός καθεαυτός, περιορισμένος σε μια στιγμή. Αλλά όταν η Χρυσή Αυγή στην Ελλάδα έχει πρόσβαση σε μυστικές πληροφορίες και έχει τη συγκεκριμένη ιδεολογία που έχει, τι θα γίνει. Θα είναι τελείως διαφορετικά χωρίς το σύστημα παρακολούθησης και το έχουμε δει αυτό ε, στην Ευρώπη με τα συστήματα της κάρτας ε, που χτυπάει ο καθένας ε, το πρωί στη δουλειά τους. Έχουμε δει τι συμβαίνει και στην Γαλλία και αλλού. Θα ήταν χρήσιμο λοιπόν ε, και να δούμε και πώς το χρησιμοποιεί ο καθένας. Το πώς το χρησιμοποιούν οι Ηνωμένε Πολιτείες είναι διαφορετικό από τον τρόπο που χρησιμοποιούνται στη Γερμανία και στη Γαλλία. Ξέρουμε στις Ηνωμένε Πολιτείες γίνεται ε, για ε, παράνομα στοιχεία, για δολοφονίες κατά ανθρώπων και από εκεί και πέρα υπάρχει και κάτι ακόμα. σε πολλές πολιτείες στι Ηνωμένε Πολιτείες ισχύει θανατική ποινή που από, κατά μια μορφή είναι και αυτή μια μορφή λογοκρισίας. Και εγώ θα ήθελα να ξέρω κάποια πράγματα για το πού χρησιμοποιούνται αυτά τα στοιχεία. Από ό,τι γνωρίζω υπάρχει σίγουρα οικονομική κατασκοπία και ε, οι Ηνωμένε Πολιτείε λένε ότι σταματούν την οικονομική κατασκευή με τη χρήση αυτού του προγράμματο. Ε, είναι συναρπαστικό αυτό το στοιχείο, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Εγώ νομίζω ότι είναι κατάφορο ψεύδος. Ε, νομίζω ότι η δημοκρατική διαδικασία μπορεί να λειτουργεί καλά για εσά, αλλά δεν λειτουργεί για εμά, αλλά σας βοηθούμε. Σίγουρα χρησιμοποιείται για πολέμους, από προσωπική και επαγγελματική πείρα με συναδέλφου, ε, γνωρίζω ότι χρησιμοποιείται και για πολιτικές διώξει, και αυτό είναι σαφές. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν για να εξεύρουμε τη δέουσα ισορροπία. Νομίζω ότι αυτό το οποίο θα πρέπει να κατανοήσουμε εδώ είναι ότι υπάρχουν κατάσκοποι οι οποίοι σε γενικέ γραμμέ είναι εγκληματίε και λένε ότι πρέπει να του χρησιμοποιούμε ε, στην πρώτη γραμμή τη ασφάλειά μα. Και τι κάνουμε. Είμαστε έρμεο τη ανασφάλεια. και πιστεύουμε ότι θα μας ε, προστατεύσουν. Και στη Γερμανία τι λέει η κυβέρνηση. Λέει ότι οι Γερμανοί πολίτες, οι Γερμανείς επιχειρήσεις έχουν ευθύνη οι ίδιοι να προστατεύσουν τους εαυτούς τους. Και νομίζω ότι αυτή δεν είναι η κατάλληλη ισορροπία. Εάν ε, δεν υπάρχει ασφάλεια, οτιδήποτε χρησιμοποιεί, χρησιμοποιείται εξορισμού δεν έχει ασφάλεια, τότε έχουμε πρόβλημα. Ε, όταν κάποιον μας λέει ότι μας εξασφαλίζει, θα πρέπει να νιώθουμε ασφάλεια. Αυτή είναι εξορισμού η έννοια της ισορροπίας. Ο κύριος Άλμπρεχτ αναφέρθηκε στη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών και νομίζω ότι αυτό είναι και προφανέ από αυτά τα οποία δηλώνονται και δημοσίω και από τα έγγραφα τα οποία διέρευσαν και από τι συζητήσει που έχουν γίνει και με το Σνόντεν και με άλλου δημοσιογράφου που ε, ασχολούνται με τα θέματα αυτά. Στον 20ο αιώνα θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι υπηρεσίε πληροφοριών εργάζονταν για τη χώρα του ε, κατά των υπολείπων κρατών και υπήρχαν και κάποιε σημασίε. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι όλε οι υπηρεσίε πληροφοριών συνεργάζονται συνεργάζονται μεταξύ τους εναντίον ημών. Και νομίζω ότι αυτό μας τρομάζει τουλάχιστον. Το 70% μιλούσα με τη Ρόλα Ωρα ε, Πόλτρες ε, πριν από λίγες μέρες ε, και αυτή μου έλεγε ότι το 70% των στοιχείων που λαμβάνονται προκύπτουν από συνεργασία και με επιχειρήσεις. Άρα μπορούμε να εξασφαλίσουμε το 70% των τηλεπικοινωνιών μας εάν δώσουμε κατάλληλα κίνητρα για να υπάρχει προστασία στον τρόπο με τον οποίο ερχόμαστε σε επαφή με επιχειρήσεις και δίνουμε στοιχεία για τους εαυτούς μας. Διότι το θέμα δεν είναι αν η Αμερικανική κυβέρνηση ή μια Ευρωπαϊκή κυβέρνηση έχει πρόσβαση στα στοιχεία, αλλά τι θα γίνει αν μια Κινέζικη ε, κυβέρνηση ε, μπορέσει να παρισφρήσει στα στοιχεία. Ε, κατάφεραν, για παράδειγμα, να παρισφρήσουν στο σύστημα της Google και να δούνε κάποιους στόχους της Google. Επομένως δεν είναι θέμα του κατά πόσο εμπιστευόμαστε ή όχι την Google, αλλά το να αναγνωρίσουμε ότι δεν έχουμε δικαίωμα επιλογής, κάποιος άλλος επιλέγει αντί ημών. Και επομένως τι θα πρέπει να κάνουμε. Θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να ε, ασφαλίσουμε αυτούς. Εγώ έχω εδώ ένα τηλέφωνο κρυπτογραφικό, το οποίο μου λέει ότι υπάρχουν και δυνατότητες να ε, κάνει κάποιες παρεμβολές και να ε, ε, πάρει στοιχεία από το τηλέφωνό μου εδώ στο κτίριο. Μπορεί να είναι και κάποιος ε, μικροϊός, αλλά εγώ νομίζω ότι δεν είναι. Θα μπορέσει λοιπόν κάποιος ε, να, να υποκλέψει κάποια στοιχεία. Εγώ έχω cryptophone, redphone, tech διάφορα στοιχεία λογισμικού που κρυπτογραφούν στοιχεία και μέσω της έρευνας για να μπορέσω να έχω αποκεντρωμένα ασφαλή συστήματα, για να μπορούμε να είναι απόλυτα ασφαλή, χωρίς να υπάρχουν ε, δυνατότητες να μπει κάποιος από το παράθυρο, ε, θα μπορέσουμε να έχουμε ε, την πλήρη δημοκρατία, την ελευθερία του λόγου και νομίζω ότι αυτό μπορούμε να το επιτύχουμε. Δεν είναι μια ουτοπία, ε, υπάρχει μέσα σε αυτό το τηλέφωνο και εσείς δεν το έχετε. Γιατί να το έχω εγώ και να μην το έχετε κι εσείς. Η απάντηση είναι ότι ναι, θα πρέπει να το έχετε κι εσείς, οι περισσότεροι δεν το έχετε και χωρίς καμία αμφιβολία τους περισσότερους από εσά τους παρακολουθούν και νομίζω ότι η συγκεκριμένη συσκευή είναι πρωτότυπη μεν, αλλά αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι οποιοδήποτε ανά τον κόσμο, αν σηκώνει το τηλέφωνό του να τηλεφωνήσει, θα πρέπει να έχει αυτή τη δυνατότητα. Και γιατί δεν συμβαίνει αυτό, γιατί υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι υποτίθεται μας κρατούν ασφαλείς και τι κάνουν, στην πραγματικότητα ε, είναι αυτοί οι οποίοι μας παρακολουθούν. Στην, ε, στο GSM δημιουργήθηκε ένα τελείως διαφορετικό σύστημα για τις εξαγωγές, για να μπορούν οι υπηρεσίες πληροφοριών να παρακολουθούν κάποιες ε, ε, αποστολές. Και το σύστημα της Washington είναι ένα σύστημα το οποίο στήχησε 52,6 δισεκατομμύρια ε, δολάρια ετησίως. Ε, μετά από την 11η Σεπτεμβρίου νομίζω ότι ετησίως κάπου τόσα δαπανώνται. Δεν ξέρω αν γίνονται όλα αυτά τα οποία ε, ε, περιλαμβάνονται τα πάντα. Παραδείγματος χάρη όλες αυτές οι πτήσεις ε, της CIA ε, για τις επιστροφές δεν νομίζω ότι περιλαμβάνονταν εδώ. Δεν μπορώ να απαντήσω βέβαια όλες τις ερωτήσεις που ετέθησαν. Για παράδειγμα υπάρχει μια ερώτηση για το Five Eyes, αν οι χώρες αυτές, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Νέα Ζηλανδία, ο Καναδάς, οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεργάζονται και ανταλλάζουν εθνική νομοθεσία. Εδώ η απάντηση είναι σαφής. Ναι, υπάρχει και ε, ένα κτίριο στη Washington όπου ε, είναι κοινό για κάποιες υπηρεσίες πληροφοριών. Δεν το έχω δω ή έχω κάποιες δορυφορικές φωτογραφίες όπου γίνεται αναμετάδοση των στοιχείων μεταξύ των δύο πλευρών ώστε ο ένας να παρακολουθεί από τη μία πλευρά και ο άλλος να υποκλέπτει από την άλλη. Και ε, δεν χρειάζεται να πω εγώ τίποτα άλλο, θα τα πει ο Ντάνκαν Τώρα, αν η NSA έχει υποκλέψει ευρωπαϊκούς ε, υπολογιστές, η απάντηση εδώ είναι ναι, αδιαμφισβήτητα. Όσον αφορά τους ε, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, νομίζω αντίστοιχη ερώτηση μπορείτε να θέσετε και για πυρηνικά εργοστάσια, νοσοκόμια, ε, ευρωβουλευτέ. Ναι, η απάντηση είναι όλους τους παρακολουθούμε. Και πραγματικά εγώ θα ανησυχούσα διότι ε, υπάρχουν προβλήματα. Τι γίνεται αν γίνει κάτι κατά λάθο ένα σύστημα ελόγχου και το σύστημα καταρρεύσει. Ποιο είναι υπεύθυνο, αυτό θεωρείται πολεμική δράση, ε, υπάρχει οικονομική ευθύνη γι' αυτό. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολύ σοβαρέ συνέπειες αν ε, ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση. Και υπάρχει και όλη αυτή η συζήτηση για του hackers, ε, και αν οι Κινέζοι για παράδειγμα είναι τόσο κακοί άνθρωποι γιατί ε, έκαναν υποκλοπή σε τόσες πληροφορίες τι θα γίνει με την NSA που παρακολουθεί όλο τον κόσμο και τίποτα δεν συμβαίνει ε, τίποτα γι' αυτό είναι πολύ πιο ανησυχητικά τα πράγματα και υπάρχει και μεγάλο ψυχολογικό κόστος εγώ τα τελευταία τέσσερα χρόνια για τη συμμετοχή μου με τα Wikileaks υπήρξα στόχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ε, μου έχουν στείλει διάφορα διοικητικά εντέλματα, κατασχέσεις, δημεύσεις, ε, κάποια πράγματα τα οποία ίσως δεν επιτρέπεται να σας πω, κάποιες νομικές δυνατότητες που αν ε, ε και αν υπήρχαν δεν θα μπορούσα να σας πω. Κάποιος ε, ε, μου είπε ότι ακόμα και αν μάθαινα ότι υπάρχει μια επιστολή εθνικής ασφαλείας σημαίνει ότι έχει διαρρεύσει επιστολή. Και πραγματικά χρησιμοποιείται ορολογία τρομοκρατίας για τα Wikileaks, το οποίο είναι μια ανοησία. Τα Wikileaks δεν είναι τρομοκρατία, είναι δημοσιογραφία. Και όπως είπε και ο Γάλλος δημοσιογράφος, η Guardian ήταν αυτή η οποία έδωσε στοιχεία. Η Wikileaks έκανε ε, μεγάλη προσπάθεια να μην δώσει ονόματα, ε, έχει αφαιρέσει ονόματα από στοιχεία και προσπαθούν να είναι ιδιαίτερα προσεπτικοί και να μην δίνουν ονόματα για ε, πληροφοριοδότες. Και το Υπουργείο Εξωτερικών έδωσε και το όνομά μου σε κάποιους, παρεπιπτόντως σας το λέω αυτό. Αλλά τα πράγματα δεν σταματούν μόνο στην τεχνολογία. Δεν ε, σημαίνει ότι υποκλέπουν μόνο τους υπολογιστές μου, τα τηλέφωνά μου, αλλά έχουν υπάρξει και άτομα της οικογένειάς μου και ε, ε τα οποία ε, αντιμετώπισαν προβλήματα. Η σύντροφός μου ξύπνησε στη νύχτα και είδε κάποιον να την στοχεύει με ένα όπλο. Ε, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν κάποιος ε, μου δημεύει την περιουσία και με συλλαμβάνει, πραγματικά με θεωρούν τρομοκράτη, δεν μου δίνει τη δυνατότητα να έχω δικηγόρο, ε, δεν μου δίνει τη δυνατότητα να πάω καν στην τουαλέτα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ε, σαν συνέπεια όλων αυτών εγώ πλέον ζω στη Γερμανία γιατί είναι καλύτερα να είμαι μετανάστη στο Βερολίνο παρά να είμαι πολίτης των Ηνωμένων Πολιτειών. Και αυτό νομίζω ότι σας λέει λίγα πράγματα για την κατάσταση. Και δείτε και τον Γκλέν, ο οποίος ζει πλέον στο Ρίο και... Ε, και η Πόιτερη, η οποία είναι γειτόνισά μου στο Βερολίνο. Ε, νομίζω ότι το τι ακριβώς έχουν κάνει ε, εξηγεί τα πράγματα. Κανένας από εμά δεν βιάζεται να πάει στις ΗΠΑ και να καταλήξει σαν την Τζέλσι Μάνινγκ ή σαν τον James Rising. Νομίζω ότι είναι τεράστιο πρόβλημα γιατί ο Ομπάμα δεν τηρεί τις δηλώσεις του για, τις προστασία, την προστασία των δημοσιογράφων και γι' αυτό και τους παρακολουθεί. Ε, γι' αυτό βάζει κοριούς και όταν ε, όλοι υπό όρκο ε, λένε ψέματα για τις παρακολουθήσεις, ε, ορισμένες φορές ε, βλέπουμε ότι είναι αδίστακτοι, τους αποτελούν στόχο ως πολιτικοί εχθροί και νομίζω ότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτό το οποίο μου δίνει ίσως ελπίδα είναι ότι στην Ευρώπη γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση για αυτά τα πράγματα και πραγματικά υπάρχει ελευθερία του τύπου, παρά το γεγονός ότι το πρώτο εδάφιο του Αμερικανικού Συντάγματο είναι πολύ καλό, υπάρχουν πολλές αμερικανικέ ε, εκδόσει οι οποίε δίνουν τα ε, άρθρα του ε, στη CIA πριν τα δημοσιεύσουν. Ε, και αυτό το οποίο έγινε με τα Wikileaks και τους New York Times ε, με ε, κάθε σεβασμό προς τους New York Times και στον Κέλλερ νομίζω ότι αυτό είναι προσβλητικό. Όταν εργάζεται κάποιος για το Spiegel δεν υπάρχει τέτοια συνεργασία. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι επαληθεύουν ότι όντως είναι πραγματικότητα τα στοιχεία και δημοσιογραφούν και αρθρογραφούν για αυτά τα οποία συμβαίνουν. Δεν θα μπορούσα εγώ να κάνω κάτι τέτοιο από τις ΗΠΑ και πάλι, τουλάχιστον όχι για πολύ καιρό και θα πρέπει επίσης να ε, σπάσει αυτός ο μύθος, να καταρρεύσει αυτός ο μύθος ότι όλα αυτά έχουν προκύψει σαν συνέπεια της 11 Σεπτεμβρίου. Δεν είναι. Υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο λέγεται Shamrock, το οποίο σας ενθαρρύνω να το εξετάσετε και ένα άλλο πρόγραμμα το οποίο ήταν πρόγραμμα του FBA, λέγεται Corental Pro Counter Intelligence Program και εκεί έχουν ε, ε, τα στοιχεία για τον ασμό του Μάρτιν Λούθερ Τζούνιορ και από πολλών άλλων ανθρώπων και αυτό το οποίο βίωσε η σύντροφός μου, τη κράτησή μου σε αεροδρόμια ή ε, το να μπαίνουν ε, στο σπίτι μου και να μην, αφήνουν, να μην παίρνουν τίποτα απλώ να μου ψάχνουν το σπίτι. Όλα αυτά πλέον γίνονται ηλεκτρονικώ και τώρα, σε αντίθεση με τη δεκαετία του 70, η Αμερικανική κυβέρνηση λέει ότι είναι απολύτω νόμιμο και ε, βάσει της, ε, του νόμου Πάτριο, το ορισμένε φορέ έχουν και δίκιο. Πολλά είναι για να απαντήσω άλλε ερωτήσει. Εν συντομία λοιπόν να σας πω όταν ο Ομπάμα λέει ότι δεν χρειάζεται να φοβόμαστε, καταρχά νομίζω ότι προσβάλλει καθέναν από εσά εδώ στην αίθουσα. Διότι λέει στου Αμερικανού μην ανησυχείτε, δεν ε, κατασκοπεύουμε Αμερικανού. Και τι γίνεται για όλου του υπόλοιπου πολίτε του πλανήτη. Για μένα αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό και ζητώ συγγνώμη εξ ονόματος αυτού του απίστευτα προσβλητικού Προέδρου μου που λέει κάτι τέτοιο για τον καθένα από εσά, διότι αυτό είναι απαράδεκτο στον πολιτισμένο κόσμο. Και επίσης κάνει και λάθος, διότι η εμπειρία που έχω για το Wikileaks είναι ότι οι Αμερικανοί πρέπει να φοβούνται ακόμα περισσότερο και ο λόγος είναι γιατί υπάρχει ένα σύστημα και μια νοοτροπία καταπίεσης που ορισμένες φορές είναι τόσο απλή που μπορεί κάποιος να μην κάνει τηλεφώνημα γιατί θα φοβόταν ότι θα διαρέσουν τα στοιχεία από το τηλέφωνό τους. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν γνωρίζουν, ε, δεν έχουν τηλέφωνο που να είναι γνωστό τους, ε, της πάση και απλώς το βάζουν στην πρίζα όταν πρέπει να κάνουν ένα επίγον τηλεφώνημα. Τώρα, τι γίνεται με ολοκληρωτικά καθεστώτα, χρησιμοποιείται προς αυτόν τον τρόπο, χρησιμοποιείται για ε, διάφορους σκοπούς, ναι, παραποιούνται στοιχεία. Εμένα με έχουν κρατήσει στα σύνορα και μου έχουν πει ότι θα είχα πολύ σοβαρά προβλήματα, αλλά τελικώς δεν μπορούσαν να με συλλάβουν, το οποίο είναι συναρπαστικό να το σκεφτεί κανεί. Δεν μου δόθηκε ο φάκελος, δεν μπορώ να το διορθώσω, δεν έλαβα γνώση, τον είδα κατά λάθο όταν με είχαν σε μια αίθουσα ανάκρισης και δεν ήταν τόσο καλός αυτός ο διπλός καθρέφτης. Και σε αυτή την περίπτωση είπα τα στοιχεία αυτά είναι λανθασμένα και μου είπαν όχι δεν μπορείτε να τα δείτε. Και είπα μα τα είδα. Και μου είπαν όχι δεν τα είδατε. Εντάξει δεν τα είδα. Κάποιοι κάνουν λάθη, τώρα αν γίνονται και αυτά τα λάθη είναι παπά Ευαγγέλια. Τώρα το πώς μπορούμε να το κάνουμε ε, χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας ως συσκευή ανείχνευσης. Κάνετε ένα τηλεφώνημα, δείτε αν σας παρακολουθεί κάποιος. Και μέσω της εξωτερικής ανάθεσης ε, τα ε, στοιχεία που περιλαμβάνει το τηλέφωνό σας, το κινητό σας τηλέφωνο, στέλνονται σε ένα κτίριο στο Ισραήλ ε, και ουσιαστικά το προϊόν δεν τους ενδιαφέρει καθόλου, δεν τους ενδιαφέρει τι γίνεται με τις χρεώσεις ή οτιδήποτε άλλο. Θα πρέπει λοιπόν να ζούμε σε έναν κόσμο που θα έπρεπε να είναι αδύνατες αυτές οι αναθέσεις εξωτερικούς. Τελικά. Αυτή η τρίτη εκδοχή των Wikileaks χτες βγήκε στη δημοσιότητα. Ήδη τώρα που μιλάμε ε, δημοσιοποιείται και αυτό δείχνει κάποιες ε, τεχνικές που έχουν στις αγορές των δισεκατομμυρίων αυτές οι υπηρεσίες και οι εταιρείε που προωθούν αυτά τα ποσά. Έχουμε και την υπηρεσία αντικατασκοπίας που ασχολείται την αγούκη λέξη που διαπίστωσε ότι πάρα πολλοί αυτούς που παρακολουθούσαν ταξίδευαν από την Ευρώπη σε αυταρχικά καθεστώτα για να, για να πουλήσουν και software για να παρακολουθήσουν κάποιους που τους ξέρω. Μισογραφούς στο Μαρόκο, στην Αιθιοπία ή ε, στην Αίγυπτο. Οπότε επ' αυτού πολλά θα μπορούσε να κάνει η Ευρώπη σταματώντας αυτού του είδους τις εξαγωγές ή τουλάχιστον να αναγνωριστεί το δικαίωμα προσφυγής στα δικαστήρια κάποιου που φύγεται. Γιατί έτσι προκύπτει ζημία εις βάρος αθώων με αυτού του είδους την παρακολούθηση. Τέλος, θα πρέπει να σας πω ότι έχουμε τον ιδιωτικό βίο και από τη μία και από την άλλη έχουμε την ε, ασφάλεια, την κρατική. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να ε, μελετήσουμε αυτό το επιχείρημα και να το αποδομήσουμε. Είναι λάθος, είναι έολο. Και αυτό διότι ο ιδιωτικός βίος πάει χέρι-χέρι με την κρατική ασφάλεια. Δεν είναι δυνατόν να θεωρήσουμε ότι υπάρχει ιδιωτικό βίο, να κανεί απεμπολίσει το δικαίωμα στο ιδιωτικό βίο. Δεν έχει, δεν έχει, δεν έχει νόημα αυτό. Ε, ξέρετε ότι η ΚΙΠ στην Αμερική ε, παρακολουθεί ακόμα και τις ερωτικές σχέσεις κάποιου στόχου της. Επομένως, θα πρέπει κάποιος κάτι να κάνει. Άρα το θέμα είναι αξιοπρέπεια η θέμα ελευθερίας και όλα αυτά από την άλλη μεριά έχουν να κάνουν με την ακαιριότητα, με, με, τη διαβάθμιση, το απόρριτο, με τη συνένεση. Όλα αυτά απουσιάζουν. Απλώς λειτουργούν αυτά τα συστήματα. Ή πολλές φορές, ε, τέλος πάντων, τα συστήματα είναι έτσι φτιαγμένα που να μας ε, παραβλάπτουν τα συμφέροντα. Τι να σας πω, έχουν φτάσει όλοι οι ρεπόρτες όσοι κάνουν έρευνες, δημοσιογράφοι, να φύγουν από την Αμερική και να έρθουν να μείνουν στην Ευρώπη. Και έχετε εδώ πέρα έρευνα, έχετε ανάπτυξη, ούτω ώστε να προκύψει, να αναγνωριστεί το ότι χρειάζεται η ασφάλεια, αλλά θα πρέπει να το δούμε αλλιώς, να είναι η εξαίρεση το να κατησχύει η ασφάλεια της Δυτικού Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε. κύριε Τζέκοβα Ήταν πάρα πολύ συναρπαστικά όσα είπατε. Μπράβο για το θάρρος σας. Οπωσδήποτε. Έτσι όπως μιλήσατε, ακούσαμε κάποιον που μιλάει ειλικρινά, με ευθύ τρόπο. Ήταν πολύ χρήσιμο το τι ήθελατε να μας μιλήσετε. Και ακούσαμε την πραγματική σας δημιουργία υπέρ αυτών των ε, αξιών που ασπάζεστε. Όπως σας είπα, έχουμε μείνει πίσω. Και θα πρέπει τώρα να δούμε το δεύτερο πάνελ που αφορά τις παρακολουθήσεις, τις υποκλοπές βάσει του Έσελον. Ο, ο, ο κύριος ε, Κάρλος Κοέλιο, ο συνάδελφος, ο δημοσιογράφος, ο κύριος Ντάνκαν Κάμπελ, Καλώς ορίσατε. Θα μιλήσετε εσείς δεύτερος, κύριε. Ο Κόλλη, ευχαριστώ πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος και δεν έχω πολύ χρόνο. Και θα ξανά έχω την ευκαιρία να σας τα πω, αλλά όχι ο κύριο Κάμπελ. Οπότε νομίζω θα ήταν πιο ενδιαφέρον να ακούσουμε τον κύριο Κάμπελ. Τέσσερα θέματα έχω να θίξω. Πρώτα πρώτα ήταν αρκετά εύκολο να προεδρεύσω στην Επιτροπή που ασχολήθηκε με το έσωρον. Διότι είχαμε ως θεμέλιο την έρευνα του κυρίου Κάμπελ. με τον Γκέρχαρντ Σμιτ που ήδη μας μίλησε, που ήταν ο εξαιρετικός μας εισηγητής. Κατά δεύτερο λόγο, ότι υπάρχει το έσωρον. Αυτό σημαίνει όταν κάποιος μίλησε σήμερα για το σύστημα, το πρόγραμμα των πέντε ε, ματιών. Αφορούσε τις υποκλοπέ το δίκτυο μεταξύ Ζηλανδία, Αυστρίας, Καναδά ή Αγγλία. και αυτοί λοιπόν παρακολουθούν και μοιράζονται τις πληροφορίες. <clears throat> Επίσης αποδείξαμε κατά τρίτον ότι μετά την πτώση του τείχους και το τέλος του ψυχρού πολέμου μεταξύ Σοβιετικής Ένωσης και είπα έγινε προσανατολισμό. Αντί να παρακολουθούν ιστορικού στόχου, παρακολούθησαν επιχειρηματικού ε, στόχου απλών φυσικών προσώπων. Είναι επομένω οικονομική, οικονομική και κατάσκοπη και αποδείξαμε ότι υπάρχει ένα τέτοιο σχέδιο. Μιλήσαμε με τον James Γουλσάιτ, ε, έναν πρώην διευθυντή τη CIA όταν πήγαμε στην Αμερική και στις 22 Μαρτίου του 2000 αναγράφηκε αυτό στην ε, Wall Street Journal. Υπήρξε ένα άρθρο που έλεγε «Γιατί η Αμερική να κατασκοπεύει τους συμμάχους της». Ο δε τίτλος του άρθρου δεν ήταν με ερωτηματικό. Ε, δεν ήταν ε, τι, γίνεται αυτοί αμφιβάλλουν για το τι κάνουμε εμείς. Όχι, ήταν το θεώρησε δεδομένα και, και, και έτσι ετίθεται το ερώτημα. Οπότε και αυτό είχε σχέση με τις ενδιαφέρουσες επαφές που έχουμε με τους Αμερικανούς. Να πάτε να διαβάσετε το άρθρο, δεν σας λέω τι άλλο έλεγε. το έχει, το έχει. Ε, το Κοινοβούλιο ή στα αρχές της Επιτροπής για τέσσερα. Τώρα, τι άλλαξε από το 2000 μέχρι σήμερα. Όπως θα σας πει και ο κύριος Κάμπερ, είμαι βέβαιος, το δίκτυο έσυλων μπορούσε να υποκλέπτει σήματα ασύρματου, σήματα από δορυφόρο, τηλέφωνα, μηνύματα, φαξ, αλλά τότε υπήρχε κάποιο προσεκτική περιγραφή σε σχέση με το α, που κανείς κάνει τις τι, τι, τι κατασκοπεύει. Δηλαδή ότι οι Αμερικανοί προσέχανε ε, να κατασκοπεύσουν τους Αμερικανούς και οι Βρετανοί όταν θέλανε να παρακολουθήσουν βρετανικές, βρετανικούς στόχους απευθυνόντουσαν στους Αμερικανούς. Ο κ. Κάμπελ είχε πάρα πολλά στοιχεία από αυτού του είδου τη συνεργασία. η Επιτροπή μα έκανε το ίδιο. Συλλέξαμε στοιχεία για αυτήν την συνεργασία. Σήμερα δεν έχω καμία ανάγκη να κάνω κάτι τέτοιο. Οι μυστικές υπηρεσίες κατασκοπεύουν την ιδέα τους στη χώρα. Και φυσικά τις πληροφορίες για τους δικούς τους συμπολίτες τις δίνουν και στις άλλες μυστικές υπηρεσίες. Είναι αυτό που προηγουμένως συζητήσαμε. Τίποτα, έχουν ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Το τελευταίο τώρα θέμα που θέλω να θίξω, αν κατακλείδη, είναι το εξή. Εάν καταφέρουμε να αποδείξουμε, το καταφέρουμε το 2000, γιατί, παρά το καταφέρουμε, δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι για να φρενάρουμε το πρόγραμμα εκείνο. Εγκρίθηκε η εκθεσία Σιόλων δύο μήνες πριν την επίθεση της 10 ε, Σεπτεμβρίου. Οπότε φυσικά κατόπιν υπήρχε μεγάλη συναισθηματική ε, φόρτιση και υπήρχε ελεγγύη προς τους Αμερικανούς ε, φίλους και κανείς τότε δεν έθεσε τάπητος αυτές τις αποκαλύψεις που κάναμε τίποτα για όλε αυτέ τι δραστηριότητε που είχαμε αποδείξει ότι υπάρχουν. Ότι δηλαδή και ε, ε, κατασκόπευαν φίλους, κατασκόπευαν συμμάχους και κανένας δεν τόλμησε αυτό να το ψάξει. Γι' αυτό σας λέω. Η επίθεση 11 Φεβρουαρίου όχι μόνο άλλαξε την οπτική αλλά και μετά διαμορφώθηκαν αυτές οι απειλές προς τις δημοκρατικές ελευθερίες. Αυτές τις οποίες εμείς έχουμε θεμέλει. Και επίση αυτό ήταν η ταφόπλακα για την έκθεση που συντάξαμε για το ΕΣΕΛΟΝ. Όλα αυτά μετά την, μετά την τρομοκρατική επίθεση. Όλα αυτά τότε είχαν συζητηθεί. Ναι, Είχαμε κάποιες διαφορές, διχογνωμίες, ε, υπήρχε διαφορά με τη σημερινή κατάσταση, το επίπεδο της τεχνολογίας, οπότε καταλαβαίνω και για δύο, ο τελευταίος ομιλητής μας είπε πριν από λίγη ώρα, ότι το Echelon ήταν αστείο σε σχέση με το τι ισχύει σήμερα με το πρίσμα. Η υποκλοπή, το είδος των ε, δεδομένων, σας είπε για τη τεχνολογία, σας είπε για τα μεταδεδομένα, επομένως αυτά ήθελα να θέσω. Οπότε τώρα αντί της κυρίας Νετφέλ θα δώσω εγώ το λόγο στον κύριο Κάμπελ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, όντως είναι τεράστια ηρωνία γιατί εξ όσων θυμάμαι ακριβώς 12 ε, χρόνια έχουν περάσει από την 5η Σεπτεμβρίου του 2001 που εγκρίθηκαν 24 συστάσεις στη έκθεση Γκέρχαρτ Σμιτ και ομόφωνα αν θυμάμαι καλά εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο ακριβώς 12 χρόνια πριν και είναι τραγικό και αυτό μας κληροδότησε ε, ίσως η 11η Σεπτεμβρίου, ε, ότι κατάφεραν οι τρομοκράτες να πλήξουν τόσο πολύ με τη δράση τους τα ατομικά μας δικαιώματα και τις ελευθερίες. Και τα χρόνια ήδη πριν από την 11η Σεπτεμβρίου. Και πριν μιλήσει ο Σνόντεν, είχαμε ε, αυτή την κατάσταση και με την επόμενη δεκαετία συνήθισαν συμφωνίες ε, μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ηνωμένου Βασιλείου και των τριών άλλων αγγλόφωνων ε, εταίρων τους. Και ευρύτερε συμφωνίες ε, αποκαλύπτονται σήμερα. Ακόμα και για το έτος που αναφέραμε, το Ηνωμένο Βασίλειο στη βορειοδυτική Αγγλία είχε εγκαταστάσεις για υποκλοπές όλων των επικοινωνιών. Όχι μόνο τα μέτα στοιχεία με τα δεδομένα, αλλά και αναγνώριση φωνής και μια σειρά άλλα. Ολόκληρο πύργο χτίσανε και στο δείχνω για να ε, υποκλέπτουν τα ραδιοκύματα και τις διεθνείς ε, επικοινωνίες. Βλέπετε στη διαφάνεια τον πύργο. Αυτό το σύστημα έσελων ήταν εύκολο να εντοπιστεί και να ε, το δει κανεί γιατί ήταν ορατό. Είχαν ολόκληρες ε, τέτοιε εγκαταστάσεις και δορυφορικές, με δορυφορικέ κερές. Ενώ σήμερα το κέντρο συλλογή συλλογής όλων των στοιχείων διαδικτύου 1 είναι λιγότερο ορατό αυτές οι δορυφορικές κεραίες στην αρχή ήταν πάρα πολύ ε, ορατές και ήταν τμήμα και των δορυφόρων. Αλλά τώρα βλέπετε τα νέα κτίρια που έχουν προσθεθεί για το σχέδιο Tempora που ε, αποκάλυψε ο Σνόντεν και τόσα πολλά ακούσαμε σχετικά. Επίσης, οι αποκαλύψεις μας είπαν και τι πρόκειται να έρθει από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όταν ένα Αμερικανός έδωσε σχέδια και έγγραφα και εικόνες για το πόσο οπτικές ίνες μπαίνουν ε, στη δυτική όχθη των ΗΠΑ στις επικοινωνίες ε, των διαδικτύων. Και τότε αρχίσαμε πολλοί από εμά να ψάχνουμε μυστικές αίθουσες τέτοιες ε, παντού. Αλλά μόνο και 2008 ένας δημοσιογράφος στη Βρετανία έμαθε αυτό το πρόγραμμα ελέγχου του διαδικτύου ε, πάρα πολύ ισχυρό το οποίο κατέληξε στο πρόγραμμα Tempora με ε, πολλές άλλες, πολλούς άλλους σταθμούς και κλιμάκια. Το σύστημα Echelon λοιπόν όχι απλώς λειτουργεί απλώς αλλά έχει ε, πολλαπλασιαστεί και έχει αλλάξει όνομα. Το λένε Fornsat τώρα. Αυτό είναι μία από τις διαφάνειες του Snowden που δημοσιεύτηκε το πριν ένα μήνα στη Βραζιλία και δείχνει όλους τους υποσταθμούς έσελων αλλά τον κόσμο. Ε, το πιο κοντινό μας τώρα εδώ είναι στη Γερμανία, αλλά βλέπετε ότι υπάρχουν νέοι σταθμοί στην Ινδία, στην ε, Ταϊβάν, στην Κένια, τη Βραζιλία. Απανταχού της γης, όχι μόνο στις Ηνωμένε ε, Πολιτείες, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Ομάν, σε διάφορους συμμάχους. Εκεί στο Ομάν καλύπτει τη Μέση Ανατολή ο σταθμός αυτός. Έχει αυξηθεί το σύστημα αυτό, είναι ένα κλάσμα και μόνο και τώρα καταλαβαίνουμε πόσο μικρό ήταν το έσελον σε σχέση με την αράχνη που προέκυψε από τις τεχνικές εξελίξεις. Και το είπε και τη μοιραία χρονιά 2001 το Κοινοβούλιο. Αμάν Κοριός μπήκε στο σύστημα μια στιγμή. Να, αυτό είναι από τα στοιχεία του Snowden, αλλά και στην Ιαπωνία βλέπετε το σταθμό Έσελον. Εδώ ε, τις δυνατότητες το είχαμε πει από το 2000 από το Έσελον, από την έκθεση που είχα κάνει για την Επιτροπή με εισηγητή τον κύριο Σμιτ ε, που το συμπεριέλαβε μετά από επαλήθευση και στα συμπεράσματα. Και άλλοι σταθμοί εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό που ίσως έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για να καταλάβουμε είναι πώς γίνεται η συλλογή των διαφόρων input, τα στοιχεία πώς τα συνδυάζουν ε, για την ανάλυση του συστήματος του διαδικτύου που έχει καλύψει όλο τον πλανήτη. Το σύστημα αυτό το είπε προηγουμένως ο Jacob Applebaum και οι άλλοι. Ex-key score και cross-key score. Αυτά τα ξέρουν αυτοί ε, που εργάζονται με ε, τους υπολογιστές. Ε, δι' δεύτερη καριέρα μου, μετά το εσελόν μπήκα σε αυτή την κατηγορία forensic computers. Πώς μπαίνουν τα στοιχεία στο σύστημα. Με τρεις τρόπους. Βλέπετε εδώ κάτω στη διαφάνεια με σκοτεινούς κώδικες. Ένας λέγεται Fonsat που είπαμε ότι είναι το νέο όνομα του Echelon και των δορυφόρων για τις εμπορικές ε, τηλεπικοινωνίες. Και το τρίτο δεξιά, SSO, είναι ε, επιχειρήσεις ειδικών πηγών. Και αυτό τι σημαίνει. Είναι οπτικές, είναι εμπορικά καλώδια και καμιά φορά ίντερνετ και τηλέφωνο με μυστικές συμφωνίες που έχουν κάνει με εταιρείε τηλεπικοινωνιών. Και ο τρίτος τρόπος εισόδου των στοιχείων και είναι ενδιαφέρον αυτό το F6 που είναι ε, ένα τμήμα μιας εθνικής υπηρεσίας πληροφοριών και μιας υπηρεσίας που συλλέγει στοιχεία και κάνει υποκλοπές ανά τον κόσμο σε 75 ή 80 τόπους, ε, σε πρεσβείες της Βρετανίας ή σε ε, άλλα τέτοια κτίρια. Στόχος είναι τα υποθαλάσσια καλώδια, τα καλώδια και οπτικών ινών που συνδέουν τα πάντα τώρα και τα εμπορικά και το, το ε, ήταν στους δορυφόρους, αλλά τώρα έχουμε περάσει οπτικές ίνες και στα καλώδια. Και όπως μάθαμε από το Snowden, το Ηνωμένο Βασίλειο πρωταγωνιστεί εδώ, σκουπίζει όλο το ελεύθερο δωρεάν ίντερνετ. Και ποια είναι η είδηση εδώ. Μέχρι το 2010 περίπου, μόνο 18 υποθαλάσσια καλώδια προς το Ηνωμένο Βασίλειο παρακολουθούντο και έμπαινε στο σύστημα τα στοιχεία. Ορισμένες εμπορικές εταιρείες δεν είχαν ακόμα εμπλακεί τόσο πολύ, αλλά στη συνέχεια υιοθετήθηκε ένα σύστημα από τους θερματικούς σταθμούς των Καλωδίνων. Βλέπετε που βρίσκεται το Μπιούτ στην νοτιοδυτική ε, Αγγλία. Είτε με τη συνένεση των εταιριών ε, παρακολουθούνται τα καλώδια και οι οπτικές ίνες και συλλέγονται τα στοιχεία ή ακόμα και χωρίς καν τη γνώση χωρίς τη συνένεση με μυστικές υποκλοπές ε, σε εταιρείε που ξέρουν ότι δεν θα συμφωνήσουν. Και ε, μπαίνουν κρυφά λοιπόν στα συστήματα αυτά. Και ποια είναι η έκπληξη εδώ. Έχουμε μια νέα οργάνωση που μπήκε στα πέντε μάτια, στα πέντε Five Eyes και τώρα φαίνεται ότι είναι ο μεγαλύτερος συνεργάτης του GCHQ εκτός της αγγλόφωνης ε, σφαίρας και αυτή είναι η Σουηδία εδώ και χρόνια και έχουν περάσει τώρα και νέα νομοθεσία για το διαδίκτυο για να υπάρχει πρόσβαση στα, υπόγεια, στα υποθαλάσσια μάλλον καλώδια. Λέρκελ λέγεται η τοποθεσία κοντά στο Γιώτεμπορκ και ζητώ συγγνώμη για την προφορά μου, που είναι αυτός ο υποσταθμός ε, παρακολουθήσεων. Έχει σημασία αυτό για την οργάνωση Five Eyes ε, και για τη Σουηδία. Ε, ποιο είναι η σημασία, γιατί έχουν πρόσβαση σε καλώδια που δεν έχει κανένας άλλος. Συμμετέχει λοιπόν και μια χώρα ε, εκτός της δικής μου του Ηνωμένου Βασιλείου αλλά και μια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Σουηδίας και διαφέρει ο τρόπος συνεργασίας είναι πολύ ε, και ευρύς και αυτό μπορεί να σας ενδιαφέρει ε, χρησιμοποιούνται μυστικά ονόματα κώδικοι για ε, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένε Πολιτείε για να κρύβονται αυτά και όταν ε, παγιδεύουν ένα καλώδιο, ένα τηλέφωνο, δίνεται ένας κωδικός σε ένα μυστικό όνομα. Και βλέπετε εδώ τις διάφορες βάσεις. παρακολουθείτε το διαδίκτυο παγκοσμίω, το είπαν και προηγούμενοι ομιλητέ, κάθονται οι αναλυτές ε, στην κονσόλα τους και ε, έχουν αλλάξει και λεξιλόγιο. Τώρα συνδέουν ε, όλους τους συλλέκτες. Παλιά το λέγανε αυτό επί λεξικό. Τώρα έχουν αλλάξει ορολογία. Και εδώ έχουμε ένα κέντρο συλλογής στοιχείων ε, στην Ερυθρά Θάλασσα και πάλι ένας υποσταθμός έσελων που ε, έχει αυξηθεί η ε, λειτουργία του και η χωρητικότητά του. Υπάρχουμε και αστικού τύπου κέντρα συλλογής F6 από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών ο συνήθως με τέτοιους πύργους όπως αυτόν που ανακαλύφθηκε ε, το 99 στη βορειοδυτική Αγγλία. Τέτοιους πύργους έχουν οι πρεσβείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Εδώ είναι στη Γενέβη. Ήταν πάντα προφανές. Αν, αν περάσετε κοντά και δείτε προσεκτικά θα καταλάβετε. γιατί στην ταράτσα του κτηρίου υπάρχει αυτή η κατασκευή. Άκουσα, δεν ξέρω αν ισχύει, ότι δούλευε ακριβώς εκεί ο Έντουαρτ Σνόουντεν σε αυτή τη συγκεκριμένη εγκατάσταση πριν από λίγα χρόνια. Αντίστοιχα βλέπουμε και στη Λευκοσία στην Αμερικανική πρεσβεία και επίσης και στη Ρωσική πρεσβεία στην Λευκοσία. Παντού ε, όλοι τα ίδια κάνουν. Η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στις Βρυξέλλες που φαίνεται αρκετά ε, αυλαβής ε, και σχεδόν μπορούμε να τη δούμε με γυμνό μάτι από εδώ που καθόμαστε, αλλά αν τη δείτε από τον αέρα βλέπετε τι έχουν ε, προσθέσει ως εγκαταστάσεις στην ταράτσα του κτηρίου. Υπάρχει λοιπόν τεράστια δυνατότητα για τη συλλογή των συστημάτων ε, αυτών και των πληροφοριών. Εκεί που νομίζαμε λοιπόν ότι υπάρχει ένα μεγάλο σύστημα από το 1999 στο 2001, Τώρα έχουμε πέντε συστήματα που επικαλύπτονται και μπορούν ταυτόχρονα να συλλέγουν στοιχεία ε, σε υποκλοπές από, από δορυφόρους, από καλώδια, ε, από ανταλλαγές. Χρησιμοποιούν ε, τεχνική πρόσβαση, τακτική πρόσβαση. Hackers χακάρουν τα δίκτυα και τα κομπιούτερ αυτό ονομάζεται και εκμετάλλευση του δικτύου των υπολογιστών. CNE. Εν περιπτώσει υπάρχουν πολλοί τρόποι να πάρει κανείς στοιχεία από εμά, τους πολίτες, από τις εταιρείες, από κυβερνήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο ε, και στους provider ε, των Ηνωμένων Πολιτειών που δίνουν ε, πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ε, αν έχετε χρόνο ή ενδιαφέρον να κοιτάξετε τα διαγράμματα που δημοσιεύτηκαν στην Washington Post, ας πούμε, ε, ως αποκαλύψεις ε, του Snowden, βλέπετε ότι δεν είναι μόνο η NSA, αλλά και το FBI το ίδιο συλλέγει στοιχεία και η CIA και άλλες υπηρεσίες. Είμαστε όλοι πελάτες. Δεν ε, τα έχω, έχει αποκαλύψει όλα ο Σνόντεν ή αν τα έχει δεν τα λέει. Δεν λέει τι γίνεται με τους δορυφόρους σε ό,τι αφορά τις ε, ατομικές μας ε, προσωπικές ή εμπορικές επικοινωνίες. Οι γεωστατικοί δορυφόροι, ας πούμε, τι κάνουν και τι, τι συγκεντρώνουν. Ό,τι δεν μπορεί να συγκεντρωθεί με άλλο τρόπο. Η Αμερικανική κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι έχουν χάσει όλα τους τα μυστικά, έχουν αποκαλυφθεί. Δεν ισχύει αυτό, είναι πολύ κατακαιρματισμένα τα συστήματα. Τι έγινε μέσα σε 12 χρόνια λοιπόν που πέρασαν έκτοτε. Με τη μαζική ε, συλλογή και αποθήκευση στοιχείων αυξάνεται μαζικά και ο κίνδυνος. Και υπάρχει και τεράστιος αντίκτυπος στην κοινωνία των πολιτών. Αυτό ο κόσμος δεν τα καταλαβαίνει. Ε, εκτός ε, της, ε, του κόσμου των μυστικών υπηρεσιών. Η ανάλυση του δικτύου με χρησιμοποίηση των μεταδεδομένων, των μεταστοιχείων, δηλαδή ποιος τηλεφωνεί σε ποιον και τα λοιπά, έχει γίνει ένας χάρτης ολόκληρος και παρακολουθεί και φακελώνει ολόκληρη την ανθρωπότητα. Πραγματικά είναι απίστευτη ε, το θράσος και ανέδεια που έχουν αυτές οι υπηρεσίες και συλλέγουν όλα τα στοιχεία για όλους και τα αποθηκεύουν. Για πάντα ουσιαστικά. Το χακάρισμα των ε, ηλεκτρονικών υπολογιστών οργιάζει. Ε, το ξέραμε ότι υπήρχε, αλλά σε τέτοια κλίμακα είναι πρωτοφανή αυτά που συμβαίνουν. Ποια προβλήματα έχουμε τώρα απέναντί μας σε επίπεδο θεμελιωδών ε, ελευθεριών και δικαιωμάτων. Το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών και το Χάρτη των Δικαιωμάτων και ιδιαίτερα το τέταρτο εδάφιο θεωρεί και ερμηνεύεται με τρόπο ώστε να πιστεύουν ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα αφορούν μόνο τους πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών. Οπότε όταν πρόκειται για Ευρωπαίους πολίτες ή άλλους δεν υπάρχει πρόβλημα, κανένα όριο, κανένας περιορισμός, είμαστε εντάξει. Ωραία, πολύ ωραία. Θαυμάσιο, αλλά από ό,τι φαίνεται απέτυχε ή δεν ισχύει ε, για τους Αμερικανούς πολίτες ή εκείνους ε, που ε, έχουν την σύνεση να επικοινωνούν μόνο εντός των ΗΠΑ. Οι ΜΚΟ άργησαν να κατανοήσουν τη σημασία των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι οικουμενικά. Έχουμε και διακήρυξη, έχουμε και χάρτη και στις Ηνωμένε Πολιτείε και υπεγράφει και ειδικό πρωτόκολλο ε, σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Είχατε προσκαλέσει και Αμερικανούς, αλλά δεν ήρθαν να το δουν. Στη Γαλλία και στο Ηνωμένο Βασίλειο γίνονται κάποιες απόπειρες και στις Ηνωμένε Πολιτείες για την ενημέρωση, για τα συστήματα αυτά, ε, τα δόλια και ε, τα συστήματα παρακολούθησης. Παρά τις ε, αποτυχίες του, το σύστημα εφαρμογής του νόμου είναι ένα σύστημα το οποίο έχει ανοιχτούς ελέγχους και, και γίνεται ως κατάλληλος έλεγχος και οποιαδήποτε παρακολούθηση γίνεται από ε, συστήματα τα οποία κάνουν υποκλοπή θα πρέπει να είναι βασική απειλή την οποία θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε. Και μια ουσιαστική πτυχή κατά την άποψή μου είναι αν ανατρέξετε στο παρελθόν. Το ΕΣΕΛΟΝ ξεκίνησε το 1968. Αποκαλύφθηκε το 1988 από τον υποφαινόμενο και μετά έμεινε στη, κρυμμένο μέχρι που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενδιαφέρθηκε γι' αυτό 12 ε, χρόνια μετά. Αλλά τότε οι ηλεκτρονικοί υπολογιστέ ήταν πρωτόγονοι, είχαν ένα σύστημα το οποίο λεγόταν ε, dictionary, το λεξικό, το οποίο ήταν ε, πρωτοπόρο πριν από 10 χρόνια, αλλά αυτή τη στιγμή ε, είναι το ίδιο με το να ψάχνει κάποιο ένα εγχειρίδιο ή να κάνει μια αναζήτηση στο Google, κάτι που κάνουμε όλοι μας συνέχεια. Αλλά το πιο εκπληκτικό είναι ότι η αιτιολογία για την αυτόματη συλλογή όλων των στοιχείων, χωρίς να υπάρχει κάποια πρώτερη υποψία ή κάποιος ε, συγκεκριμένος λόγος, αιτιολογείται από τα όσα κάνουν αυτοματοποιημένες ρομποτικές διαδικασίες. Φαίνεται ότι οι νέες έννοιες έχουν ε, εισέλθει λόγω της προόδου της τεχνολογίας και θεωρείται ότι είναι ασφαλής να ανατίθεται η εποπτεία και η συλλογή πληροφοριών της ιδιωτικής μας ζωής σε ρομπότ τα οποία χρησιμοποιούν άνθρωποι που εργάζονται χωρίς κανέναν έλεγχο ε, για την καθημερινή τηλεπικοινωνία σε ε, κάτι το οποίο είναι πολύ εύκολο να γίνει. Είναι κάτι το οποίο είναι καινούριο στην ιστορία. Πρόκειται για ένα δεοντολογικό πρόβλημα το οποίο θα αντιμετωπίσουμε πολλοί από εμά του επόμενου μήνε ε, και εδώ και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μια τελευταία μου παρατήρηση για τα checks and balances, για το γεγονό ότι θα πρέπει να υπάρχουν έλεγχοι και να υπάρχει λογοδοσία, είναι ότι θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τους ε, κοριούς τους οπτικών ινών και υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις στις οποίες όντως βοήθησε την τρομοκρατία ε, και ε, ταυτόχρονα έχει και υπονομεύσει τις πολιτικές μας ελευθερίες. Αυτό το οποίο όμως αποδείχθηκε τους τελευταίους τρεις μήνες είναι ότι η έλεγχη και η λογοδοχησία, το γεγονός ότι θα, πρέπει να γνωρίζει το κοινό τι συμβαίνει, είναι το πιο σημαντικό το οποίο μπορεί να γίνει για τη δημοκρατική μας κοινωνία. Και το καλύτερο το οποίο θα μπορούσε να κάνει η Ευρώπη, και αυτό προτείνω, είναι να δοθεί καταφύγιο στον Έντουαρτ Σνόντεν γιατί είναι ο πληροφοριοδότης ο οποίος μας προσέφερε τόσους πολλές γνώσεις και ε, μας βοήθησε να κατανοήσουμε τι συμβαίνει. Σας ευχαριστώ. Thank you, Mr. Campbell, for ε, Ευχαριστούμε κύριε Κάμπελ. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα όσο και αν είναι θλιβερά αυτά τα οποία μας ε, παρουσιάσατε. Ε, ναι, είδατε. Ό,τι κάνουμε, ό,τι κάνουμε, ό,τι κάνουμε παρακολουθείτε, να ήταν και εκείνοι που με τη χύτρα εκείνη είδατε τι καταφέρανε οι δύο φοιτητέ. Εμά μένει ένα δεκαλεπτάκι συναδελφοί, γιατί μείναμε πίσω σχέση με το χρονοδιάγραμμα κατά μία ώρα. Οπότε και εγώ σα προτείνω. Να δώσουμε το λόγο. Στον Κλοντ Μωράη που είναι ο εισηγητή και ισω εχουμε έχουμε δύο-τρία λεπτά για κάποιες παρεμβάσεις πάρα πολύ σύντομε από τους σκιώδεις εισηγητάς, εάν πραγματικά το θέλουν. Συμφωνείτε? Κλώδη, συμφωνείς? Ναι. Ωραία, άξιλ φως. Δύο παρέμβαση. Ε. <laughs> Μόνο αν έχεις ανάγκη έτσι απόλυτη, αν δεν κρατιέσαι. Κράλος, μίλησες για την έκθεση Έσελον Και είπες γιατί δεν είχε συνέχεια και συνέπειες. Αν θυμάμαι καλά, στην έκθεση Έσελον. υπήρξαν πολύ μεγάλες νομικές δυσκολίες να γίνει κάτι σε ευρωπαϊκό καν επίπεδο. Δεν έχω την αίσθηση ότι έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα έκτοτε αλλά θα ήθελα πάρα πολύ σύντομα να μας πεις τη γνώμη σου γι' αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και για τη συντομία. Ο Γιάν Άλπρεχτς. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σλούβικ, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίασή σας και ελπίζω ότι όλες αυτές οι πληροφορίες πρόκειται να ληφθούν υπόψη και από τον κόσμο, διότι έχω την εντύπωση ότι ε, θα, δεν πρέπει να μείνουν ε, εδώ στους τοίχους Και έχουμε μόνο σε αυτό το σύστημα παρακολούθησης που είπατε κύριε Κάμπελ και μήπως θα μπορούσατε να μας πείτε ποια ήταν τα κράτη που ενεπλάκησαν πώς χρησιμοποιήθηκε το τέμπορα, το πρίσμ, το έσελον. Δεν κατάλαβα πολύ καλά πώς συναρμόζονται όλα αυτά, πώς συντεριάζουν. Έρνστ, ένα λεπτό. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τους τρεις. Ε, δεν είναι πάρα πολύ ε, επικοδομητικό να ακούμε την ώρα που σχολάμε περίπου <laughs> τι έγινε ε, σε σύγκριση με σήμερα από την εποχή του Έσελον. Μια ερώτηση έχω και μόνη. Τι θέλετε να συγκρατήσουμε τώρα εμείς, να κρατήσουμε ως βουλευτές από αυτά που ακούμε για να αντιμετωπίσουμε αυτό το μεγάλο θέμα. Τι να κάνουμε, τι, τι συμβουλές έχετε να μας ε, δώσετε για τις έρευνες που καλούμε θα να ε, κάνουμε και ποια είναι η συγκεκριμένη σας εμπειρία από την τότε Επιτροπή Έσελον. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κάμπελ παρακαλώ πάρα πολύ σύντομα να απαντήσει στις ερωτήσεις και μετά ο Κλοντ Μωράες για να κλείσει. Um, Κάμπελ. Ναι, το έξικισκο ήταν παραφιάδα του, του Φόνσελ. Ε, οι δορυφόροι υπέκλειπταν από το Ιντερνετ και το σύστημα αυτό είναι το αμερικανικό αλλά έχουν το δικό τους οι Άγγλοι. Ναι σε σχέση με το πρόγραμμα Τέμπορα. Από ό,τι φαίνεται λειτουργεί με παραμείο τρόπο. Άλλωστε τα υλικά τα αγοράσαν από τους Αμερικανούς. Επομένως, το συμπέρασμα είναι ότι υπήρχε μία βάση δεδομένων, η Αμερικανική ΚΙΠ χρησιμοποιούσε τη Βρετανική βάση δεδομένων, η οποία είχε πρόσβαση εις ε, τα μεταγενικά στοιχεία και έχουμε ε, κάποια όχι τόσο σαφή απεικόνηση του που ε, έτρεχε το σύστημα και η δική μου ερμηνεία είναι ότι επρόκειτο για το σύστημα αυτό το οποίο έτρεχε στις Αμερικανικές Πρεσβείες σε διάφορες χώρες εκεί όπου μπορούσαν να έχουν τις αναλυτικές δυνατότητες να χρησιμοποιούν αυτό το το σύστημα. Γιατί αυτό εκτός, έξω από αυτές τις πέντε βασικές χώρες που είπαμε δεν έχουμε καταγράψει πού αλλού έτρεξε. Απλώς ξέρουμε τις αποκαλύψεις από πλευρά Snowden. Και οι βασικές χώρες που ίσως είχαν πρόσβαση στο εξκίσκο είναι η Ινδία, το Ισραήλ, ε, η Σουηδία και η Γαλλία. Αυτά τώρα είναι συμπεράσματα ε, από τις αποκαλύψεις σε πολλά έγγραφα. Οπότε θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι αυτά ε, χρησιμοποιήθηκαν από τα πέντε μάτια, τους πέντε, τους συμμάχους. Και εν μέρει χρησιμοποιούσαν το σύστημα για κάποια εξωτερική. Οπότε, Τώρα γίνονται αποκαλύψεις, κάποια θέματα αποχαρακτηρίζονται. και οι μέσα από την ΚΙΠ απεκάλυψαν όλα αυτά. Οπότε απεκαλύφθηκε, τέλο πάντων προκύψε συμπέρασμα ότι ίσω και 30 χώρε μπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε αυτή τη βάση δεδομένων. Τώρα έχουμε άλλε ερωτήσει όσον αφορά τι πολιτικέ πτυχέ, τι νομικέ πτυχέ από τον κύριο Καρλό Κουάλια. Είναι αλήθεια ότι κάποια από αυτά τα ζητήματα ε, είναι εκτός κοινοτικού δικαίου. Αλλά όμως ως κοινοβούλιο εμείς θα να προβαίνουμε σε συστάσεις για να κατονομάζουμε τους ε, υπετίους ε, γιατί όπως και στο παρελθόν πρέπει να ξανακάνουμε το ίδιο. Να προβούμε σε συστάσεις προς τη ΣΥΠΑ για να προχωρήσουν σε κάποιες διεθνείς συμβάσεις που στις οποίες προχωρήσει μέχρι τώρα. Και να απευθυνθούμε και στον ΓΑΜΑ του ΟΗΕ, στο Συμβούλιο της ε, Ευρώπης. Μπορούμε να τα κάνουμε αυτά. Να προβούμε σε κινήσεις, να προστατεύσουμε τη μυστικότητα, το απόρριτο των συνομιλιών μας, την επικοινωνία μεταξύ Επιτροπής και Κοινοβουλίου, μεταξύ μόνο και των αντιπροσωπιών μας όλο τον κόσμο. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν μορφή των συστάσεων. Μπορεί να μην υπάρχει ε, αρμοδιότης με την νομική έννοια, αλλά έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε τις συστάσεις. Και το είπα στον Κλοντ Μωρές να ρίξει μια ματιά στις τότε 54 ε, συστάσεις μας. Μερικές από αυτές δεν στέκουν σήμερα, αλλά οι περισσότερες από εκείνες μπορούσαν κάλλιστα να επαναδιατυπωθούν και γιατί είναι απίστευτο το πόσο από εκείνες τις συστάσεις ακόμη ισχύουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εξετάσαμε τρία βασικά ζητήματα σήμερα. Εδώ ολοκληρώσαμε τη δουλειά μας. Ελευθερία του τύπου, παρακολούθηση από πλευράς ε, υπηρεσιών πληροφοριών και τρίτον τα σημεία που πρέπει να αντιλήσουμε από την ερευνητική του Πραγματική Επιτροπή για το Echelon. Και τώρα, ο συγκεκριτής μας, ο κ. Κλόντ μπορεί να προβεί στις καταληκτικέ παρατηρήσεις. Ναι, Σοφή, ξέρω ότι έχουμε αργήσει, δεν θέλω να ταλαιπωρήσω τους ακροατές, να ξαναλύσω την υπομονή του. αλλά... Πάρα πολλοί μας ακούνε από το ίντερνετ, Πρόκειται για μια ακρόαση. Δεν ήθελα να υποβάλω και εγώ ερωτήσεις στο πάνελ με το έσυλον, οπότε πρώτα από όλα κάποια διαδικαστικά. Πρόκειται για την πρώτη έρευνα. Είχαμε όλους αυτούς που σήμερα, είχαμε όλους αυτούς που ακούν, ε, μιλούμε για μια ερευνητική επιτροπή που θα κρατήσει τέσσερα, ε, τέσσερις μήνες. Ε, ρίξτε μια μεθιά στι παλαιότερε ερευνητικές επιτροπέ. Είχαν πάρα πολύ δύσκολο έργο σε σχέση με αυτά που ακούσαμε σήμερα. Σήμερα είχαμε το πιο, το πιο έντονο έργο. Έχουμε τέσσερις ε, μήνες ακόμα. Έχουμε για τον, πάμε μέχρι τον Ιανουάριο 2014 και ψηφοφορία το Δεκέμβριο. Οπότε από την μια μεριά έχουμε ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα για όλους μας και όλες κλπ. Θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, θα πρέπει να είμαστε και φιλόδοξοι, γιατί εδώ πέρα αυτό εμφανίζεται ως παράδοξο, αλλά νομίζω ότι με την πρώτη συνδρίαση καταλάβαμε ότι μπορούμε να εισφέρουμε με ποιότητα και επομένως ε, αυτό θέλω να σας πω με αυτές τις ε, καταληκτικές παρατηρήσεις ότι θα το χειριστούμε αυτό το θέμα φιλόδοξα. Κατόπιν των σημερινών και το θέμα της ελευθερίας των ΜΜΕ και το θέμα της, της, της, της, ε, της, των συμπερασμάτων από την υπόθεση έσελον. Όλα αυτά θα είναι έμπνευση για μας. Ε, ακούσαμε την και ο Καροσκόλιο για την επίδραση σε όλα αυτά ε, της 10 Σεπτεμβρίου. Άρα πρέπει να είμαστε αμερόληπτοι κλπ. Δεν θέλω επομένω σήμερα να σπεύσω να εξαγάγω συμπεράσματα θα τα κάνουμε όλα αυτά, θα δούμε και τις συστάσεις για το SLM. Αλλά αυτό που θα σας πω είναι το εξή. Τώρα αισθάνομαι ακόμα πιο φιλόδοξος και αισιόδοξο και ορεξάτο για αυτούς τους τέσσερις μήνες όπως τα είπε και η Σοφία. Έχουμε όμως αυτούς τους τέσσερις μήνες μπροστά μας. Πέραν της εμπειρογνωμοσύνης νομίζω ότι μπορούμε πολλά να πετύχουμε. Εάν είμαστε ε, συνεπείς όπως ήμασταν σήμερα για να διατυπώνουμε ε, ερωτήσεις, να ψάχνουμε τα πράγματα. Γιατί οι συστάσεις του έσουν δεν εισακούστηκαν λόγω εξωτερικών παραγόντων. Αυτό ήταν το ζουμί, όπως ακούσαμε τώρα τα τελευταία λεπτά. Αυτά θέλω να ολοκληρώσω, Πρόεδρε. Θα έχουμε 12 με 15 συναντήσεις. Την Πέμπτη στο Στασβούργο επόμενη συνάντηση. Θα ενημερωθεί όλος ο κόσμος, θα έχουμε επίσης και μετάδοση της συνάντησης από το ίντερνετ. Θέλουμε πλήρη διαφάνεια στις συναντήσεις μας. Ναι. Συστάσεις πρακτικά όλα, όλα. Όλα θα είναι ανοιχτά, όλα θα είναι ε, γεμάτα διαφάνεια, ακριβώ όπω θα περίμενε κανεί από μια τέτοια ερευνητική των πραγμάτων επιτροπή. Ε, ευχαριστούμε όλου όσου βοήθησαν για σήμερα. Thank Ευχαριστούμε πέρα τη συνεδριάσεω. Και όπω θα είπε ο Κλοντ Μωρέ, η επόμενη συνάντηση θα είναι την Πέμπτη στο Στρασβούργο. Στι 10 η ώρα. Mm. Ευχαριστούμε που ήρθατε.